Καλημέρα, αγαπητοί συνάδελφοι. Ξεκινάμε. Με την ε, δήλωση της Κομισιόν για το πρόγραμμα εργασίας της για το 2020 και δίνω τον λόγο στον Αντιπρόεδρο, κύριε Σεύκοβιτς. Παρακαλώ. Uh, uh, Ευχαριστώ κύρια Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Ευρωβουλευτές. Είναι τιμή μου που βρίσκομαι εδώ σήμερα για να συζητήσουμε το πρώτο πρόγραμμα εργασίας Κομισιόν υπό την Προεδρία της κυρίας Φοντερ Λάιν που εγκρίναμε χτες. Το πρόγραμμα αυτό είναι σημαντικό για δύο λόγους. Πρώτον γιατί δεν θα αποτελέσει απλά τη βάση εργασίας μας για το πρώτο έτος της ε, θητείας μας, αλλά γιατί παρουσιάζει την κατεύθυνση των πέντε ετών και ακόμα παραπέρα. Ας δούμε παραδείγματος χάρη την ε, μεγαλύτερη πρόκληση της εποχής μας, ε, την οικολογική και ψηφιακή μετάβαση που θα μας επηρεάσει όλους μας. Δεύτερον, επειδή ε, ξεκινάει μια ειδική σχέση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θα ξεκινήσω από αυτό που είναι σημαντικό και θεσμικά και πολιτικά και μου είναι ιδιαίτερο αγαπητό. Η έγκριση του προγράμματος του 2020 ήταν κάτι το οποίο κάναμε από κοινού. Είχαμε τη συνεισφορά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε κάθε φάση που ελήφθη υπόψη. Ήδη παίξατε κέριο ρόλο στην κατάρτιση των πολιτικών κατευθυντήριων γραμμών οι οποίες τώρα μεταφράζονται σε ένα πρόγραμμα. Είχα την ευκαιρία λοιπόν να συζητήσω διάφορες ε, πολιτικές μαζί σας με διάφορες συνθέσεις. Βασικό θεσμικό κομμάτι ήταν μια συνάντηση με την διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών ε, ε, η οποία μας έδωσε την ευκαιρία να συζητήσουμε τις προτεραιότητες και τις προσδοκίες μας ε, και εκτιμώ ιδιαίτερο στο εγκάρδιο κλίμα που επικράτησε σε αυτήν την συζήτηση. Η συζήτηση της διάσκεψης των Προέδρων με την Πρόεδρο Φόντερ Λάιεν ε, συνεισέφερε στην αλλαγή του προγράμματος αυτού πριν το εγκρίνουμε χθες. Θα έλεγα λοιπόν ότι αυτή η ειδική σχέση δείχνει πόσο σημαντικό είναι να συνεργαζόμαστε και αυτό θα συνεχιστεί σε ολόκληρη την θητεία μας. Εάν μου επιτρέπετε τώρα θα ήθελα να έρθω στο πρώτο θέμα, το περιεχόμενο του προγράμματος εργασίας. Έχουμε 43 στόχους ή πακέτα όπως λέμε. 28 πρωτοβουλίες θα είναι νομοθετικές για να έχουμε αρκετό χρόνο για την έγκριση και εφαρμογή της. Επίσης εξετάζουμε όλες τις προτάσεις ε, που αναμένουν λήψη απόφασης από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Στην περίπτωση αυτή προτείνουμε να αποσύρουμε 32 από αυτές. Κάποιες από αυτές δεν ανταποκρίνονται στις πολιτικές φιλοδοξίες κομισιών. Για άλλες ε, θα σκεφτούμε πιο φιλόδοξους ε, τρόπους για να επιτευχθούν οι στόχοι. Τέλος, υπό το πρόγραμμα ε, Refit ε, βρήκαμε 44 νομοθετήματα τα οποία θα πάνε προς αναθεώρηση ή αξιολόγηση. Αγαπητοί βουλευτές, σας έχουμε ήδη παρουσιάσει την ανακοίνωση για το πράσινο deal, την στρατηγική της ανάπτυξης και το σχέδιο επενδύσεων για να στηρίξουμε τις περιφέρειες εκείνες που επηρεάζονται περισσότερο από την ενεργειακή μετάβαση. Το επόμενο μεγάλο βήμα είναι η κλιματική νομοθεσία που θα προτείνει δεσμευτικό στόχο κλιματικής οδετερότητα μέχρι το 2050. Θα γίνει μια αξιολόγηση αντικτύπου μέχρι το καλοκαίρι. Στόχος είναι να είμαστε έτοιμοι για την Γλασκόβη την 26η διάσκεψη που έχει προγραμματιστεί για το τέλος Οκτωβρίου. Θα προτείνουμε τη στρατηγική του 2030 για την βιοπικιλότητα για να προστατεύσουμε το φυσικό περιβάλλον και να δούμε ποιες είναι οι φιλοδοξίες μας ε, για την ε, διάσκεψη που έρχεται αλλά και μια στρατηγική από το χωράφι μέχρι το πιάτο και για την βιώσιμη ανάπτυξη. Όλα αυτά λοιπόν θα γίνουν σε συνεργασία με τις περιφέρειες, κοινότητες, ε, σχολεία και άτομα και κοινωνία των πολιτών. Χτες εγκρίναμε την ανακοίνωσή μας για την κινητή τηλεφωνία πέμπτης γενιάς και θα εκδοθεί και μια λευκή βίβλος για την ε, τεχνητή νοημοσύνη. Πρέπει να προστατεύσουμε τα θεμελιώδη δικαιώματα, αλλά θέλουμε να εργαστούμε με την τεχνητή νοημοσύνη. Θα έχουμε λοιπόν προσεχώς τον νόμο περί ψηφιακών υπηρεσιών για να δούμε πώς οι μικρότερες επιχειρήσεις θα μπορέσουν να έχουν ίσους όρους ανταγωνισμού και σαφήνεια του δικαίου όσον αφορά και τον εταιρικό φόρο. Θα ζητήσουμε λοιπόν μια συνολική λύση, αλλά αν αυτό δεν είναι δυνατόν θα σκοπεύσουμε να έχουμε μια ευρωπαϊκή Παράλληλα θα παρουσιάσουμε μια νέα στρατηγική για τις δεξιότητες. Όσον αφορά την οικονομία μας θα προωθήσουμε την κοινωνική δικαιοσύνη όσον αφορά την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση και θα ευθυγραμμιστούν όλες οι πολιτικές μας ε, ενσωματώνοντας τους στόχους του ΟΗΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους ε, εργαζόμαστε σε μια πρωτοβουλία για να διασφαλίσουμε δίκαιο βασικό μισθό για όλους τους εργαζόμενους στην Ευρωπαϊκή Ένωση σεβόμενοι τις ιδιαιτερότητες του κάθε κράτους μέλους. Η Κομισιόν επίσης θα ξαναδεί το πλαίσιο οικονομικής διακυβέρνησης και θα δούμε το πώς λειτουργήσαν οι κανόνες τα τελευταία χρόνια. Θα ξεκινήσουν λοιπόν διαβουλεύσεις με τα κράτη-μέλη και άλλου ενδιαφερόμενους για να δούμε πώς θα μπορέσουμε να βελτιώσουμε το πλαίσιο οικονομικής διακυβέρνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προσεχώς θα εγκρίνουμε ένα σχέδιο δράσης για να εμπαθύνουμε την Ένωση Κεφάλαια Αγορών ε, να βγάλουμε από τη μέση τα εφιστάμενα εμπόδια έτσι ώστε οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να έχουν πρόσβαση στην χρηματοδότηση η ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης, ένα ισχυρό πλαίσιο καταπολέμησης του ξεπλήματος χρήματος, το σχέδιο περί ε, επιδομάτων ανεργίας είναι επίσης προτεραιότητα μας. Όσον αφορά τώρα το γεωπολιτικό πεδίο θα προσπαθήσουμε να συναψουμε συμμαχίες για να προωθήσουμε τις αξίες μας και να προωθήσουμε τα συμφέροντά μας για ανοιχτό και δίκαιο εμπόριο. Θα εντείνουμε τις επαφές μας με τα Δυτικά Βαλκάνια και θα σχεδιάσουμε μια νέα στρατηγική ανατολικής εταιρική σχέσης. Όπως ξέρετε, προσεχώς θα ξεκινήσει και μια νέα στρατηγική με την Αφρική. Η εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να ασχολείται με ζητήματα δημοκρατίας, χρηστής διοίκησης, κλιματικής αλλαγής μετανάστευσης και ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είναι λοιπόν σημαντικό να ενισχύσουμε μια πολυμερή τάξη η οποία θα βασίζεται σε κανόνες. Γι' αυτό ακριβώς θα προχωρήσουμε σε μια αναθεώρηση του ΠΟΕ. Την Άνοιξη θα παρουσιάσουμε το νέο πακέτο για το άσυλο και τη μετανάστευση που θα είναι μια συνολική προσέγγιση που θα καλύπτει όλες τις ε, πτυχές και θα διασφαλίσει μεγαλύτερη συνοχή μεταξύ εσωτερικών και εξωτερικών πολιτικών. Προωθώντας επίσης τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής ε, θα έχουμε ένα σχέδιο δράσης για την ένταξη και μια στρατηγική ασφάλειας Ευρωπαϊκής Ένωσης θα καλύπτει και την ψηφιακή και την ε, ε, φυσική παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης έχουμε ένα σχέδιο για να κατανικήσουμε τον καρκίνο. Βεβαίως θα αναφερθώ και στο κοινό εγχείρημα των τριών θεσμικών οργάνων και σε στενή συνεργασία με τα Εθνικά Κοινοβούλια και τους εταίρους μας για να διοργανωθεί μια διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης οικοδομούμε αυτή τη στιγμή την σχετική δομή μέχρι το τέλος 2020 θα παρουσιάσουμε το σχέδιο δράση για τη δημοκρατία για να δούμε τα θέματα της παλαιοφόρησης των ελεύθερων ΜΜΕ και την ελευθερία λόγου. Όσον αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα η τεχνολογία πρέπει να υπηρετεί τους ανθρώπους και όχι το αντίστροφο και βεβαίως θα πρέπει να δούμε τα ζητήματα τη τεχνητής νοημοσύνης και τη αναγνώριση προσώπου. Τέλος, για το κράτος δικαίου. Η Κομισιόν θα εντείνει το προληπτικό της έργο, παραδείγματο χάρη με την πρώτη έκθεση περί κράτους δικαίου που θα αξιολογήσει την κατάσταση σε όλα τα κράτη-μέλη. Θα πρόκειται για μια έκθεση με εδραία μεθοδολογία που θα αποτελέσει την βάση για το περαιτέρω έργο μας. Επίσης σκοπεύουμε να έχουμε μια Πολιτική στρατηγικής πρόβλεψης των μακροχρόνιων ε, τάσεων για τη χάραξη πολιτικής. Για το σκοπό αυτό ε, έχουμε συστήσει ήδη το σχετικό δίκτυο εντός της ε, Κομισιόν και σε επαφή με εσάς και τα κράτη-μέλη συντονιζόμαστε. Βασίζομαι ιδιαίτερο στην συνεργασία με εσάς. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει πάρα πολλά δεδομένα και αρκετή ευφυΐα στις επιτροπές του. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, ε, αυτή ήταν μια σύντομη παρουσίαση του προγράμματος ε, του 2020. Χρειάστηκα λίγο παραπάνω από 10 λεπτά, αλλά ήθελα να σας πω ότι πραγματικά ε, κάνουμε αυτό το οποίο σας υποσχεθήκαμε. Μια φιλόδοξη αλλά ρεαλιστική ατζέντα για τις προτεραιότητές μας για το πρώτο έτος αυτής της Κομισιόν. Βεβαίως θα έχουμε τη μελλοντική σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο Πρόκειται λοιπόν για μια συγκινητική στιγμή χτες. Ε, θέλουμε όμως να σας διαβεβαιώσουμε πως είμαστε δεσμευμένοι για τη μεγαλύτερη δυνατή διαφάνεια όσον αφορά την ε, διαδικασία αυτή. Μαζί με τους συναδέλφους μου στην Κομισιόν αναμένουμε την συνεργασία μας ε, για την ειδική μας αυτή σχέση. Πρέπει να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να υπάρχει ένας μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός ο οποίος ανταποκρίνεται στις κοινέ μας προκλήσεις και από εδώ και μπρος πρέπει όλοι να εντείνουμε τη δουλειά μας στην διαδικασία λήψης αποφάσεων. Η κοινή δήλωση για τις νομοθετικές προτεραιότητες θα αποτελέσει ένα συγκεκριμένο οδικό χάρτη που θα εμπλέκει και τα τρία θεσμικά όργανα και θα ακολουθήσει το πρώτο πολιετές πρόγραμμα μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Πρόεδρε. Και αραμένω να ακούσω ότι έχουν να πούνε οι βουλευτές. Thank you very much. Σας ευχαριστώ. Για το ΕΛΚ τώρα, Ολμπρίχτ για πέντε λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Η πολιτική μου ομάδα, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, γενικά θα έλεγα ότι υποστηρίζει το πρόγραμμά σας για το 2020. Το έγγραφο το οποίο ε, συμβουλευτήκαμε και αν δεν έχουν υπάρξει τροποποιήσεις από χθε, είναι μια πολύ σημαντική πηγή πληροφοριών που μας επιτρέπει να δούμε το τι σκοπεύει να κάνει το 2020 η Κομισιόν. Πρέπει να ξεπεράσουμε τα συνθήματα, να φανούμε συγκεκριμένοι και γι' αυτό η διαδικασία που ακολουθείτε σήμερα είναι θα έλεγα καθοριστική. Έχουν ολοκληρωθεί οι εκλογικές διαδικασίες, μπορούμε να μιλήσουμε για απόφαση πλέον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και υπάρχουν και αρκετά ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμά σας αν και με κάποιες διαφορές. Πάντως θα θέλαμε ε, η συζήτηση αυτή και η φωνή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να φαίνεται, να ακούγεται στην κοινή δήλωση των τριών Προέδρων. Θα πρέπει να περιλαμβάνεται επίσης και στα πλαίσια του πολιετούς δημοσιονομικού. Έχει σημασία για μας για να δούμε ποιες είναι οι διαδικασίες που ακολουθήθηκαν και τι έχει αλλάξει ή και τι έχει εγκαταλειφθεί. Θα θέλαμε από εδώ και πέρα οι συνομοθέτες να δράσουν με υψηλή ταχύτητα και να επιταχύνουν γενικότερα το νομοθετικό τους έργο. Ελπίζουμε συνεπώς ότι όλα τα θεσμικά όργανα θα ακολουθήσουν υψηλές πλέον ταχύτητες. Σχετικά με την ουσία τώρα της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει μια αντίληψη γεωπολιτική και στα πλαίσια της αντίληψης αυτής ε, θα έλεγα υπάρχουν και θέματα εσωτερικά μεν που επηρεάζουν όμως και τα εκτός. Καταρχάς συμφωνούμε ότι τα βασικά στοιχεία πάνω στα οποία ε, πατάμε είναι το Green Deal όπως λέμε, είναι η υπογράμμιση της σημασίας του ψηφιακού κόσμου και μάλιστα σε σχέση με το Green Deal έχετε κάποιες προτάσεις ε, για θέματα όπως η οικονομία ε, των δασικών περιοχών. Πολύ σημαντικά για πολλές χώρες. Στο έγγραφο λοιπόν της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν μένουμε σε κάποιες ε, θεωρητικές διαπιστώσεις αλλά συζητιώνται πρακτικά θέματα. Το ίδιο ισχύει και για την ε, ψηφιακή οικονομία. Αναφέρεστε στον τομέα της έρευνας, της ανάπτυξης, δεν είναι μόνο τεχνολογικό, είναι και πιο πολιτικό, είναι και πιο οικονομικό. Γενικά είναι δοσμένα τα στοιχεία με οριζόντιο τρόπο για την αγορά κεφαλαίων και τα κοινωνικά χαρακτηριστικά. Έχει σημασία για μας που είμαστε ένα κόμμα χριστιανοδημοκρατικής προέλευσης. Για πάρα πολλά χρόνια ακούγαμε να συζητάμε για τη στρατηγική για την Αφρική. Άλλαξε αυτό. Τώρα λέτε στρατηγική πολιτική με την Αφρική. Αυτό είναι πολιτική δήλωση, διαφοροποίηση. Τι θα κάνει η Επιτροπή λοιπόν, θα πρέπει να δουλέψει με την Αφρική και όχι για την Αφρική. Παρατηρούμε επίσης με ενδιαφέρον ότι θέλετε ε, σε ετήσια βάση να ε, συντάσετε μία έκθεση για το κράτος δικαίου. Πολύ καλή ιδέα. Και μία κριτική τώρα για το τέλος. Για μας το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο το πι δελτα πι λοιπόν ε, δεν είναι αυτός σκοπός. Πριν δημιουργήσουμε ε, τις πολιτικές θα πρέπει να γνωρίζουμε τι μέσα έχουμε και είναι κάτι το οποίο θα έλεγα θα παίξει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο, θα παίξετε ρόλο διαιτητή. Ε, δεν έχουμε να κάνουμε με μια λογιστική συζήτηση αλλά με μια πολιτική συζήτηση και έχετε σαν Επιτροπή συγκεκριμένο ρόλο. Στηρίζουμε λοιπόν την πρότασή σας για το 2020. Ευχαριστώ για τους σοσιαλδημοκράτες. κυρία Γκαρθία Πέρεθ για 3,5 λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Αντιπρόεδρε, η δικιά μας πολιτική οικογένεια εκτιμάει θετικά τις κύριες προτάσεις σας όσον αφορά την οικολογική αλλαγή, την οικονομική κτλ. Πράγματα τα οποία χρειάζονται και χαιρόμαστε που συμπεριλαμβάνονται στο πρόγραμμα εργασίας σας. Πρόκειται για ένα εξαιρετικό παράδειγμα συνεργασίας ανάμεσα σε εσά κύριε Σεύκοβιτς και το κοινοβούλιο μας. Γενικά μιλώντας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πολύ σωστά εντόπισε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα το ευρωπαϊκό οικοδόμημα αλλά και τα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας ή που χρειαζόμαστε για να υλοποιηθούν οι πολιτικές αυτές. Αλλά ο διάβολος όπως γνωρίζετε βρίσκεται στη λεπτομέρεια και πιστεύουμε ότι η πρόταση αυτή ε, δεν έχει λεπτομέρειες, λείπουν κάποια πράγματα. Γι' αυτό και θέλω να ρωτήσω και να σας πω ότι η στήριξη της δικιάς μας ομάδας στην Επιτροπή δεν είναι επιταγή λευκό. Θα παρακολουθούμε από κοντά τι γίνεται με την υλοποίηση κάθε μία από τις προτάσεις αυτές. Το πρόγραμμα εργασίας συμπεριλαμβάνει τα μέσα επίσης για την υλοποίηση της Πράσινης Συμφωνίας μέσα από μια δίκαια μετάβαση. Όμως λυπούμαστε που δεν συμπεριλαμβάνεται τίποτα για την μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα για το 2050. Η Επιτροπή το είχε πει εδώ και εμείς πιστεύουμε ότι έτσι θα καταπολεμήσουμε την κλιματική αλλαγή και ελπίζουμε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο να δείξουν ότι και αυτοί θέλουν να κάνουν την προσπάθεια. Η κλιματική ουδετερότητα θα παραμείνει λόγια κενά περιεχομένου Επίσης, περιμένουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάτι πιο συγκεκριμένο, να αναγνωρίσει την ευκαιρία που αποτελεί η μετανάστευση για να αντιμετωπιστεί το δημογραφικό πρόβλημα και να συνεχίσουμε να χαίρουμε από ένα κράτος ευημερία. Και πώς θα εντάξουμε τους πρόσφυγες της κοινωνίας μας. Χτες εδώ στο Κοινοβούλιο συζητήσαμε για την κατάσταση των προσφύγων στα ελληνικά νησιά. Δεν μπορούμε να καθυστερήσουμε άλλο ούτε ένα λεπτό. Μιλάμε για τη ζωή, για την αξιοπρέπεια χιλιάδων ανθρώπων οι οποίοι περιμένουν την αλληλεγγύη από εμά και κάποια υπευθυνότητα από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά η αλληλεγγύη σημαίνει συγχρόνω το ευρωπαϊκό σχέδιο για κοινωνικά δικαιώματα. Να υλοποιηθεί επίση και να συμπεριλάβουμε και την εγγύηση για τα παιδιά ώστε να μην υπάρχει φτώχεια για τα παιδιά. Χρειαζόμαστε ένα πλαίσιο επίση για ελάχιστου μισθού που είναι αξιοπρεπή για του εργαζόμενου. Αλληλεγγύη επίση σημαίνει μια προσπάθεια ακόμα από την Ευρώπη ε, απέναντι στου γείτονέ μα που έχουν δεχτεί τι δικέ μα αξίε και αρχέ. Άρα πρέπει να αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις με την Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία. Αλληλεγγύη επίσης σημαίνει και προστασία και ενίσχυση των δημοκρατιών μας. Εξού και πρέπει να υπάρχει ένας νέος μηχανισμός για την διασφάλιση του κράτους δικαίου. Να είμαστε σοβαροί. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο εφόσον υπάρξει μια συμφωνία για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Και εδώ θέλω να κάνω έκκληση απέναντι στο Συμβούλιο να αναλάβει την ευθύνη για να υπάρξει συμφωνία πάνω σε αυτό το θέμα για να πετύχουμε όλους αυτούς τους στόχους. Αλλιώς δεν θα τα καταφέρουμε δεν θα τα καταφέρουμε να χρησιμοποιήσουμε τα μέσα τα οποία τόσο πολύ χρειαζόμαστε. Το οφείλουμε να τηρήσουμε τις υποσχέσεις μας. Γι' αυτό ζητούμε υπευθυνότητα από την Επιτροπή και από το Συμβούλιο, ώστε από κοινού να κάνουμε πραγματικότητα την Ευρώπη που τόσο πολύ χρειάζονται οι πολίτες μας. Ευχαριστούμε εκ μέρους του Ρινιού. Ο κύριος Τσόλος έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Ξεκινάει η εντολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Είμαστε και συνέθετοι εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θέλουμε φιλοδοξίε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα ψηφιακά, για την Πράσινη Συμφωνία για παράδειγμα, που θα ανανεώσουν πλήρω την οικονομία και τον τρόπο ζωή στην Ευρώπη. Το αποτέλεσμα τη θητής αυτή θα εξαρτηθεί σε ένα μεγάλο βαθμό από το κατά πόσο θα μπορέσουμε να υλοποιήσουμε του στόχου μα, αλλά πρέπει να δούμε και ποιοι θα είναι οι πόροι που θα έχουμε στη διάθεσή μα για να υλοποιηθούν όλοι αυτοί οι στόχοι. Χρειαζόμαστε πολιετέ δημοσιονομικό πλαίσιο, φιλόδοξο, στο ύψο των ε, στόχων μας. Ούτε φτάνει να στηρίξουμε τον ιδιωτικό τομέα ε, και τις χώρες μέλη για την αναδιάρθρωση των οικονομιών. Ελπίζω να έχουμε ολοκληρωμένα οικονομικά μέσα που να συμπληρώνουν το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο και τον προπολογισμό και τα νομοθετικά μέτρα που περιμένουμε από εσά πρέπει να προσφέρουν λύσεις. Πολλές φορές Νομίζει ο κόσμο ότι η Ευρώπη το μόνο που κάνει είναι ότι όλο και περισσότερε ρυθμίσει υιοθετεί. Εμεί θα πρέπει να προσφέρουμε μια πραγματική ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία με μέτρα που θα προτείνουμε εδώ, τα οποία θα οδηγούν στην ευημερία, θα οδηγούν στην προστιθέμενη αξία, πέρα από αυτά που μπορούν από μόνοι του να καταφέρουν οι χώρε μέλη. Η ομάδα μα λοιπόν δεν πρόκειται να περιμένει τι προτάσει τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχουμε ήδη τι δικέ μα ιδέε και τι δικέ μα προτάσει για το ποια θα πρέπει να είναι η λύση για το ζήτημα της μετανάστευσης, πόσο πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή η Πράσινη Συμφωνία. Και τις επόμενες μέρες θα παρουσιάσουμε και την άποψή μας για το πόσο πιστεύουμε εμείς ότι πρέπει να ρυθμιστεί η τεχνητή νοημοσύνη πέρα από την ευμερία και τον πλούτο, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να διασφαλίσει στους πολίτες να ε, κυκλοφορούν ελεύθερα για να εργάζονται ή να σπουδάζουν αλλού, αλλά επιπλέον όλες οι χώρες να σέβονται το κράτος δικαίου και τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όταν παραβιάζονται οι αρχές του κράτους δικαίου θα πρέπει να υπάρχουν συνέπειες. Ανεξάρτητα από το για ποια χώρα μέλος πρόκειται πρέπει να είναι ξεκάθαρο το σχέδιο επ' αυτού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Την επόμενη εβδομάδα το Ηνωμένο Βασίλειο θα αποτελεί μια τρίτη χώρα για μας. Πρέπει να πάρουμε τα μαθήματα του παρελθόντος, τι σημαίνει το Brexit τελικά. Και η διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης θα μπορούσε να μας επιτρέψει ακριβώς όλες αυτές τις ιδέες και τα μαθήματα που έχουμε πάρει να τα συγκεράσουμε πρέπει να γίνει αυτή η συζήτηση με τους πολίτες. Γιατί πρέπει με τους εκλογείς μας, οι οποίοι μας έφεραν εδώ, να μοιραστούμε όλες αυτές τις ιδέες και τις λύσεις για το μέλλον. Ευχαριστώ. Η κυρία Κέλλερ για δύο λεπτά. Αγαπητοί συνάδελφοι, πρόκειται για μια στιγμή δραματική και θλιβερή η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου. Αλλά εγώ δεν δέχομαι ότι είναι το τέλος ούτε βεβαίως θα τερματίσει η φιλία μεταξύ των Βρετανών και της Ευρωπαϊκής Υπήρου, ούτε παρετούμαστε από την ελπίδα ότι θα επιστρέψει κάποια στιγμή το Ηνωμένο Βασίλειο εδώ που ανήκει. Αλλά, ενώ πρόκειται για μια θλιβερή στιγμή, ε, δεν είναι μια στιγμή που μας φέρνει πιο κοντά σε οποιοδήποτε τέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως θα ήθελαν κάποιοι. Κάθε άλλο. Αν δεν είχαμε την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα έπρεπε τώρα να την εφεύρουμε και οι Ευρωπαίοι ενώθηκαν γιατί υπάρχουν κάποια προβλήματα που μπορούν να λυθούν μόνο από κοινού και ε, ενωμένοι είναι πιο ισχυροί και υπάρχουν πολλές προκλήσεις σήμερα και πρέπει να τις αντιμετωπίσουμε. Γι' αυτό είναι τόσο σημαντικό αυτή την εβδομάδα να συζητήσουμε και το πρόγραμμα εργασίας. Έτσι θα δείξουμε τι αξίζουμε. Και η Κομισιόν ανέφερε στην ομιλία τη ε, την κλιματική κρίση που είναι μια τεράστια πρόκληση που αντιμετωπίζει κάθε χώρα σε κάθε ήπειρο και έχει φτάσει η στιγμή να δράσουμε κατεπηγόντω. Χαιρόμαστε για το ότι η Κομισιόν δίνει έμφαση σε πρωτοβουλίε που αντιμετωπίζουν το θέμα του κλίματο και τη βιοπικιλότητα. Βεβαίω είναι πάρα πολύ νωρί να πούμε αν επαρκούν. Αυτό θα εξαρτηθεί από τι λεπτομέρειε τη πρότασή σα αλλά θα εξαρτηθεί και από το αν η πλειοψηφία του Κοινοβουλίου θα υποστηρίξει φιλόδοξη νομοθεσία και τα κράτη-μέλη βεβαίως. Οπότε θα εξαρτηθούν αυτά από όλους μας ε, πόση κλιματική δράση θα αναλάβουμε και πόσα θα συνεισφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση στις παγκόσμιες προσπάθειες αφού είχε συνεισφέρει στην καταστροφή του πλανήτη. Η Κομισιόν επίσης ε, είναι ο θεματοφύλακας ε, των ε, συνθήκων και θα πρέπει πράγματι τα κράτη-μέλη να μην αποκλίνουν από το κράτος δικαίου. Θα πρέπει λοιπόν να κινητοποιηθούμε και φέτος θα δείξουμε προς τα πού πηγαίνει η Κομισιόν. Χρειάζονται θαραλέα βήματα προς τα εμπρός για μια νέα Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την ομάδα ID. Τον λόγο έχει ο κύριος Βιλίμσκι για ένα λεπτό. Με συγχωρείτε επί της διαδικασίας, κύριε Σφέστ. Κοιτάξτε, δεν έχω ε, όρεξη να μιλάω κάθε λίγο με τους κλητήρες για τις σημαίες. Ε, δεν είναι δική σας δουλειά η διεύθυνση της ε, συνεδρίασης όμως, λέει η πρόεδρος. Χωρίς μικρόφωνο ο μιλητής. Δεν έχετε το μικρόφωνο. Λοιπόν, θα τα ξεκαθαρίσουμε αυτά, αλλά ένα είναι σαφές. Ο κανονισμός είναι σαφής. Το είπαμε χτες και στην συζήτηση του Brexit. Θα λαμβάνουν τον λόγο μόνο όσοι τηρούν τον κανονισμό. Το έχουμε πει πολλές φορές. Αν δεν συμφωνείτε, υπάρχει ο τρόπος να διαμαρτυρηθείτε δεν θα συζητηθεί πλέον στην Ολομέλεια όποιος έχει σημαιακια δεν θα λαμβάνει το λόγο επί της διαδικασίας πάλι θα ήθελα να μάθω ποιο άρθρο του κανονισμού είναι αυτό στο οποίο αναφερθήκατε για να μην δίνετε το λόγο στους συναδέλφους μου ο συνάδελφος ε, μίλησε για την διεύθυνση της συζήτησης. Κοιτάξτε, δεν είναι ε, δουλειά του ε, βουλευτού αυτό, είναι θέμα σεβασμού του προεδρεύοντος. Έχει ξεκαθαρίσει πολλές φορές το ζήτημα, λοιπόν σας παρακαλώ να χρησιμοποιήσουμε το χρόνο για την συζήτηση. Ο κύριος Βιλίμς και έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Κοιτάξτε, μέχρι τώρα πάντα ασκούσα κριτική στην Κομισιόν. Σήμερα θα κάνω μία εξαίρεση και θα ήθελα να τους επενέσω γιατί το πρόγραμμα που παρουσίασε είναι ένα πρόγραμμα το οποίο ε, θα καταφέρει να λύσει τα ζητήματα ασύλου και μετανάστευσης. Ε, τα προβλήματα του νομίσματος με μηδενικά επιτόκια θα καταφέρουν ως διαμαγείας να εξαφανίσουν την αναργία. Αυτό το οποίο θα κάνουν όμως τελικά είναι ένα Green Deal με το οποίο θα πάρουν ακόμα περισσότερα λεφτά από τις τσέπες των ανθρώπων. Αν είναι κάποιος ε, έτσι ευγενικός θα μπορούσε να μιλήσει για μια κομισιόν Χάρι Πότερ. Αλλιώς θα το έλεγε απλά βουντού. Κυρίες και κύριοι, χτες έφυγαν οι Βρετανοί από εδώ και απευθύνω έκκληση. Εάν δεν θέλετε να δείτε κι άλλη χώρα να αποχωρήσει, πρέπει να συγκεντρωθείτε στα μεγάλα και τα σημαντικά. Άσυλο, μετανάστευση, οικονομία και νόμισμα, κοινωνικά και αγορά εργασίας. Εκεί πέρα περιμένουμε αποτελέσματα και όχι αυτά τα οποία μας λέτε ότι θα γίνουν ως διαμαγείας. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, η κυρία Νικολσόνοβα τώρα για το ECR. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, ε, το πρόγραμμα εργασίας Κομισιόν προσπαθεί να έρθει πιο κοντά στους ε, πολίτες. Ε, καμιά φορά μιλάμε για λαϊκισμό. Αλλά ο Βασικό μισθός ε, θα μας απασχολήσει για δύο χρόνια. Τελικά δεν θα έχει αποτέλεσμα γιατί ήδη πολλές χώρες έχουν ε, βασικό μισθό και επίση ε, θα είναι πάρα πολύ υψηλό, ειδικά στι νέε χώρε. Πολλοί κόσμοι περιμένει ότι μια μέρα στην άλλη θα πάρει μια αύξηση. Θα απογοητευτεί. Και τελικά θα ρίξουμε νερό στο μήλο των λαϊκιστών. Λοιπόν, εκτιμώ πολύ το ότι έχετε εκεί πέρα την ε, ψηφιοποίηση και τα σχετικά και την εγγύηση για τα παιδιά. Τα παιδιά χρειάζονται πρόσβαση σε καλές υπηρεσίες. Η Νέα Κομισιόν υποσχέθηκε ότι ε, θα ε, κάνει κάτι για το θέμα αυτό και αυτό αναμένουν Σλοβάκοι και λοιποί στους οποίους ε, περικόψαν τα επιδόματα παιδιών. Τρία λεπτά κύριε Ομπρή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αυτή η εβδομάδα είναι μια κρίσιμη καμπή στην ευρωπαϊκή ιστορία με την αποχώρηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση του Ηνωμένου Βασιλείου. Το χειρότερο θα ήταν να μην πάρουμε κανένα μάθημα και να συνεχίσουμε σαν να μην έχει συμβεί τίποτα. Να μην αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει μια απόσταση που όλο και μεγαλώνει ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τι χώρε μέλη. Ακριβώ αυτή είναι η πρόκληση που πρέπει να καθοδηγήσει το πρόγραμμά σα για ε, την ε, χρονιά αυτή. Θα σας μιλήσω για κάποιου πολίτες. Τι λέω, που συνάντησα σε μια οργάνωση, σε μια εκδήλωση για το κλίμα που μου μίλησε για το οικονομικό μοντέλο μας που καταστρέφει και τον πλανήτη. Τι θα κάνει και πώς θα εκπλαγεί όταν διαπιστώσει ότι τελικά δικιά σας Ευρωπαϊκή Συμφωνία ακολουθεί το δόγμα της οικονομικής μεγένθησης και κάνει λιγότερα για το κλίμα. Και άλλοι ζητούν κάποια συνοχή και δεν καταλαβαίνουν γιατί στηρίζεται τις μεγάλες βιομηχανίες ε, του αγροτροφικού τομέα. Και φανταστείτε και το θυμό τους για τις συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών που προβλέπει να υπογράψει ακόμα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ΛΕΑ θα ήλπιζε η Ευρωπαϊκή Ένωση να στηρίξει τα προϊόντα Κίνα, τα οποία δεν κάνουν τρει φορές στο γύρο του πλανήτη πριν καταλήξουν στο πιάτο μας. Η ΛΕΑ ελπίζει μια πραγματικά κοινωνική νέα πράσινη συμφωνία με κατάλληλα μέσα. Η αναθεώρηση του εξαμήνου του Ευρωπαϊκού θα πρέπει να δώσει τα μέσα για μια πιο οικολογική προσέγγιση. Η Μαρή που είναι νοσοκόμα σε ανεργία, σε απεργία, συγγνώμη, εδώ και καιρό γιατί δεν καταλαβαίνει πώς είναι δυνατόν η Ευρωπαϊκή Ένωση ενθαρρύνει την ιδιωτικοποίηση των δημοσίων υπηρεσιών μας και τη κοινωνικής προστασίας. Έχει δουλέψει κάποιος άλλος για την Καστόραμα. Έχασε τη δουλειά του όμως στην Πολωνία γιατί αλλού η εργασία στοιχίζει φθηνότερα. Δεν πρόκειται όμως να πετύχει η πρότασή σας με τα μέτρα τα οποία προβλέπετε. Έπειτα πρέπει να σταματήσει η εκμετάλλευση των εργαζομένων που βρίσκονται σε επισφαλή εργασία. Η Μαρία, Πιέρ, Κέβιν δεν καταλαβαίνουν γιατί αυξάνονται οι φόροι τους ενώ οι πολυεθνικές δεν πληρώνουν φόρους και δεν καταλαβαίνουν πώς είναι δυνατόν να δέχεστε την επιρροή των λόμπι στις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το πρόγραμμά σας δεν βρήκα καθόλου ίχνη ηθικής που υποσχεθήκατε όμως εσείς για τις πολιτικές αυτές. Οπότε για αυτή την αγανάκτηση θυμό τι τις ελπίδες, τι θα κάνετε. Πρέπει να δράσετε. Αν δεν το κάνετε για την ομάδα μας Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς, για τους βουλευτές που βρίσκονται εδώ στο ημικύκλιο, τότε κάντε το για τη Λέα, για τη Μαρή, για τον Πιέρ, για τον Κέβιν και για τόσους άλλους Ευρωπαίους πολίτες, οι οποίοι δεν θα σας συγχωρήσουν αν επιμείνετε να ακολουθήσετε και φέτος τις ίδιες συνταγές οι οποίες οδήγησαν στην κλιματική κρίση και στην αύξηση των ανισοτήτων στην Ευρώπη. Ευχαριστώ. Ολοκληρώσαμε τον γύρο των ομιλητών των ομάδων. Είχαμε και ένα θέμα το οποίο αναβάλαμε από χτες. Παρακαλώ λοιπόν να είστε σύντομοι. Σίντσιτς για 1,5 λεπτό. Επίτροπε Σεύκοβιτς αναφερθήκατε στο πρόγραμμα εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφερθήκατε επίσης και για τη δημοκρατία και τις εξωτερικές σχέσεις Χονγκ Κόνγκ, Βολιβία, Βενεζουέλα, Αφρικανικές χώρες αλλά το θέμα με τη δημοκρατία είναι κάτι το οποίο δυσκολεύει και ακόμα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην Κροατία το 2000 14 είχαμε περισσότερους εκλογείς 400.000 περισσότερους από τους πραγματικούς εγγεγραμμένους τους εκλογικούς καταλόγους. Το ε, φέτος οι 400.000 έγιναν 200.000 Δεν χρειάζεται να υπογράφει κανείς τον εκλογικό κατάλογο για να αποδειχθεί ότι πήρε μέρος στις εκλογές. Δημιουργούνται καταστάσεις αντιδημοκρατικές και ενάντια στην ίδια τη λογική. και γενικά η νομοθεσία γύρω από τις εκλογικές διαδικασίες είναι απαράδεκτη αλλά το κρατικό καθεστώς δεν θέλει να αλλάξει και αυτό αποδεικνύει το πόσο διεφθαρμένο είναι. Είναι παράλογο λοιπόν ο Κροάτης Επίτροπος να είναι υπεύθυνο για τέτοια θέματα. Ευχαριστώ Νίμπλερ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κυρία Αντιπρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Θεωρώ πως η Κομισιόν έχει ένα φιλόδοξο πρόγραμμα για το 2020, έχει δώσει έμφαση στα σωστά πράγματα, βεβαίως το θέμα τώρα είναι η εφαρμογή. Και εδώ πέρα σημασία έχει η ποιότητα και όχι η ποσότητα, οπότε καλύτερα μια αξιολόγηση αντικτύπου πριν παρά μια λανθασμένη νομοθεσία. Για το πράσινο ντύλι ήδη ακούστηκαν αρκετά θα ήθελα να αφαιρθώ σε άλλα πράγματα. Πρώτον, θεωρώ ότι είναι θετικό ότι προσεχώς θα υπάρχει μία βάση συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη και μία στρατηγική για τα δεδομένα και με μεγάλη μου χαρά άκουσα το ότι θα αποτελέσει βασικό κομμάτι εδώ πέρα η ασφάλεια των δεδομένων. Χαίρομαι ιδιαίτερος για το ότι τον Μάρτιο θα υπάρξει και μία βιομηχανική στρατηγική και θα δοθεί βάρος στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, ε, στις οικογενειακές επιχειρήσεις. Εκεί πέρα είναι οι θέσει εργασίας, εκεί πέρα δημιουργούνται οι δουλειές, εκεί εκπαιδεύονται οι νέοι. Καλό είναι λοιπόν το ότι η νέα Κομισιόν εστιάζει ειδικά στις ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και τέλος, ε, μετανάστευση, ένα βασικό θέμα Αναμένω λοιπόν τις νέες σας προτάσεις. Αν δεν το λύσουμε αυτό θα έχουμε μακροπρόθεσμα πρόβλημα. Ευχαριστώ. Ακολουθεί η κυρία Μποναφέ για ένα μισή λεπτό. Ευχαριστώ πρόεδρε. Εμείς έχουμε παρουσιάσει το, ή μάλλον βλέπουμε το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τις προτεραιότητές της και μας ικανοποιεί γενικά. Αλλά παρόλα αυτά για κάποια κεντρικά θέματα περιμέναμε περισσότερο. Σαν παράδειγμα στη Νέα Συμφωνία για την Μετανάστευση, η οποία βάζει στο κέντρο την αλληλεγγύη ανάμεσα στα κράτη. Περιμέναμε περισσότερα για να πιο ε, ήρεμη και ισορροπημένη πρόταση στον τομέα της φοροαποφυγής των μεγάλων επιχειρήσεων επίσης και για την καταπολέμηση της φτώχειας ε, διότι δυστυχώς χωρίς πόρους ε, κύριε Σεύκοβιτ δεν γίνεται τίποτα για το Green Deal όλος ο κόσμος βλέπει αυτό το οποίο θέλουμε να κάνουμε καλά είναι αυτά τα δίστα οποία προβλέπατε αλλά θα θέλαμε περισσότερα χρήματα από τώρα για το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης που να μην τα αφαιρείται από άλλα ταμεία. Συνεπώς λοιπόν έχει μεγάλη σημασία να δούμε με ποιο τρόπο μπορούμε να κάνουμε τις αλλαγές αυτές και στον οικονομικό τομέα. Στο πρόγραμμα δεν υπάρχει καμία υποχρέωση που να αναλαμβάνεται για το ε, σύμφωνο ε, ανάπτυξης ε, ε, αν δεν υπάρξει ανάπτυξη δεν υπάρχει σταθερότητα. Η ανάπτυξη θα δώσει μεγαλύτερη ευελιξία στα κράτη και για τις επενδύσεις και στον τομέα της πράσινης οικονομίας. Υπάρχουν πάρα πολλές προκλήσεις και ελπίζω η Επιτροπή να μπορέσει να κάνει περισσότερα από όσα έχει ήδη πει. Ευχαριστώ Ασμάνη για ένα λεπτό. Ναι, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ήμουν παρόν αυτή την εβδομάδα στο Auschwitz-Birkenau με την αντιπροσωπεία του κόμματός μας και χτες ακούσαμε τα εντυπωσιακά λόγια της ε, κυρίας Σέγερ. Οι μνήμες της ε, μας υπενθυμίζουν ε, το πώς είναι ένας κόσμος χωρίς σεβασμό για τις φιλελεύθερες αξίες. Μας υπενθυμίζουν ότι δεν είναι δεδομένες αυτές οι αξίες. Ο αντισημιτισμός εξακολουθεί να υπάρχει στην Ήπειρό μας το κράτος δικαίου υφίσταται πίεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ΡΙΝΙΟΥ καλωσορίζει την φιλοδοξία της Κομισιόν να καταστήσει τις ευρωπαϊκές αξίες ε, και το κράτος δικαίου προτεραιότητα, αλλά χρειαζόμαστε δράση, ένα μηχανισμό κράτους δικαίου. Υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις που πρέπει να δούμε. Χρειαζόμαστε μία προσέγγιση για τη μετανάστευση να ανακτήσουμε έλεγχο. Γι' αυτό προτείναμε ένα σχετικό πακέτο πριν από λίγε εβδομάδε, μια συνολική απάντηση. Τώρα λοιπόν πρέπει η Κομισιόν να δράσει. Ο μετασχηματισμός της οικονομίας μας σε μια πράσινη και καινοτόμο οικονομία είναι άλλη μια προτεραιότητά μας. Και στην παγκόσμια σκηνή πρέπει να εκμεταλλευτούμε την οικονομική μας δύναμη μαζί με διπλωματία και την αμυντική πολιτική. Μόνο τότε θα γίνει ένας παγκόσμιος παίκτη η Ευρωπαϊκή Ένωση και ζητώ από την Κομισιόν να αγκαλιάσει και την δική μας ε, τη φιλοδοξία για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στην υπόσχεση της Ευρώπης. Σας ευχαριστώ. Άντερσον για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ Θα ήθελα να πάρω το λόγο εξ ονόματος του λαού της Σκωτίας. Σας ευχαριστώ για τις προσπάθειες που κάνατε τις τελευταίες ε, εβδομάδες δυστυχώς η κάρτα αυτή θα ισχύσει μόνο για λίγες μέρες ακόμα αλλά θα συνεχίσουμε τις συζητήσεις και για την Πράσινη Συμφωνία και για την αηφόρο γεωργία και άλλους τομείς. Η εκκλησία μου είναι να μην ξεχνάτε τη Σκοτία παρακαλώ στο πρόγραμμα εργασίας σας ε, για μια χώρα σαν τη Σκοπία η οποία είναι πιστή στην Ευρώπη. Τρεις φορές το έχει επιβεβαιώσει αυτό, τώρα απομακρύνεται. Ε, εμείς δεν ζούμε στο Ηνωμένο Βασίλειο, ζούμε σε ένα βασίλειο που μόνο ενωμένο δεν είναι, αλλά ναι. είμαστε ανθεκτικοί και θα αντέξουμε ακόμα και τώρα, μοιραζόμαστε την ιστορία μας ε, με ε, την Ευρώπη και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε και στο μέλλον. Αύριο θα καταθέσει η κυβέρνηση της Σκοτίας τις ε, προτάσεις της για τις προοπτικές και αν είναι να διαλέξουμε ανάμεσα σε δύο ενώσεις είναι προφανές ότι θα διαλέξουμε εμείς στη Σκοτία την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κύριος Ριβιέρ, σας παρα... έχετε προειδοποιηθεί ότι τον λόγο λαμβάνουν μόνο τηρούν τους κανόνες, δεν τηρήσατε τους κανόνες, δίνω τον λόγο στον κύριο Λούντγκρεν. Α, κατεβάστε τη σημαία. Και θα μείνει κάτω. Ωραία. Έχετε τον λόγο λοιπόν. Ευχαριστώ. Ναι, κατεβάσω τη γαλλική σημαία, όχι για να τιμήσω αυτό το σώμα για να δεχτώ μια ήττα, αλλά για να έχω την ευκαιρία να απευθυνθώ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τους συναδέρφους και να σημειώσω, ξέρετε, σήμερα στον εσωτερικό κανονισμό του Κοινοβουλίου μας δεν απαγορεύει την παρουσία αυτής της σημαίας, η οποία προστατεύεται από το άρθρο 2 του Γαλλικού Συντάγματος άρα από μια νομοθεσία. Αλλά αυτή η τρίχρωμη σημεία, ε, σημαία ενσωματώνει όλα όσα τελικά μισή αυτή η Ευρώπη όπως μισεί τους λαού, Ο Αλεξάνδρ Σολβενίτσι μας προειδοποίησε εδώ και καιρό ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση φέρει μέσα της ε, τη, τον ολοκληρωτισμό. Χτες όλοι ακούσαμε με συγκίνηση την κυρία Σέγκρε και ενώ τιμούσαμε την απελευθέρωση του στρατόπεδου του Auschwitz, μας εξήγησε τη συγκίνησή της όταν μπήκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δύο φορές είπε πόσο συγκινήθηκε όταν είδε όλες αυτές τις σημαίε, σημαίε των εθνών όχι ιδιαίτερα από την ευρωπαϊκή σημαία. Μα ακούστε την. Τα λόγια της έχουν νόημα. Οι λαοί δεν θέλουν πια αυτή τη γραφειοκρατία. Αλλά απέναντι στους λαούς τι κάνετε. Την Παρασκευή φεύγουν οι Βρετανοί. Θα πρέπει να τους ακούσετε. Το ευρωπαϊκό σχέδιο ήταν ωραίο σχέδιο, αλλά η ιστορία θα σας κρίνει αυστηρά. Και να ξέρετε ότι αυτή η πρώτη αποχώρηση είναι το πρώτο χτύπημα ε, που φέρετε σε αυτόν τον τείχο ολοκληρωτισμού που είσαστε εσείς. Δεν έχουμε ε, κάποιο πρόβλημα με τις σημαίες, είναι εδώ από πίσω μας. Όλοι είμαστε περήφανοι για αυτές τις σημαίες, αλλά όλες μαζί όχι ο καθένας στο έδρανό του. Σας ευχαριστώ Λούντκριν για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να αναφερθώ σε κάτι, λέτε εδώ πέρα νέα όθηση για την ευρωπαϊκή δημοκρατία. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας αποσχολήσει στην σημερινή συζήτηση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μια δημοκρατία η οποία δεν υπάρχει σε άλλα μέρη. Ε, η εθνική αυτοδιάθεση είναι ένας σημαντικός ε, στόχος όπως και η κυριαρχία των ε, διαφόρων εθνών. Εδώ πέρα λοιπόν ισχύει ο κανόνας ότι δεν επιτρέπονται οι εθνικές σημαίες. Και στην ψηφοφορία όμως πάλι θα εμφανιστούν σημαίες. Αν θέλετε να τα απαγορεύσετε πρέπει να είμαστε συνεπείς. Ε, να δεχτώ λοιπόν μια απόφαση να μην υπάρχουν ε, σημαίες στην αίθουσα. Ε, δεν πρέπει να υπάρχουν και αυτές οι σημαίες εδώ πάνω και η σημαία ευρωπαϊκή. Σας υπενθυμίζω ότι το, το θέμα το οποίο συζητάμε είναι το πρόγραμμα της Κομισιόν για το 2020. Καλό είναι να συζητάμε αυτό το θέμα. Α, καταλαβαίνω βεβαίως ότι το θέμα είναι ε, έντονο και θελήσατε να μιλήσετε γι' αυτό. Α είναι. Λοιπόν, τον λόγο έχει η κυρία Μπιόρκ για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να πω ότι ολοκληρώνεται μια διαδικασία η οποία είχε ξεκινήσει εδώ και ε, πάρα πολλά χρόνια. Κανονικά θα πρέπει να κάνουμε την αυτοκριτική μας, αλλά δεν το κάνει ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ασχολείται με ένα πρόγραμμα εργασίας το οποίο επίσης ε, να ε, αναφέρεται στα θέματα της σωστής παρουσίας της Ευρώπης στον υπόλοιπο κόσμο και στα πλαίσια των Ηνωμένων Εθνών. Υπάρχουν τώρα κάποια επιμέρους θέματα. Καταρχάς, κλιματολογικές αλλαγές, βιοπικιλότητα. Όχι μόνο 50% αλλά 80% το 50%. Επίσης στον τομέα των, της κρίσης στην οποία ε, βρισκόμαστε ακόμα, οι αντιδράσεις έτσι όπως τις προβλέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αρκούν. Σας ευχαριστώ. Τέναντ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μετά την ιστορική ψηφοφορία χτες, ένας ε, συνάδελφός μας ζήτησε εδώ πέρα να τραγουδήσουμε το Old Lang Syne οι λαοί της Ευρώπης είναι φίλοι μας, πάντα ήταν και πάντα θα είναι. Δεν έχουμε κάποια διαμάχη με τους λαούς αυτής της απίστευτης Υπήρου. Απλά με τις πολιτικές δομές και τα θεσμικά όργανα τα οποία αποχαιρετούμε αύριο. Δεν ξεχνάμε τις παλιές ε, γνωριμίες. Ε, τραγουδάμε εδώ αυτό το τραγούδι την παραμονή της χρονιάς ε, γιατί όπως λέει όπως λένε και τα λόγια, αποχαιρετούμε τον παλιό το χρόνο. Δεν χάνουμε τους παλιούς φίλους, κάνουμε νέους και παίρνουμε νέες αποφάσεις για το μέλλον. Τους επόμενους μήνες θα έχουμε έντονες διαπραγματεύσεις και θα κυριαρχήσουν σε μεγάλο βαθμό στο πρόγραμμα της Κομισιόν. Δυστυχώς αυτή είναι η τελευταία φορά που μιλάω εδώ μέσα και σας αποχαιρετώ όλους. Όμως Όσο και αν διαφωνήσαμε, δεν κρατάω κακία σε κανέναν. Θα μπορούσα να πω τόσα πολλά, αλλά υπάρχει τόσο λίγος χρόνος. Οπότε θα αναφέρω μόνο το εξής. Ζητώ στο πνεύμα της συνεργασίας ένα απλό πράγμα από την Κομισιόν και την Βρετανική κυβέρνηση, κάτι το οποίο έχει ιδιαίτερη σημασία μην χρησιμοποιήσετε τους ψαράδες του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως αντικείμενο διαπραγμάτευσης ή τους πολλούς ανθρώπους που απασχολούνται στην επεξεργασία των ψαριών. Μην ξεπουλήσετε τους ψαράδες. Έχουν τραβήξει τόσα πολλά τα τελευταία 40 χρόνια. Μην τους υποβάλλετε σε άλλη δοκιμασία. Οπότε αποχαιρετούμε την Πολιτική Ένωση και καλωσορίζουμε την Νέα Βρετανία. Και πάντα θα είμαστε σύμμαχοι των Ευρωπαίων γειτόνων μας. Ελπίζω η νέα μας σχέση να είναι όλα όσα θα πρέπει να είναι. Ελπίζω λοιπόν να έχουμε αρμονικές σχέσεις. Γεια σας. Ευχαριστώ. Σας έδωσα λίγο χρόνο παραπάνω αφού ήταν η τελευταία σας παρέμβαση, κάποια στιγμή πρέπει να τελειώσει. Μονσεράτ, για ένα μισή λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συζητάμε το πρόγραμμα εργασίας Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2020 και το οποίο στηρίζουμε. Χτες όμως έγινε πραγματικότητα το Brexit και πρέπει να μάθουμε από τα σφάλματά μας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι για την ειρήνη, για την πρόοδο. Όμω ο ευρωσκεπτικισμό, ο λαϊκισμός δυσκολεύει το ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Έχουμε πετύχει πολλά μέχρι τώρα. Δεν πρέπει να δούμε το μέλλον μας μόνο νομοθετικό. Πρέπει να φροντίσουμε για το κράτος δικαίου, για τις αξίες της Ένωσης, για την ελευθερία, την ισότητα, την οικονομική και κοινωνική πρόοδο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι θεματοφύλακα των συνθήκων για όλα τα κεκτημένα και πρέπει να υποχρεώνονται όλες οι χώρες μέλη για όσα αποφασίζουμε. Το 2017 εγκρίθηκε ένα καθεστώς κυρώσεων για ορισμένες ε, χώρες και σε σχέση με την Βενεζουέλα. Επίσης το 2018 συμπεριέλαβε και την κυρία Ντέλση Ροντρίγκες που είναι αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Μαδούρου και της απαγόρευσε την είσοδο. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι παραβίασαν και επέτρεψαν στην κυρία αυτή να βρεθεί σε ισπανικό χώρο, στο χώρο του Σέγγεν. Ζητούμε λοιπόν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συγκεντρώσει πληροφορίε και να ζητήσει από τον κύριο Σάντσε να τηρήσει τι αποφάσει του Συμβουλίου. Γιατί δεν μπορούμε να δεχτούμε ότι μια ευρωπαϊκή κυβέρνηση δεν τηρεί το ευρωπαϊκό δίκαιο γιατί τότε απομακρυνόμαστε από τους Ευρωπαίους. Όλοι μαζί πρέπει να προχωρήσουμε προς το μέλλον στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστούμε κυρία Ντάλη. Ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, στις εκλογές αλλά και τους τελευταίους μήνες εμείς σοσιαλδημοκράτες ξεκαθαρίσαμε ότι στην περίοδο αυτή θέλουμε αλλαγές κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές. Και ακριβώς ε, φέτος πρέπει να αρχίσουμε να δουλεύουμε για την αλλαγή αυτή, για την οποία τόσο πολύ μιλάμε και στην οποία πιστεύουμε. Και δεν πρόκειται για ένα όνειρο μόνο αυτή η αλλαγή. Πρέπει να είναι μια αλλαγή που θα γίνει πραγματικότητα. Οι πολιτικέ αποφάσει που θα ληφθούν φέτο θα δείξουν τον δρόμο για τι οικονομίε που θέλουμε για τι χώρε μα και θα μα καθοδηγήσουν στις τεχνολογίες πάνω στις οποίες πρέπει να επενδύσουμε. Όμως οι χώρες ε, μέλη πρέπει να υλοποιήσουν αυτά τα μέτρα, να τα εφαρμόσουν και τις νέες αυτές πολιτικές. Οπότε πρέπει να επικεντρωθούμε σε καθαρές ε, βιομηχανίες, σε κινητικότητα, σε πιο καθαρή κινητικότητα, τόσο στον αέρα όσο και ε, χερσαίος και να απομακρυνθούμε από τα ορυκτά καύσινα. Αλλά για όλα αυτά χρειάζονται χρήματα. Πρέπει να βοηθήσουμε τους εργαζόμενους, στις περιφέρειες, ε, της χώρες για να μπορέσουν να κάνουν την αλλαγή αυτή. Αυτό είναι το μέλλον όμως. Αυτή είναι η απόφαση που πρέπει να πάρουμε για τις χώρες που εκπροσωπούμε και για τις οικογένειές μας βεβαίως επίσης. Ευχαριστώ Μιχαήλο για λεπτό. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε να εκφράσω πρώτα απ' όλα την υποστήριξή μου για το κύριο μήνυμά σας. Μετάβαση. Για μια μετάβαση η οποία προσφέρει ευκαιρίες για κάθε πολίτη, για κάθε κράτος μέλος. Ευκαιρίες για να έχουμε μια δίκαιη Ευρώπη κλιματικά ουδέτερη που θα βασίζεται στο κράτος δικαίου, την ε, έφτακτη μετανάστευση και τις εμπορικές συμφωνίες. Οι Ευρωπαίοι θέλουν να δουν συγκεκριμένη δράση από εμάς. Η συνεργασία αυτή είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Πρέπει να συνεργαστούμε για να υλοποιήσουμε αυτό το πρόγραμμα εργασία. Πρέπει να προσφέρουμε στους Ευρωπαίους πολίτες μια μετάβαση η οποία θα αυξήσει την ανταγωνιστικότητά μας και θα βελτιώσει τον τρόπο ζωής. Ευχαριστώ. shooter, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε, Κύριε Επίτροπε, ευχαριστώ για την παρουσίασή σας. Αναλυτικό το πρόγραμμα σας. Εγώ θα αναφερθώ μόνο στο θέμα τη ψηφιοποίηση. Οι δουλειέ ε, υψηλή εξειδικεύση προσφέρονται μόνο σε άντρε ή έγχρωμοι άνθρωποι οι οποίοι λαμβάνουν λιγότερε υπηρεσίε. Αυτά θα έχουμε εάν δεν παρέμβουμε στην αυτόματη λήψη αποφάσεων. Γι' αυτό χρειάζονται σαφεί κανόνε για την τεχνητή νοημοσύνη. Το ίδιο ισχύει και για τους ψηφιακούς ενδιάμεσους. Δυστυχώς το πρόσφατο παρελθόν είχαν πολλά παραδείγματα αναρτήσεων μίσους ή τρομοκρατίας ή περιεχόμενο το οποίο κατέβηκε αδίκως ή δεν μπόρεσε να ανέβει καν. Και βεβαίως πρέπει να διατηρήσουμε την ελευθερία λόγου. Οι ιδιωτικέ εταιρείε ή τα αυτόματα φίλτρα δεν μπορούν ποτέ να υποκαταστήσουν τους ανθρώπους. Κύριε Επίτροπε, το να βρεθεί η σωστή ισορροπία μεταξύ της προστασίας ε, και της ελευθερίας ε, είναι κέρια σημασίας και βεβαίως αναμένουμε τις προτάσεις σας στον τομέα αυτών. Μπιτσότο για ένα λεπτό έχουμε να κάνουμε με μια Ευρώπη η οποία επιμένει, δεν θέλει να κάνει τίποτα, θέλει να τιμωρήσει την Ιταλία με τη συνενοχή της αριστερής της κυβέρνησης για την κρίση στη Λιβύη με τους κινδύνους για τον Ισλαμικό φονταμενταλισμό η Ευρώπη είναι απούσα και στον τομέα τον οικονομικό δυστυχώς ε, εξακολουθείτε να τιμωρείτε ε, τους Ιταλούς ε, οι οποίοι θα πληρώσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα επόμενα χρόνια 900 εκατομμύρια στην Ένωση και θα πάρουν μόνο 160. Ο Τζεντιλόνι, ο νέος επίτροπος, ποιους υπερασπίζεται, τους πολίτες της Ιταλίας, όχι. Η Ιταλία ποτέ δεν θα πεθάνει σκλάβα των Παρισίων, του Βερολίνου και των Βρυξελών. Ευχαριστώ πρόεδρε. Νομίζω ότι η, βασικές, η βασική πρόταση του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι το Green Deal. το, θυμίζει το μεγάλο άλμα στο μέλλον του Μαουτσετούγκο. Όλα συγχωρούνται και όλα επιτρέπονται. Θανατώσεις, υποχρεωτικές μετακινήσεις πληθυσμών, διακανονισμοί, έλεγχοι συμπεριφορών Ολόκληρες ε, περιοχές λοιπόν της Ευρωπαϊκής Ένωσης κινδυνεύουν ε, νομίζω ότι θα πρέπει να δώσουμε στην προσπάθεια ε, επιπλέον 270 εκατομμύρια το χρόνο και αυτό για εντελώς ιδεολογικές ε, αιτιολογίες. Νομίζω ότι κινδυνεύει η Ευρώπη, στην ουσία η ιδεολογία λειτουργεί ιδεολειπτικά και εις βάρος των ελευθεριών των Ευρωπαίων. Ευχαριστώ. κύριος Γιόγκιση για ένα μισή λεπτό. Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, είδα την υλοποίηση της, του κοινωνικού πυλώνα στην, ε, στο πρόγραμμα εργασίας σας και ότι αυτό αποτελεί προτεραιότητα. Τώρα υπάρχει όλο και μεγαλύτερη ανησυχία στις χώρες μέλη της περιφέρειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι τα ωφέλη από την εσωτερική αγορά είναι άνισα και ότι οι κανόνες, οι ενιαίες στην εσωτερική αγορά ε, το μόνο αποτέλεσμα που έχουν είναι φτηνό εργατικό δυναμικό. Συνεπώς, η εσωτερική αγορά κινδυνεύει γιατί οι κοινωνικές εντάσεις το μόνο που θα κάνουν είναι ότι θα αυξηθούν αν δεν αντιμετωπίσετε τις προκλήσεις και θα γίνει ακόμα χειρότερη η κατάσταση με την ψηφιοποίηση που εντοπίζετε εσείς σαν μία από τις μεγάλες τάσεις της εποχής μας. Η λύση είναι να μην υπάρχουν ανισότητες στις αμοιβέ και ούτε διαφορές στις αμοιβέ ανάλογα με το σε ποια χώρα βρίσκεται κανείς. Και η πολιτική συνοχής πρέπει να βασίζεται στην ελεγγύη μεταξύ των χωρών μελών. Αν δεν τα καταφέρετε, τότε ο αντιγωνισμός θα καταλήξει σε λαϊκισμό κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέσα από πραγματικό κοινωνικό διάλογο λέτε ότι προσπαθούμε να ενισχύσουμε την κοινωνία των πολιτών για να βρεθούν λύσεις και να δίνουν και εκείνοι λύσει. Αυτό είναι σωστό, αλλά ε, μία σύσταση. Κοιτάξτε λίγο τι γίνεται και στην περιφέρεια και στις κοινότητες της περιφέρειας και στις αρχές εκεί που πρέπει και αυτές να δίνουν τη γνώμη τους γιατί είναι αυτοί που βρίσκονται πιο κοντά στους πολίτες. Υπάρχει μπλε κάρτα από τον συνάδελφο Σφαμπ. Τη δέχεστε? Δέχεστε την μπλε κάρτα? Δέχεστε μπλε κάρτα, ναι. Ωραία. 30 δευτερόλεπτα παρακαλώ κύριε Σβάπ. Αγαπητέ συνάδελφε, πιστεύω ότι συμφωνούμε στον αγώνα κατά του λαϊκισμού. Ε, λέτε ότι οι άνθρωποι στην περιφέρειά σας ε, βλέπουν ότι τους εκμεταλλεύονται. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει προσφέρει στους ανθρώπους στην περιφέρεια τεράστια ευκαιρία να κερδίσουν περισσότερα και ε, ίσως ε, άνθρωποι σε άλλα κράτη-μέλη έχουν την τελείως αντίστροφη άποψη. Πώς θεωρείτε ότι θα μπορέσουμε να κάνουμε τη σωστή επιλογή και να βρούμε την σωστή ισορροπία. 30 δευτερόλεπτα για να απαντήσετε. Ευχαριστώ για την ερώτησή σας. Ε, σωστό είναι αυτό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ένα μέσο το οποίο υπάρχει για να γεφυρώσει τις διαφορές μεταξύ των κρατών μελών. Λέγεται πολιτική συνοχή. Το πρόβλημα είναι ότι η πολιτική συνοχή είναι αντικείμενο κατάχρηση. Πολλά από τα κονδύλια της συνοχή πάνε είτε σε διάβλους διαφθοράς, είτε σε έργα τα οποία δεν βοηθούν την ανταγωνιστικότητα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μια σημαντική ευθύνη να επιβλέπει την διαχείριση των κονδυλίων της συνοχής, να πηγαίνουν σε έρευνα και ανάπτυξη και σε εκπαίδευση για να βελτιώνουν την χρήση αυτών των κονδυλίων για να βελτιωθεί η οικονομία των κρατών μελών. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ. Τον λόγο έχει τώρα ο κύριο Μέλο για ένα μισή λεπτό. E- ευχαριστώ. Τα σχέδια διασυνδεσιμότητας ανάμεσα στην Πορτογαλία, την Ισπανία και τη Γαλλία επιτρέπει να μεταφέρει φυσικό αέριο Πορτογαλία προ την Ευρώπη. Και αυτό είναι μία από τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το υποστηρίζει η Επιτροπή και το θεωρεί έργο κοινού ενδιαφέροντος για να διασφαλιστεί η ασφάλεια ε, προμήθειας και φοδιασμού στην Ευρώπη, να μην εξαρτώμαστε από την Ρωσία για το φυσικό αέριο, για παράδειγμα. Το σχέδιο αυτό όμως αντιβαίνει με τα ενεργειακά συμφέροντα τελικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μια που δεν θεωρείται καθαρό. Οπότε θέλω να μάθω περισσότερα. Και όσον αφορά το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο, ξέρω ότι γίνονται δύσκολες διαπραγματεύσεις εξαιτία του Brexit και χρειάζονται πολιτικές αποφάσεις ώστε να ξέρουμε τι θα γίνει το 2021. Πρέπει να υπάρχει ένα ε, σχέδιο για έκτακτες περιπτώσεις που να μας προστατεύσει την επόμενη δεκαετία. Οπότε μίλησα για την μείωση εξάρτησης από τη Ρωσία για την ενεργειακή μας προμήθεια, κάτι το οποίο θα μπορούσε να βοηθηθεί κατά πολύ από την προμήθεια φυσικού αερίου από την Πορτογαλία. Θα ήθελα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν να μου εξηγήσει τι συμβαίνει για αυτά τα δύο, κυρίως για την περίπτωση φυσικού αερίου που δεν καταλαβαίνω Ευχαριστώ. Φριτσόν για ένα λεπτό. Ε, en framtid som eh, Κοιτάξτε, μιλάτε για προετοιμασία για το μέλλον. Ένα μέλλον το οποίο θα χαρακτηριστεί από ψηφιοποίηση, παγκοσμιοποίηση, τις κλιματικές ε, προκλήσεις. Έχουμε λοιπόν ένα πρόγραμμα εργασίας ε, το οποίο προβλέπει μια πιο ισχυρή Ευρώπη, κοινωνική Ευρώπη. Πρέπει λοιπόν να δούμε τα θέματα των κοινωνικών δικαιωμάτων και τις εγγύσεις ε, των παιδιών, αλλά βεβαίως υπάρχουν πράγματα που λείπουν από την πρωτοβουλία αυτή. Χρειαζόμαστε μια αναδιατύπωση ε, των δυνατοτήτων απασχόλησης των γυναικών, ένα καλύτερο εργασιακό περιβάλλον και να ενισχύσουμε τον κοινωνικό διάλογο. Οι συμπολίτε μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση θέλουν αποτελέσματα. Αυτό πρέπει να κάνουμε για να ξεκινήσουμε από τώρα. Σας ευχαριστώ. Αγία για ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε. Ε, προσπαθείτε να καλύψετε τις ανάγκες οι οποίες υπάρχουν και σας συγχαίρουμε γι' αυτό. Τώρα σχετικά με ένα σημαντικό θέμα, το δικαίωμα πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Για να το ασκήσουμε αυτό πρέπει να γνωρίζουμε, πρέπει να είμαστε ενημερωμένοι. Όμως βλέπω ότι μερικές φορές οι πληροφορίες έρχονται με πάρα πολύ μεγάλη καθυστέρηση. Ένα πρώτο παράδειγμα το σύστημα μπακ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δηλαδή όλες οι δαπάνες για τα ευρωπαϊκά προγράμματα δεν είναι διαθέσιμο, ενώ είμαστε αρχή επί του προϋπολογισμού. Και ένα πιο πολιτικό παράδειγμα είναι η διάδοση στον τύπο πριν μερικούς μήνες για τα κέρδη της εσωτερικής αγοράς για κάθε κράτος μέλος, που δείχνουν τα θετικά στοιχεία για κάθε χώρα μέλος στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων για το επόμενο πολιετές πρόγραμμα όλα αυτά έχουν μεγάλη σημασία. Κύριε Επίτροπε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι εταίρο σας και γι' αυτό θα πρέπει να μας δώσετε εγγυήσει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μας δίδει όλα τα στοιχεία τα οποία χρειαζόμαστε. Από την κυρία Γκραπίνη Μπλε Κάρτα. Ευχαριστώ Πρόεδρε που δεχθήκατε την ερώτησή μου. Το θέμα είναι η διαφάνεια η οποία θα πρέπει να υπάρχει ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Κοινοβούλιο. Ένα παράδειγμα. Όταν συζητούσαμε για τη διπλής χρήση, ή διτής χρήσης προϊόντα Υποτίθεται ότι ε, προτίμασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μια έκθεση από εμπειρογνώμονες συντεταγμένοι η οποία ε, όμως ε, στην ουσία δεν μας δόθηκε τα βασικά χαρακτηριστικά μας δόθηκαν τα υπόλοιπα παρέμειναν απόρριτα νομίζω ότι κάτι τέτοιο δεν είναι σωστό ε, χρηματοδοτεί ε, κάποιες έρευνες με ευρωπαϊκά χρήματα και μετά δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τι ακριβώς έχουμε παραγγείλει για έρευνα. Θέλετε να δώσετε μια απάντηση. Κοιτάξτε, απλά σημειώνω αυτό το οποίο είπατε, δεν έχω να κάνω κάποιο σχόλιο. Ο κύριος Γιγόλτ, ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κύριε Αντιπρόεδρε Σεύκοβιτς. Το πρόγραμμα εργασίας της Κομισιόν επί της αρχής ε, έχει τη σωστή έμβαση. Η προστασία του κλίματος, οικολογική κρίση, ε, νέα ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, κτλ. Σωστά αυτά. Αλλά ταυτόχρονα το πρόγραμμα έχει μια αδυναμία. Είναι πολύ γενικό και δύναμο όταν μιλάμε για την προστασία του κράτους δικαίου. Πολλοί πολίτες έχουν χάσει σεβασμό στα λόγια μας όταν λέμε ότι η Ευρώπη είναι μια κοινότητα αξιών όταν τα κράτη-μέλη παρασιάζουν θεμελιώδη δικαιώματα όπως την ελευθερία των ΜΜΕ καταπολέμηση της δημοκρατίας δεν μπορεί λοιπόν να τα αφήσει έτσι η Κομισιόν. Δεν έχει νόημα να φτιάχνουμε λίστες, χρειάζεται εφαρμογή και κυρώσεις που δεν υπάρχουν στο πρόγραμμά σας. Αναμένουμε λοιπόν να λάβετε σκληρά μέτρα. Αλλιώς οι πολίτες χάνουν το σεβασμό για την θαυμάσια Ευρωπαϊκή μας Ένωση. Σας ευχαριστώ Ράιλ για ένα λεπτό. Και πάλι σήμερα μιλάμε για τον πυλώνα των κοινωνικών δικαιωμάτων και μιλάμε για ευρωπαϊκό επίδομα ανεργίας. Δηλαδή πάλι μιλάμε για μια ένωση μεταβάσεων. Αυτό δεν είναι κοινωνική δικαιοσύνη, αντιθέτως. Είναι αντικοινωνική. Ανταμείβει τα κράτη που έκαναν λάθη στο παρελθόν και τιμωρεί αυτά που έκαναν κάτι σωστό. Να σας δώσω το παράδειγμα της Γερμανίας. Είμαστε η μεγαλύτερη οικονομία τη Ευρωπαϊκή Ένωση και ο μεγαλύτερο καθαρό εισφορέα. Τι γίνεται όμω με την κοινωνική δικαιοσύνη. Οι καθαροί μισθοί τη Γερμανία έχουν πέσει κατά 10% από όταν μπήκε το ευρώ. Η μόνη χώρα στην οποία συνέβη αυτό. Η φτώχεια των λυκειωμένων έχει διπλασιαστεί. Οι Γερμανοί μένουν στο δρόμο, δεν μπορούν να πληρώσουν τον νίκη. Γιατί πιέζονται όλο και περισσότεροι άνθρωποι στους χαμηλόμισθους ενώ ταυτόχρονα έχουν ανέβει τα νίκια κατά 50% έτσι πάνε τα πράγματα στην πλούσια Γερμανία λοιπόν η κοινωνική δικαιοσύνη πρέπει να παραμείνει εθνική υπόθεση ευχαριστώ ευχαριστώ Τόμασιτς για ένα λεπτό Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε η παρουσίαση του νέου προγράμματος εργασίας είναι μεγάλα λόγια, δίκαια ε, μετάβαση, πράσινη οικονομία, οικονομία ε, στην υπηρεσία των πολιτών κλπ. κλπ. Πολύ φιλόδοξη η πράσινη συμφωνία, όλοι το λένε, αλλά ε, κανείς δεν λέει πόσο θα κοστίσει στους Ευρωπαίους πολίτες κατά πόσο είναι προς το συμφέρον των πολιτών. Αυτό που χρειάζονται οι πολίτες είναι δουλειές και η ευρωπαϊκή οικονομία μέχρι τώρα αυτό φρόντιζε για τους πολίτες. Τα άλλα ακούγονται ρομαντικά και από πίσω κρύβουν πολύ γραφειοκρατία από τις Βρυξέλλες που θα επιβάλλει πράγματα στις χώρες μέλη. Ο τρόπος ζωής μας θα, θα έπρεπε να είναι αυτό που θέλουν οι ευρωπαϊκοί λαοί και όχι αυτό που επιβάλλουν οι Βρυξέλλες. Ευχαριστούμε Στέφανετς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Η νέα Κομισιόν ε, έχει θέσει πολύ φιλόδοξους στόχους, εγώ όμως θα ήθελα να επισημάνω κάτι συγκεκριμένο. Μιλάμε για το ότι τα κοινά εργαλεία ελέγχου θα έχουν περισσότερες δυνατότητες ε, για να περιορίσουν την δύναμη των ολιγαρχών που δολοφόνησαν δύο ανθρώπους στην ε, Σλοβακία, τον δημοσιογράφο και την ε, αραβωνιαστικιά του. Πριν από αυτούς είχε δολοφονηθεί η κυρία Γκαρουάνα Γκαλίτσια στη Μάλτα γιατί αποκάλυψε την εγκληματική διαπλοκή. Πολλά από αυτά τα κλεμμένα λεφτά είναι από ευρωπαϊκά κονδύλια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν που τα μοιράζει έχει υποχρέωση να ελέγχει το πώς χρησιμοποιούνται και θα χαιρόμουν αν στο τέλος του 2020 έχει επιτευχθεί σαφής πρόοδο στην προστασία των οικονομικών συμφερόντων της κοινότητας. Η Κομισιόν έχει σε αυτό την στήριξή μου. Σας ευχαριστώ, Αντριέ. Ευχαριστώ, Επίτροπε. Θέλουμε να γίνουμε η πρώτη Ήπειρος χωρίς άνθρακα μέσα σε κάποια χρόνια και θέλουμε να είμαστε καινοτόμοι και σε σχέση με την προστασία του περιβάλλοντος. Θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας τρεις ανησυχίες. Πρώτον, προϋπολογισμός το ελεγκτικό συνέδριο θεωρεί ότι έχουμε ανάγκη από 100 εκατομμύρια τον χρόνο ε, για την πράσινη μετάβαση, ενώ η Επιτροπή πιστεύει ότι χρειάζεται το ποσό αυτό για 10 χρόνια. Δεύτερο θέμα είναι το θέμα της ε, συνοχής, σύγκλησης μάλλον. Δίνουμε μάχη για την ε, ανανέωση στον τομέα της ενέργειας και από την άλλη υπογράφουμε συμφωνίες απαράδεκτες. Το να κουβαλάμε κρέας από 10.000 χιλιόμετρα μακριά είναι μια περιβαλλοντική ύβρις και επίσης το κοινωνικό θέμα. Η οικολογία και η κοινωνία συνδέονται μέσω ακριβώς της αλλαγής του οικονομικού μοντέλου. Και όμως το κοινωνικό θέμα δεν περιλαμβάνεται στις προτάσεις σας, κάτι το οποίο δεν μπορούμε να αποδεχτούμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ε, πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Αντιπρόεδρε, ευχαριστώ για αυτό το πρόγραμμα εργασίας και για τη σημασία που δίνεται στην ψηφιακή μετάβαση στην Ευρώπη. Πράγματι, χρειαζόμαστε φιλόδοξες ψηφιακές πολιτικές ώστε οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να αναπτυχθούν και να προχωρήσουν σε καινοτομίες στην Ευρώπη, αλλά και προκειμένου οι Ευρωπαίοι να μπορέσουν να αποφεληθούν από την ψηφιακή μετάβαση πρέπει τώρα να προχωρήσουμε για να προλάβουμε άλλους παίκτες. Εμείς είμαστε αυτοί που θα θέσουμε τις προδιαγραφές παγκοσμίω. Για την πράξη αυτή ψηφιακή χαίρομαι για το όσο αναφέρονται όσον αφορά τα δεδομένα, όσον αναφέρονται για την ασφάλεια στο κυβερνοχώρο, για την τεχνητή νοημοσύνη κλπ. Πρέπει να αποφασίσουμε πώς θα ρυθμίσουμε όμως τον ψηφιακό κόσμο. Αυτό είναι η προτεραιότητα. Σίγουρα θα είναι κάτι που θα κυριαρχεί όχι μόνο ε, στην ατζέντα του 2020 αλλά και για πολλά χρόνια μετά. Πρέπει να ξεκινήσουμε όμως τώρα και θυμηθείτε η απάντηση στα προβλήματά μας δεν είναι πάντα περισσότερη ρύθμιση αλλά καλύτερη ρύθμιση. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Η κυρία Ντελή τώρα. Ένα λεπτό παρακαλώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε Αντιπρόεδρε, όπως υπενθύμησα και χτες εδώ σε αυτό το εμικύκλιο και πολλές φορές μέχρι τώρα το κλίμα επήγει. Και δεν επήγει για το 2025, για το 2030. Όχι. Η δράση για την ε, κλιματική αλλαγή τώρα επήγει. Δεν θα σώσουμε τον πλανήτη με ένα κατάλογο ε, ωραίων ε, λόγων και επιθυμιών. Δεν μπορούμε να περιμένουμε ένα χρόνο παραπάνω. Τώρα πρέπει να ξεκινήσουμε με δυνατά μέτρα και κυρίως στον τομέα των μεταφορών που είναι υπεύθυνο για το 30% των εκπομπών ε, ρίων του θερμοκηπίου. Και γι' αυτό λοιπόν, κύριε Αντιπρόεδρε, θα ήθελα να κλείσει ο φάκελος πια όσον αφορά ε, τους φόρους που πρέπει να πληρώνουν ε, τα φορτηγά. Και επίσης να ξέρετε ότι ναι, συμφωνούμε με την αρχή ο Ριπένο να πληρώνει το, εμείς. Το Συμβούλιο όμως δεν μπορεί να συμφωνήσει και άλλαξε το κείμενο και είναι απαράδεκτο. Οπότε εμείς ζητάμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να έρθει με νέα δυνατή πρόταση ώστε να μπορέσουμε να έχουμε αυτές τις εισφορές από τα φορτηγά στο ύψος που πρέπει. Ευχαριστούμε. Νταρέ, ένα λεπτό παρακαλώ. Το 2020 είναι μια κρίσιμη χρονιά για την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει να αντιμετωπίσει πολλά θέματα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Brexit, το προπολογισμό από το 2021 μέχρι το 2027. Ε, είναι απαραίτητο λοιπόν να φανούμε πολύ προσεκτικοί έτσι ώστε κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων να μην αγνοηθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις όπως επίσης και τα εξαίρετα προϊόντα μας με ονομασίες προέλευσης. Επίσης υποτίθεται ότι θα αυξήσετε ακόμα περισσότερο το πρόγραμμα Εράσμους. Προτείνει ε, τον διπλασιασμό η κυρία Φάντερ Λάιεν. Ξέρει τι σημαίνει αυτό οικονομικά Εύκολα είναι να τα λες αυτά, αλλά δύσκολα να τα κάνεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είπατε ότι θα είναι μια επιτροπή με γεωπολιτική αντίληψη. Αυτό έχει ανάγκη η Ευρώπη. Το θέμα είναι τα λόγια να τα κάνουμε πράξη. Ποια είναι τα μέτρα τα οποία θα υιοθετήσετε. Υπάρχει ας πούμε το North Stream που διαιρεί την Ευρώπη και αυξάνει την πίεση της ε, Ρωσίας στην Ήπειρό μας. Παρ' όλα αυτά έχουμε ανάγκη το φυσικό αέριο. Θα πρέπει επίσης ε, η Νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δουλέψει ε, σεβόμενη αυτά τα οποία ήσαν οι αξίες μας. Θέλουμε να είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά μια ένωση η οποία να σέβεται τα κράτη-μέλη και να μην επιβάλλει τίποτα στα κράτη-μέλη. Γιατί ανακατεύεστε στα εσωτερικά των κρατών μελών, γιατί ανακατεύεστε με θέματα τα οποία είναι αποκλειστική τους αρμοδιότητα και επειδή συνδέεται αυτές τις πολιτικές συμπεριφορές με τον προϋπολογισμό. Αυτό θα μας οδηγήσει σε περισσότερες διαιρέσεις. Γκλάβακ. Κυρία Γκλάβακ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχουν περάσει δεκαετίες από τις συνθήκες της ε, Ρώμης και ο κόσμος είναι πολύ πιο ασταθής ε, κλιματική κρίση, μεταναστευτικό, αλλάζουν τον τρόπο ζωή μας. Πρέπει, κύριε Επίτροπε, να εστιάσουμε στην ισότητα και ισότητα ευκαιριών για όλους. Άντρες, γυναίκες, ανατολικούς, δυτικούς, νέους, γέρους. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει 47 μέτρα κλειδί, και ένα δισεκατομμύριο ευρώ, χίλια εκατομμύρια ευρώ δηλαδή για το κλίμα και το περιβάλλον. Το συμφέρον των πολιτών είναι ε, η ίση αμοιβή για ίση εργασία, αναφέρεται και στη στρατηγική για την ισότητα των φύλων. Αυτό θα είναι τεράστια πρόκληση. Οι γυναίκε βγάζουν 16% ε, τις 100 λιγότερα από του άντρε, αν και κατά μέσο είναι πιο μορφωμένε. Νέα θέματα για την Ευρωπαϊκή Δημοκρατία. Εδώ πρέπει να περιλάβουμε τους νέους πολίτες, κοινωνία των πολιτών, ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα ως ε, συμμετέχοντες σε αυτή τη συζήτηση. Ποιο μπορεί να μιλήσει για την δημοκρατία καλύτερα από μια ήπειρο που την ε, επινόησε. Πρέπει να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη λοιπόν στο ποιοι είμαστε και στο πού πηγαίνουμε. Το πρόγραμμα αυτό είναι ένας καλός τρόπος να το πετύχουμε. Ευχαριστώ. Πίτσουλα. Για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ. Πρόεδρε, κύριε Χαίρομαι για την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά πρέπει να δούμε και πόσο θα κοστίσει η μετάβαση αυτή για μια πιο οικολογική και βιώσιμη Ευρώπη. Υπάρχουν πολλές περιφερειακές κοινότητες που θα πρέπει να συμπεριληφθούν στη διαδικασία ε, και κυρίως να ληφθούν υπόψη για το Ταμείο της Δίκαιας Μετάβασης. Είναι αναγκαίο και για την Κροατία που είναι μια χώρα που έχει ανάγκη τους πόρους αυτούς. Χαίρομαι πάντως για τη στρατηγική. Ο προσανατολισμός επίσης για τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης που περιλαμβάνονται στην Πράσινη Συμφωνία είναι και αυτό κάτι πολύ σημαντικό για τους πολίτες και χαιρόμαστε που επίσης αναφέρεται και στην εγγύηση των ε, νέων και των ε, παιδιών ο Επίτροπος. Ο γεωστρατηγικός τώρα ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι και αυτό που χρειάζεται και καλό θα ήταν να ξεκινήσουμε διαπραγματεύσεις με την Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία και κυρίως πριν από τη διάσκεψη στο Ζάγκρεπ, μια που ετοιμάζονται τώρα, γίνονται οι προετοιμασίες. Ο κύριος Γκαρκάνο. Είναι η τελευταία μέρα που έχουμε το Ηνωμένο Βασίλειο εδώ μαζί μα και τι αρνητικέ συνέπειε θα τι δούμε μέσα στι επόμενε εβδομάδε, τόσο για εμά όσο και για αυτού. Ένα θέλω να αναφέρω που με ανησυχεί ιδιαίτερα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια υπερδύναμη με το Ηνωμένο Βασίλειο εντό. Εκτό η Ευρώπη καθίσταται πιο αδύναμη το Imperial College, το Cambridge, η Oxford, όλα αυτά τα πανεπιστήμια είναι πανεπιστήμια τα οποία βρίσκονται στην ε, πρώτη γραμμή στην Ευρώπη. Δείτε τα 50 καλύτερα πανεπιστήμια της Ευρώπης, 12 από αυτά είναι στην Ασία, 21 στις Ηνωμένες Πολιτείες, 11 στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ελβετία και ένα από τα 50 καλύτερα βρίσκεται στην ε, υπόλοιπη Ευρώπη. Αυτό είναι κάτι πολύ σοβαρό. Μιλάμε για την καινοτομία, μιλάμε για την κοινωνία τη γνώση, αλλά δεν επενδύουμε στα πανεπιστήμια μας. Και το πρόγραμμα εργασία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν αναφέρεται καν ε, στα πανεπιστήμια. Έχουμε προβλήματα κινητικότητα και άλλα. Ε, λοιπόν, αυτό πρέπει να κάνει η Ευρώπη. Θα πρέπει να γίνουμε μια υπερδύναμη στον τομέα τη εκπαίδευση. Ευχαριστούμε. Στρίκ. Ένα λεπτό. Ε, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Το πρόγραμμα εργασίας ε, δεν έχει αποφασίσει ακόμα για το κοινό σύστημα ασύλου γιατί ε, σχεδιάζονται τα νέα σύμφωνα για το άσυλο που έχει ήδη ανακοινώσει η Πρόεδρος. Πρέπει να βρεθεί μια λύση για την κατανομή των ετούντων ασύλου και ζητώ από την Κομισιόν και τα κράτη-μέλη να βρουν μια λύση για να αναλάβει ο καθένα τις ευθύνε του και το βάρο που του αναλογεί. Αυτό απαιτεί άμεση κατανομή των ετούντων άσυλο απευθεία από τα εξωτερικά σύνορα. Πολλά κράτη-μέλη σκέφτονται και προτείνουν τώρα μια διαδικασία στα σύνορα, δηλαδή ότι θα γίνεται μια αξιολόγηση, έλεγχο. Εγώ θα σα παρακαλούσα να μην ακολουθήσετε αυτόν τον δρόμο, γιατί αυτό σημαίνει περισσότερα hot spot, μακροσκελείς διαδικασίες και κράτηση. Εγώ ήμουν υπέρ της πρότασης των πρασίνων. Ε, μια άμεση κατανομή και να αρχίσουμε να εφαρμόζουμε τους κανόνες που έχουμε. Η υποδοχή, ε, κατανομή, να έχουμε ένα αναρμονισμένο σύστημα και να μοιραζόμαστε την ευθύνη. Ευχαριστώ. Φεστ, θέλετε τον λόγο ή όχι, ξέρετε τους κανόνες. Λόγω έχει ο κύριος Φέστ. Ευχαριστώ. Η Αντιπρόεδρος ε, και η κυρία Μπάρλεϊ ε, δίνει τον λόγο στους βουλευτές μόνο εάν σταματήσουν να επιδεικνύουν την πίστη στην πατρίδα, της, στην πατρίδα τους. Ε, αγαπητέ συνάδελφε, ε, δεν θέλω να ξεκινήσουμε τώρα συζήτηση πάλι για αυτό το θέμα. Σας παρακαλώ λοιπόν να σέβεστε το αξίωμα της ε, προεδρεύουσα. Δεν είναι δική μου η απόφαση, είναι του Προεδρείου. Εάν θέλετε, σας παρακαλώ να παραπονεθείτε αρμοδίως δια της προβλεπόμενης οδού. Ε, νομίζω αρκεί. So, για δοκιμάστε τώρα. Δεν απευθύνομαι σε εσά λοιπόν, αλλά προ το Προεδρείο. Αλλά μιλάμε για μια Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία ε, χτες ήδη μιλούσε για τα δικαιώματα των αυτοχθών στον πολιτισμό τους, ε, την παράδοσή τους και τις σημαίες τους αλλά το αρνείται αυτό στους ευρωπαϊκούς λαούς. Οι Βρετανοί ευτυχώς εντωμεταξύ έβγαλαν τα συμπεράσματα που πρέπει και αποχώρησαν και είμαι σίγουρος ότι και άλλοι λαοί θα ακολουθήσουν το παράδειγμα αυτό και κάποια στιγμή και η Γερμανία. Και αυτό θα μας έδινε διπλή χαρά γιατί έτσι θα τελειώσει και η υποταγή της Γερμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και η δική σας η μικροπρεπής ε, διεύθυνση της συζήτησης. Λοιπόν, ε, ξεπεράστε και το χρόνο. Ε, κοιτάξτε, σας ξαναλέω τις πολλές ωραίες σημαίες εδώ από πίσω για τις οποίες είμαστε υπερήφανοι. Λοιπόν, βόντρα για ένα λεπτό. Yes, thank you very much. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Χτες είχαμε μια θλιβερή ημέρα που τέλειωσε και με ένα θλιβερό τραγούδι και εδώ ξεκινάμε με τις επιπτώσεις. Χάνουμε τα αγγλικά, τη λίγκουα φράγκα, ε, την κοινή κατανόηση. Η γλώσσα βρίσκεται στην καρδιά της κοινής κατανόησης και μπορούμε να χρησιμοποιούμε τη δυνατότητα με το Brexit, γιατί τώρα τελικά γίνονται τα αγγλικά μια γλώσσα που μπορούμε όλοι να αποδεχτούμε, οι Γερμανοί, οι Γάλλοι. Αντί να γίνεται αυτό όμω, γίνεται το αντίθετο. Καθένα μιλάει τη μητρική του γλώσσα με κάποιε μόνο εξαιρέσει και οι άλλοι δεν ακούνε καθόλου. Το πρόγραμμα εργασία λοιπόν τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι γεμάτο φιλοδοξίε, χωρί μελέτη αντικτύπου και χωρί τίποτα για την πρόθεση των αγγλικών ω lingua franca. Οπότε ρωτάω, ε, σκοπεύετε να κάνετε κάτι για να σταματήσει αυτό το σύνδρομο της Βαβέλ και να προωθήσετε την κοινή κατανόηση στην επικοινωνία μεταξύ μας. Ευχαριστούμε. Λάγκε. Ένα λεπτό παρακαλώ. Ναι, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Αντιπρόεδρε, Τύπωσα το πρόγραμμα εργασίας της ε, Κομισιόν και δεν ξέρω, ε, κοίταγα και λέω πως δεν τυπώθηκε κάτι. Γιατί για τις εξωτερικές οικονομικές σχέσεις βλέπω μόνο το σημείο 30, μεταρρύθμιση του ΠΟΕ. Κάποια στιγμή δηλαδή στο μέλλον μπορεί να γίνει, αλλά δεν υπάρχει τίποτα το οποίο να έχει σχέση με την εξωτερική διάσταση του Green Deal και την εφαρμογή των στόχων ε, του ΟΗΕ στην εξωτερική εμπορική πολιτική. Οπότε, ερωτώ την Κομισιόν, πού είναι αυτή η στόχη η αναπτυξιακή στην εξωτερική πολιτική, τι γίνεται με το Ταμείο Αντιστάθμισης στα σύνορα για να μην υπάρχει ανταγωνιστικό μειονέκτημα. Πού είναι οι αλυσίδες εφοδιασμού που θα είναι δίκαιες να αναλάβουν και οι εταιρείε παγκοσμίω τι ευθύνε του. Ε, εδώ πρέπει να κάνετε κάτι. Ε. Ευχαριστούμε. Το λόγο τώρα έχει ο κύριο Μπότος για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το πρόγραμμα εργασίας Ευρωπαϊκής Επιτροπής περιλαμβάνει διάφορες πρωτοβουλίες που έχουν να κάνουν με την υγεία και τα τρόφιμα. Η στρατηγική από το χωράφι στο πιάτο, για παράδειγμα, όπως και άλλα σχέδια. Και συμφωνώ με όλα αυτά. Αλλά προσοχή, κάτι λείπει. Λείπει μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία, η οποία θα μας ε, επέτρεπε να κάνουμε κάτι παραπάνω. Οι καταναλωτές να μπορούν να επιλέγουν γνωρίζοντας τι τρώνε και θα μπορούσαμε έτσι να αποφύγουμε ασθένειες. Όλοι οι Ευρωπαίοι, ανεξάρτητα από το επίπεδο εκπαίδευσή τους... πρέπει να έχουν σωστή και αποτελεσματική πληροφόρηση για τα τρόφιμα τα οποία καταναλώνουν. Επιμένω λοιπόν ότι είναι αναγκαίο να υπάρξει μια τέτοια πρωτοβουλία για τις ετικέτες, για τη σήμανση των προϊόντων που να λαμβάνει υπόψη και να περιλαμβάνει τη θρεπτική αξία και άλλα στοιχεία. Γιατί οι πολίτες ενδιαφέρονται και αυτό θα έπρεπε να περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα εργασίας μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ρόμπερτ Ρος. Τώρα για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία είναι η νέα μας στρατηγική ανάπτυξη σύμφωνα με το πρόγραμμα εργασία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2020. Όμως το μόνο που σημαίνει αυτό και το μόνο το οποίο είναι γνωστό μάλλον από αυτού είναι ότι θα στοιχήσει 11,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Τι περιλαμβάνει και τι σημαίνει για τους πολίτες και τι επιχειρήσει, αυτό παραμένει ασαφές. Στο μεταξύ, η Πράσινη Συμφωνία συμπεριλαμβάνεται στην νομοθεσία, κάτι το οποίο καταστά την διαδικασία χωρί επιστροφή. Και η ταξινόμηση των επενδύσεων επίση θα καταστήσει την οικονομία μα μια οικονομία η οποία θα κατευθύνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό είναι ένα βρωμικό παιχνίδι, γιατί ε, τελικά θα είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία θα αποφασίσει τι είναι καθαρό και τι δεν είναι καθαρό. Και θα καταλήξουμε σε περισσότερη γραφειοκρατία και σε μια κατάσταση κεντρικά σχεδιασμένης οικονομίας, κάτι το οποίο οι συνάδελφοί μας από την Ανατολική Ευρώπη απέρριψαν εδώ και 30 χρόνια. Περισσότερα χρήματα και περισσότερη εξουσία. Αυτό θέλει η Ευρώπη και δεν τη στάνουν. Και η δημοκρατία είναι ψηλά γράμματα για αυτήν. Με αυτή την πολιτική όμω θα ακολουθήσουν το παράδειγμα των Βρετανών και άλλε χώρε. Ευχαριστώ. Muito obrigado. Agora a palavra ao deputado um ο κύριος Μάρκες, ένα λεπτό. θα πρέπει ξεκινώντας να πούμε ότι οι βασικές μας προτεραιότητες ελήφθησαν υπόψη. Η πρόταση είναι μια καλή πρόταση. Είναι σημαντική η συζήτηση την οποία κάνουμε και το έγγραφο. Αλλά Τα λόγια τα είπαμε, το θέμα είναι τώρα να δράσουμε. Ε, πρέπει να είμαστε πρωτοπόροι στην απαλλαγή από τον άνθρακα και θα πρέπει επίσης να μην εγκαταλείψουμε κανέναν πίσω. Δεν μπορούμε να κερδίσουμε τον πόλεμο με τον άνθρακα με ένα στρατό ανέργων. θα πρέπει να είμαστε αλληλέγγυοι, θέλουμε μια οικονομία για τον λαό και πρέπει να ολοκληρώσουμε και την οικονομισματική και ε, ένωση αλλά αυτό όμως σημαίνει ότι τέλειωσαν τα λόγια και πρέπει να βρούμε το χρήμα και έτσι θα συμφωνήσουμε για το πολιετές δημοσιονομικό. Ευχαριστούμε. Το λόγο τώρα έχει ο συνάδελφος Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Κύριε Σεύκοβιτς, η Επιτροπή εμφανίζεται ως μια γεωπολιτική επιτροπή. Αλλά με τα πρώτα γεωπολιτικά γεγονότα στο Ιράκ σιωπήσατε. Και όταν είχαμε την απειλή για τιμωρητικού δασμού από τον Ντόναλτ Τραμπ για τους φόρους στα ψηφιακά, πάλι σιωπήσατε. Οι πολίτες μας έχουν μεγάλες προσδοκίες για το κλίμα, την κοινωνική δικαιοσύνη, την τίμια οικονομία, όμως όποτε χρειάζεται να τα υπερασπιστείτε, σιωπάτε. Τα σχέδιά σας είναι φιλόδοξα, αλλά θα οδηγήσουν σε διενέξεις με τις Ηνωμένε Πολιτείες, με την Κίνα, με τις ευρωπαϊκές χώρες μέλη, ή για παράδειγμα όταν πρόκειται για την αντασφάλιση, για την ανεργία ή για τον προπολογισμό. Σε καθένα από αυτά τα σημεία εμείς θέλουμε να είμαστε μαζί σας, εφόσον τολμήσετε όμως να τα προχωρήσετε. Η Ευρώπη είναι μια έχει μια κοινωνική οικονομία της αγοράς πιο ελεύθερη από την Κίνα και το κομματικό της κράτος ή από τα καπιταλιστικά κατέλ της Αμερικής. Εμείς θέλουμε να αγωνιστούμε για περισσότερη ειλικρίνεια και για περισσότερη βιωσιμότητα στην Ευρώπη. Οπότε μια γεωπολιτική επιτροπή ναι, αλλά να είναι και δυνατή, με μυϊκή δύναμη. Ευχαριστούμε. Ξεκινάει η διαδικασία τώρα Κάτσε τη Υπάρχουν διάφοροι που έχουν γραφτεί. Θα πρέπει να περιοριστούμε στο χρόνο μας. Οπότε ένα λεπτό ο καθένας, παρακαλώ, για να μπορέσουμε να δώσουμε το λόγο σε όσο γίνεται περισσότερους. Πρώτος, η Μαρία Γκραπίνη. Ένα λεπτό, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Επίτροπε, είναι σαφές ότι τα όσα μας παρουσιάσατε είναι ένα πρόγραμμα το οποίο δεν μπορεί να επικρίνει κανείς. Τώρα, δεν πιστεύω ότι όλα όσα αναφέρονται στο κατάλογό σας θα υλοποιηθούν κατά τη διάρκεια της θητείας. Έχω λοιπόν μια ερώτηση. γιατί στην ουσία όλα τα προγράμματα τα οποία εγκρίνουμε εμείς μαζί σας και με το Συμβούλιο θα πρέπει να έχουν στο κέντρο τον πολίτη. Έχουμε λοιπόν στη συνοχή και στο Ταμείο Συνοχής. Πιστεύετε ότι αυτά που έγιναν στην προηγούμενη θητεία μείωσαν τις διαφορές μεταξύ των διαφόρων περιφερειών στην Ευρώπη. Και τώρα σε αυτή τη νέα θητεία θα επιτευχθεί αυτό. Και όσον αφορά τη διαφάνεια, ρωτάω κάτι συγκεκριμένο. Μιλήσατε για μια μεθοδολογία όσον αφορά το κράτο δικαίου. Μπορείτε να μα πείτε τι ακριβώ εννοείτε για την μεθοδολογία αυτή. Μπορείτε να μα την παρουσιάσετε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Μπαζέσκου. Ένα λεπτό παρακαλώ. Domnule președinte, am privit programul ε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν δούμε όλες αυτές τις προτεραιότητες σας, αναρωτιόμαστε από πού θα έρθουν τα λεφτά. Είμαστε φιλόδοξοι, θέλουμε μια Ευρώπη κλιματικά ουδέτερη, να προστατεύσουμε το περιβάλλον, θέλουμε το πρόγραμμα πέμπτης γενιάς, θέλουμε ευρωπαϊκό στρατό, Θέλουμε κοινωνικό πυλώνα. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι υπάρχουν ε, τόσες πολλές προτεραιότητες ε, ταυτόχρονα ή ότι υπάρχουν τόσα λεφτά διαθέσιμα. Και το πράσινο ντύλι πρέπει να το δούμε με ευθύνη. Ε, τόσα λεφτά σε 10 χρόνια ε, δεν επαρκούν. Ελάτε στην Ρουμανία να δείτε εκεί πέρα τα ανθρακοριχεία. Λοιπόν, πρέπει να δείτε τι φτώχεια και τι ανεργία υπάρχει εκεί. Σας ευχαριστώ. Μαρία Μανουέλ Μάρξ έχει το λόγο. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το πρόγραμμα της ε, Κομισιόν για καλύτερη ρυθμίση είναι ε, ουσιαστικά το ίδιο. Δεν βλέπω κάτι το καινούριο. Η Κομισιόν θα χρησιμοποιήσει την τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη. Πώς θα μπορέσουμε να βελτιώσουμε τις υποδομές, ε, τις υπηρεσίες, όταν μιλάμε για τα κοινωτικά ταμεία, μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε ίσως για πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων Γνωρίζουμε τώρα ότι η τεχνητή νοημοσύνη και οι νέες τεχνολογίες θα μπορούσαν να βοηθήσουν τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Τι έχετε να πείτε γι' αυτό. Σας ευχαριστώ. Τσουχαντάρου έχει τον λόγο για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ρουμάνος είμαι. Έχω τρία αιτήματα για τη Ρουμανία. Πρώτον, Σέγγεν. Δεν κοστίζει τίποτα, ε, πληρούμε τις προϋποθέσεις και δεν γίνεται τίποτα. Μετά, για τις υποδομές. Στο Ιάσιο υπάρχει ένα νοσοκομείο πάρα πολύ σημαντικό ε, για τους ε, Ρουμάνους πολίτες ε, λείπουν ε, λεφτά. Λείπουν τα πράγματα αυτά για τους ψηφοφόρους μας δεν θέλουν να περιμένουν άλλο. Μετά, εξίσωση των αγροτικών επιδοτήσεων. Δικαιοσύνη μεταξύ των κρατών μελών. Νομίζω θα μας στηρίξουν κι άλλοι. Και έτσι θα πρέπει να αποτελέσουν προτεραιότητα αυτοί, αυτοί οι τρεις στόχοι. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ που περιοριστήκατε και εντό του χρόνου. Ντόμενεκ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Επίτροπε για την παρουσίασή σας. Στηρίζω το πρόγραμμα εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και χαίρομαι που αναφερθήκατε ως προτεραιότητα στην διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης. Και ξέρω ότι εσείς προσωπικά στηρίζετε να πρόκειται για μια ουσιαστική άσκηση και φιλόδοξη. Γι' αυτό πιστεύω, όπως είπαν και άλλοι συνάδελφοι, όπως και η Σκακέλερ αλλά και άλλοι, ότι αυτό που έγινε χτες με την ψηφοφορία που αναγκαστήκαμε να κάνουμε για το Brexit είναι η ευκαιρία να ενωθούμε περισσότερο μεταξύ μας ως Ευρωπαίοι και να προχωρήσουμε στην Ευρωπαϊκή Πολιτική Ενότητα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να στηρίξει λοιπόν την τάση των μεγάλων ομάδων υπέρ της Ευρώπης. Τώρα είναι η στιγμή να κάνουμε αυτό το ποιοτικό άλμα για πολιτική ολοκλήρωση. Ακριβώς γιατί αυτή είναι η εντολή που μας έδωσαν και οι Ευρωπαίοι πολίτες στις τελευταίες ευρωεκλογέ. Ευχαριστούμε. Η Μαργαρίτα Μάρξ τώρα. Ένα λεπτό παρακαλώ. Ε, πρόεδρε Σεύκοβιτς, σας ευχαριστώ για την παρουσίαση την οποία κάνατε του προγράμματος εργασίας για το 2020 με λεπτομέρειες έτσι ώστε να κατανοήσουμε τις φιλοδοξίες της Επιτροπής. καλό θα ήταν να ήταν πιο μακροπρόθεσμο, πολιετές το πρόγραμμα, αλλά παρόλα αυτά υπάρχουν κάποια στοιχεία στα οποία θα θέλαμε λίγο λεπτομέρειες. Δεν έχω χρόνο για περισσότερα. Καταρχάς η δυσκολία που θα αντιμετωπίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έτσι ώστε οι Ευρωπαίοι πολίτες να πιστέψουν περισσότερο στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα. Η δημοκρατία είναι φυσικά το καθοριστικό ε, πράγμα και σε επίπεδο διοργανικό. Και το δεύτερο είναι η χρηματοδότηση. Ε, τα ευρωπαϊκά όργανα πιστεύετε ότι ε, θα μπορέσουν να γίνουν πιστευτά εφόσον οι πολιτικοί υπεύθυνοι κατανοήσουν ότι οι προτάσεις τις οποίες κάνουν έχουν την δυνατότητα να χρηματοδοτηθούν. Ελπίζουμε λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας βοηθήσει. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να δώσω το λόγο τώρα στον Λόπες Αγγιλάρ. Ευχαριστώ. Αντιπρόεδρε Σεύκοβιτς, ανάμεσα στις προτεραιότητες του προγράμματος εργασίας της Επιτροπής υπάρχουν δύο. Όθηση της Ευρωπαϊκής Δημοκρατίας και του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής και αυτό έχει σχέση με την ε, επιτροπή στην οποία προεδρεύω στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Καταρχάς ένας μηχανισμός κράτους δικαίου μόνιμος ο οποίος ε, θα ενισχύει όλα τα κράτη-μέλη και δεύτερος να ενημερωθεί και να επικαιροποιηθεί το έγγραφο κανονισμός για την πρόσβαση ε, στα έγγραφα τα εσωτερικά μεγαλύτερη διαφάνεια. Επίσης να ενισχύσουμε την αίσθηση της αλληλεγγύης μέσα από τη Συμφωνία του Δουβλίνου και να ενισχύσουμε με τέτοιο τρόπο θα έλεγα για να αντιμετωπίσουμε με τα επαρκή μέσα την ανθρωπιστική κρίση που αντιμετωπίζουμε στην Ελλάδα και θα πρέπει επίσης να διευκρινιστεί ακόμα καλύτερα η κατάργηση της ποινικοποίηση αυτών οι οποίοι προσπαθούν να σταθούν αλληλέγγυοι ε, με τους μετανάστες όπως και με τις χώρες της Ένωσης που είναι στα εξωτερικά σύνορα και υφίστανται τις πιέσεις. Μίλερ, με Ευχαριστώ τον Επίτροπο. Οι στόχοι τους οποίους κατέθεσε είναι ενδιαφέροντες, αλλά απ' την άλλη δεν μπορούμε να αγνοήσουμε ε, το θέμα του ελάχιστου μισθού και της κοινωνικής ασφάλισης. Σε πολλές χώρες υπάρχει ένα τέτοιο σύστημα του ελάχιστου μισθού. Ε, είναι κάτι το οποίο καθορίζεται σε σχέση και με τον ε, μέσο μισθό ε, θα πρέπει να υπάρξει μια προσπάθεια καταπολέμησης των ε, μεθόδων φοροαποφυγής και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να χρησιμοποιήσει τους ισχύοντες μηχανισμούς και να μην βασίζεται πια στην αρχή της ε, ομοφωνίας. Νομίζω ότι η πρωτοβουλία την οποία έχουμε να αντιμετωπίσουμε εδώ θα μας βοηθήσει. Ευχαριστώ πολύ. Ε, Σιλβάνα Γκονσάλες. Ε, βλέπουμε ποιες είναι οι προτεραιότητες ε, για τις ε, δράσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ιδιαίτερα με το Green Deal και την κατεπίγουσα κατάσταση στην τομέα του περιβάλλοντος θα πρέπει να προσπαθήσουμε να δούμε και τι θα κάνουμε σε επίπεδο εξωτερικής δράσης και πώς θα υπερασπιστούμε το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και να συνδυάσουμε την οικονομική ανάπτυξη με την ανθρωπιστική βοήθεια. Οι χώρες οι οποίες λιγότερο συνεισφέρουν στην υπερθέρμανση υποφέρουν περισσότερο από τις κλιματικές αλλαγές. Σε άλλες περιοχές του κόσμου έχουν προχωρήσει αρκετά. Πώς εμείς θα προστατεύσουμε λοιπόν αυτό αυτούς οι οποίοι έχουν μετακινηθεί λόγω του κλίματος. Οι συμφωνίες της Καμπάλα και οι συμφωνίες της Καρταχένα στην Κεντρική Αμερική. Θα πρέπει λοιπόν να προχωρήσετε στις γραμμές που είπατε, αλλά πώς εμείς θα προστατεύσουμε αυτούς οι οποίοι εγκατέλειψαν τις αιστείες τους λόγω των κλιματολογικών αλλαγών και πώς θα βάλουμε στο εσωτερικό των κανόνων λειτουργία μας την ιδιότητα του κλιματολογικού ή κλιματικού πρόσφυγα. Ευχαριστώ Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να αναφερθώ και εγώ στο ζήτημα της καταπολέμησης της ε, φοροδεφυγής και φοροαποφυγής. Όπως ξέρουμε, η συζήτηση επικεντρώνεται τώρα ε, στον ΩΣΑ. Εντάξει, καλώς. Το πρόβλημα είναι ότι δεν μπορούμε να ελπίζουμε σε θετικό αποτέλεσμα των συζητήσεων ε, θετικό για εμάς κάποιες χώρες θα είναι εναντίον. Αυτό το οποίο μπορούμε να κάνουμε είναι οι ευρωπαϊκές χώρες μέλη του ΩΣΑ να κάνουν κάτι, κάτι το οποίο δεν συμβαίνει πάντα. Ζητώ από την Κομισιόν να χρησιμοποιήσει το πολιτικό της βάρος για να επηρεάσει το αποτέλεσμα των συζητήσεων στον ΩΣΑ. Ευχαριστώ. Ναι, ευχαριστώ. Σάντρα Περέιρα έχει το λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. κοινωνικά, πράσινα, αρκετή προπαγάνδα στα προγράμματα αυτά, αλλά δεν επικεντρωνόμαστε αρκετά στην κοινωνική ανάπτυξη προωθείται ένα πράσινο deal αλλά δεν συνειδητοποιείται ότι έχει υπάρξει μια αποτυχία. Ένας ε, κοινωνικός πυλώνας χρειάζεται λοιπόν που θα ασχολείται με την εκμετάλλευση και τις βλαβερές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ασκείται μεγάλη κριτική στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο και σε όλα τα υπόλοιπα. Θα ανακοινώσετε λοιπόν στους Πορτογάλους ότι αυτά δεν θα ισχύουν πλέον. Σας ευχαριστώ. Γουάλας για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, είπατε στο πρόγραμμα εργασίας σας ότι θα παρουσιάσετε το πρόγραμμα δράσης για τη δημοκρατία έτσι ώστε να καταστήσει τις δημοκρατίες μας πιο ανθεκτικές. Εγώ επισκέφτηκα μια φυλακή στην Ισπανία την προηγούμενη εβδομάδα όπου υπάρχουν καταλανοί ακτιβιστές φυλακισμένοι πάνω από δύο χώρα. Έχει πραγματικά σταματήσει πια η δημοκρατία εκεί. Είναι στο εσωτερικό της Ευρώπης η Ισπανική κυβέρνηση και το Ισπανικό δικαστικό σώμα δυστυχώς δεν κάνουν τη διάκριση των εξουσιών. Το θέμα δεν είναι η ανεξαρτησία ανεξαρτησία της Καταλωνίας είναι η άρνηση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πείτε μου ε, κύριε Επίτροπε τι θα κάνετε γι' αυτό. Είναι πραγματικά ντροπή αυτό που συμβαίνει. Ευχαριστούμε. Τελευταίος το Κατστιάι. Ρόμπερτ Ατσά, ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ, κύριε Σεύκοβιτς. Κοιτάξτε, είναι πολύ φιλόδοξο το πρόγραμμα και αν το καταφέρουμε θα αποτελέσουμε υπόδειγμα για ολόκληρο τον κόσμο, αλλά θα πρέπει ο μετασχηματισμός αυτός να είναι πραγματικά δίκαιος, έτσι ώστε η πράσινη οικονομία να μην έχει καταστροφικές συνέπειες στα κοινωνικά. Μιλήσατε για ένα ταμείο δίκαιη μετάβασης. Καλό θα είναι, αλλά αυτό το οποίο χρειαζόμαστε είναι να ωφεληθούν οι περιοχές ε, αυτές που το χρειάζονται περισσότερο. Πρέπει λοιπόν να βοηθήσουμε τις χώρες για <coughs> να πάνε τα λεφτά αυτά σε χώρες ε, που τα χρειάζονται όπως η Σλοβακία και η Πολωνία. Το ενεργειακό μείγμα αυτών των χωρών ε, βασίζεται σε άνθρακα, αέριο κτλ. και πυρηνικά. Πρέπει να ενώσουμε τις δυνάμεις μας ε, για να κάνουμε ό,τι μπορούμε έτσι ώστε ο μετασχηματισμός αυτός ε, να είναι θετικός. Σας ευχαριστώ. Τώρα τελείωσαν οι παρεμβάσει και θα δώσουμε το λόγο στον Αντιπρόεδρο τη Επιτροπή, τον Μάριο Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αξιότιμοι Ευρωβουλευτέ. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτήν την τόσο πλούσια συζήτηση. Σας ευχαριστώ για όλε σα τι παρεμβάσεις και χαίρομαι που μπορώ να πω ότι και αυτή η συζήτηση επιβεβαίωσε ότι το πρόγραμμα εργασίας μας αντικατοπτρίζει τις κοινέ μας προτεραιότητες. Σας ευχαριστώ πολύ για την εθάρρυνσή σας. Σας ευχαριστώ που ανεφερθήκατε σε διάφορες λεπτομέρειες πάνω στις οποίες θα πρέπει να εργαστούμε περισσότερο. Και ευχαριστώ και για αυτά που μας είπατε ότι πιστεύετε ότι λείπουν από το πρόγραμμά μας και θα το ε, δουλέψουμε, θα συνεργαστούμε μαζί σας. Νομίζω ότι το βασικό όταν παρουσίασε και την Επιτροπή τη η νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν ότι θέλει να είναι μια γεωπολιτική επιτροπή που θέλει να κάνει περισσότερα. Με τη δικιά σας στήριξη λοιπόν, με τη δικιά σας βοήθεια πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε. Θέλω εδώ να θυμίσω αυτό που μας είπε η κυρία Νίμπλερ αλλά και ο κύριος Μάρκες που μας είπαν ότι είναι καλό να έχει κανείς φιλόδοξο πρόγραμμα αλλά αυτό που είναι ακόμα πιο σημαντικό είναι η υλοποίησή του. Και Πολλοί από εσά είπατε λίγο πολύ το ίδιο ακριβώς πράγμα. Το παίρνουμε πάρα πολύ στα σοβαρά και η συνεργασία μας με τους συνομοθέτες και με εσά και με το Συμβούλιο σίγουρα θα φέρει περισσότερα αποτελέσματα. Η κυρία Κέλλερ αναφέρθηκε με φόρτιση στη χθεσινή συζήτηση. Ήμασταν όλοι εδώ χτες και νομίζω ότι ο αποχαιρετισμό των Βρετανών φίλων είναι κάτι που άφησε το στίγμα του σε μας. Θέλω να απαντήσω λίγο σε σχέση με αυτό ότι η χτεσινή πρόκληση τι σημαίνει για μας. Σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε μια καλύτερη Ευρώπη, μια πιο αποτελεσματική, μια πιο πράσινη, πιο κοντά στους πολίτες. Και πιστεύω ότι το επικοδομητικό έργο ε, γι' αυτό το φιλόδοξο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι το πρώτο βήμα στην κυρία Γιούρις Νίκολσον θέλω να πω κάτι. Αναφέρθηκε στις προκλήσεις που έχουν να κάνουν με τους ελάχιστους μισθούς. Ε, αυτό που το οποίο εμείς θα προτείνουμε είναι ένα πλαίσιο για ελάχιστους μισθούς και εννοείται ότι θα διαβουλευτούμε με τους κοινωνικούς εταίρους, με τις χώρες μέλη και θα σεβαστούμε 100% τις εθνικές παραδόσεις και τις συλλογικέ συμβάσεις. Αλλά πιστεύουμε ότι όλοι στην Ευρώπη αξίζουν ένα δίκαιο μισθό και αυτή τη δικαιοσύνη θέλουμε. Είναι πολύ βασικό ανθρώπινο δικαίωμα για τους πολίτες μας. Όσον αφορά τώρα τη διαδικασία επί κατά της Αυστρίας. Εξετάζουμε την απάντηση της Αυστρίας στην δικιά μας αιτιολογημένη γνώμη και εννοείται ότι θα ενημερώσουμε το Κοινοβούλιο στη συνέχεια. Προς τον κύριο αναφέρθηκε στον μηχανισμό ε, σχετικά με τον άνθρακα και την απαλλαγή από άνθρακα. Ήδη βρίσκεται στο πρόγραμμα εργασία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2020-2021. Όπως γνωρίζετε είναι κάτι αρκετά περίπλοκο. Χρειάζεται πολλή προετοιμασία και τους κατάλληλου μηχανισμού. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε σε διεθνές επίπεδο γι' αυτό. Εννοείται ότι θέλουμε να δούμε και χώρε όπω η Κίνα και άλλε να έχουν επίσης φιλοδοξίες, να έχουν ένα σύστημα όπως το ETS, το δικό μας σύστημα ε, δικαιωμάτων, ώστε να έχουμε ίσους όρους με τους άλλους και να φροντίσουν και άλλες μεγάλες οικονομίες να κάνουν την ίδια προσπάθεια για λιγότερο άνθρακα στις οικονομίες τους και στα προϊόντα τους. Τώρα, πολλοί από εσά επίση επέμειναν για το πόσο μεγάλη σημασία έχει το κράτο δικαίου. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σα και είναι σαφέ ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτή έχει αναλάβει τη δέσμευση να γίνεται σεβαστό το κράτο δικαίου εξίσου σε όλε τι χώρε μέλη. Κύριε Ντεσούτερ, θέλω να σας διαβεβαιώσω και εσά για το εξή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα διασφαλίσει πλήρη σεβασμό, και το τονίζω αυτό, πλήρη σεβασμό στη Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και θα αντιμετωπίσει αναδυόμενα ζητήματα όπως είναι η τεχνητή νοημοσύνη και η αναγνώριση προσώπων. Μετά από αυτά που είπε ο κύριος Σαρμάνη, ευχαριστώ πολύ για την παρέμβασή σας και μεταξύ άλλων και επικοδομητικών παρατηρήσεων αναφερθήκατε και στον αντισημιτισμό. Είχαμε χτες τη συζήτηση, είδαμε πόσο εφορτισμένε ήταν οι μαρτυρίε που ακούσαμε σε σχέση με το ολοκαύτωμα. Συμφωνώ μαζί σα λοιπόν και για το έργο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπής ήταν επίση κάτι πολύ σημαντικό. Και ο κύριος Γκαριγκάνοφ αναφέρθηκε στο πρόγραμμα εργασία μα και στο γεγονό ότι με την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου πολλά πανεπιστήμια που αποτελούσαν μέρος του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πανεπιστημίων δεν θα είναι πια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, να ξέρετε ότι θα συνεχίσουμε καλές επαφές με το Ηνωμένο Βασίλειο. Έχουμε κοινά προγράμματα, το Έρασμος κλπ. Αλλά επιπλέον θα φροντίσουμε ο Ευρωπαϊκός Εκπαιδευτικός Χώρος να είναι πραγματικότητα το 2025. Και γι' αυτό ε, θα δουλέψουμε εντατικά, όπως επίσης και για τους στόχους μας όσον αφορά την κατάρτιση. Προς την κυρία Γε, θέλω να πω ότι οι μελέτες αντικτύπου είναι πάρα πολύ σημαντικές και είμαι εγώ υπεύθυνο. Δεν πρόκειται να υπάρξουν νομοθετικές προτάσεις χωρίς να έχει προηγηθεί κατάλληλος, ε, κατάλληλη μελέτη αντικτύπου ακούμε τα επιχειρήματα και θα συζητήσουμε και με αυτούς που είναι κατά των προτάσεών μας και θα διασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει πλήρης διαφάνεια ε, μεταξύ των ε, θεσμικών οργάνων. Θα υπάρξει επίσης διαφάνεια γιατί θα καταλήξουμε και στο Μητρό μέχρι τα τέλη της χρονιάς αυτής. Όσον αφορά τώρα το θέμα της ένδυας θα το αντιμετωπίσουμε με τον ε, κοινωνικό πυλώνα, με τους ελάχιστους μισθούς και θα δουλέψουμε επίσης και για την εγγύηση των παιδιών. Κάποιοι από εσά αναφερθήκατε και είπατε ότι είναι πολύ σημαντικό μέτρο και με τη δικιά σας συνεργασία και με την κατάλληλη χρηματοδότηση θα συνεχίσουμε ώστε να αντιμετωπίσουμε και τα περιβαλλοντικά ζητήματα, της εκπομπές του εξοδίου του άνθρακα σε ολόκληρη την Ευρώπη, το θέμα της κατοικίας, γιατί πολλοί μένουν σε κοινωνικές κατοικίες. Θα το κάνουμε και με τη δικιά σας συνεργασία. Θα μειώσουμε τους λογαριασμούς που πρέπει να πληρώνουν για θέρμανση ή για να δροσιστούν, για τον ηλεκτρισμό που καταναλώνουν κλπ, το ηλεκτρικό ρεύμα. Έπειτα για το θέμα τη φοροδιαφυγή. Είμαστε πάρα πολύ σοβαροί και φυσικά και συνεργαζόμαστε με του εταίρου μα από τον ΩΣΑ και εφόσον υπάρξει συμφωνία στον ΩΣΑ εμεί θα κάνουμε ό,τι μπορούμε και θα αναλάβουμε τα κατάλληλα βήματα για να υλοποιήσουμε τη συμφωνία και εδώ. Αλλά σα διαβεβαιώ, αν δεν υπάρχει τέτοια συμφωνία μέχρι το τέλο του 2020 η Ευρωπαϊκή Ένωση θα δράσει μόνη τη. Δεν έχουμε περισσότερη υπομονή για να περιμένουμε κι άλλο να συνεχιστούν οι συζητήσεις και να μην πληρώνονται φόροι στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπως πρέπει. Ξέρω, Πρόεδρε, ότι έχουμε περιορισμένο χρόνο, αλλά θέλω ακόμα να πω στην κυρία Φρίτσαν για παράδειγμα, ότι θα συζητήσουμε σε βάθος με τους κοινωνικούς εταίρους και θα σεβαστούμε τα προνόμια τους. Γιατί τότε έχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα όπως γνωρίζουμε. Έρχομαι τώρα στη διεύρυνση. Νομίζω ότι ήμασταν ξεκάθαροι. Έχουμε νέα μεθοδολογία. Έχουμε διάσκεψη πολύ σημαντική στο Ζάγκρεπ που οργανώνει η Κροατική Προεδρία και την ευχαριστώ όπου θα έχουμε νέα όθηση, νέα ενέργεια για τη διαδικασία αυτή και τη δέσμευσή μας για την ε, Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία. Όσον αφορά τώρα το Ταμείο Μετάβασης και το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο, Πρόεδρε, η κυρία Μποναφέ ο κ. Χάρσιν και άλλοι αναφέρθηκαν σε αυτά. Όταν μιλάμε για το Ταμείο Δίκαιας Μετάβασης, μιλάμε για νέο χρήμα. Είναι επιπλέον από τις προτάσεις για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο που γνωρίζετε πολύ καλά. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι έτοιμη να δώσει αγώνα με το Συμβούλιο, ώστε να έχουμε κατάλληλη χρηματοδότηση για όλα τα φιλόδοξα ζητήματα που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμά μας. Και βέβαια θα πρέπει να φροντίσουμε όλοι να χρησιμοποιήσουμε τα χρήματα της δίκαιας μετάβασης εκεί που χρειάζονται περισσότερο. Εκεί που οι άνθρωποι πρέπει να καταρτιστούν, να βρεθούν χρήματα για τους ανθρακορίχους να χάσουν τη δουλειά τους, για ε, την ε, βιομηχανία προκειμένου η μετάβαση αυτή να είναι δίκαια και για όλους. Για όλους τους ανθρώπους, για όλες τις περιφέρειες και συμφωνώ απόλυτα μαζί σας επίσης για το πόσο μεγάλη σημασία έχει το θέμα των πολιτών δημοσιονομικών προοπτικών που πρέπει να είναι πάρα πολύ φιλόδοξες. Τι είπατε και κυρία Νίμπλερ και ο και άλλοι. Όπως γνωρίζετε θα έχουμε έκτακτη διάσκεψη κορυφής με αυτό το θέμα στην ημερήσια διάταξη. Θα είναι το θέμα πρέπει να υπάρχουν επιχειρήματα προς τους επικεφαλείς κρατών και κυβερνήσεων για το ότι χρειάζεται συμφωνία και σύντομα. Γιατί κάθε μήνα που περνάει καθυστερούμε με το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο και άρα κινδυνεύουν τα προγράμματά μας. Και πάλι, Πρόεδρε, αξιότιμοι Ευρωβουλευτές, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα τα θέματα που θίξατε. Τώρα θα υπάρχει διαφορετικό διάλογο με όλε τι επιτροπέ, θα συζητήσουμε όλα τα προγράμματα, όλε τι λεπτομέρειε και προσβλέπω σε αυτήν ακριβώ τη συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ. Διαδικαστικό, κύριος Μέλο. Νομίζω Νομίζω ότι ξεχάσατε να απαντήσετε τις δικές μου ερωτήσεις. Ε, καταρχάς στον τομέα της ενέργειας, αγωγή φυσικού αερίου. Θα ήθελα παρακαλώ, ε, ίσως ήταν μια μικρή παράληψη, να μου δώσετε μια απάντηση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα απαντήσει και αυτές τις ερωτήσεις. Ε, ε, με άλλες διαδικασίες. Ε, ευχαριστούμε τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ολοκληρώθηκε η συζήτηση. Θα περάσω στο επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Δήλωση πάλι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την απόκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις καταστροφές μετά από τις πλημμύρες στην Ισπανία. Θα ήθελα να ζητήσω από τους συναδέλφους παρακαλώ να σεβαστούν τον χρόνο που έχουν στη διάθεσή τους έτσι ώστε να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε εγκαίρως τις ψηφοφορίες. Θα δώσω ξανά το λόγο στον κύριο Σεύκοβιτς. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι και το θέμα το οποίο θα συζητήσουμε ακριβώς ε, ε, σημαίνει ότι η κλιματική αλλαγή είναι πραγματική και είναι ε, τα αποτελέσματα από δραματικά έως σουρεαλιστικά. Τα ακραία καιρικά φαινόμενα συμβαίνουν όλο και πιο συχνά και με μεγαλύτερη ένταση. Η ε, ξηρασία και οι δασικέ πυρκαγιέ πλέον δεν περιορίζονται μόνο στην Μεσόγειο. Έχουμε τροπικούς κυκλώνε στην Ιρλανδία και πλημμύρε σε ολόκληρη την Ευρώπη οι πρόσφατες πλημμύρες ε, στην Ισπανία από την Γλώρια ε, είναι άλλο ένα παράδειγμα και βεβαίως είμαστε στο πλευρό του Ισπανικού λαού που υποφέρει ιδιαίτερα τα συλληπιτήριά μας απευθύνονται σε αυτούς ε, που έχασαν τους τους η Ευρώπη είναι στο πλευρό του λαού της Ισπανίας έχουμε καθήκον να δώσουμε βοήθεια όταν έχουμε σοβαρές φυσικές καταστροφές. Ε, σκοπεύουμε να βοηθήσουμε για την αποκατάσταση των βασικών υποδομών. Με συγχωρείτε, κύριε Πρόεδρε. Δεν ακούγεται στα ισπανικά. Εντάξει, τώρα ακούγεται. Ωραία, μια χαρά. Συνεχίστε παρακαλώ. ξεκινήσω λοιπόν από το κομμάτι το οποίο έχει ιδιαίτερη σημασία για τους Ισπανούς ε, συναδέλφους. Λοιπόν, η Ευρώπη είναι στο πλευρό των Ισπανών και έχουμε τα μέσα για να δώσουμε βοήθεια όταν υπάρχουν σοβαρές φυσικές καταστροφές. Το Ταμείο Αλληλεγγύης θα βοηθήσει τους ανθρώπους για την αποκατάσταση των υποδομών ε, και για την διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς. Ε, είναι όμως ένα μέσο το οποίο χρειάζεται λίγο χρόνο για να κινητοποιηθεί. Επιπλέον το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο πρέπει να βελτιώσουν την ενεργοποίηση του Ταμείου και τους σχετικούς πόρους όταν η Κομισιόν ε, αξιολογήσει την αίτηση του κράτους μέλους. Μόλις δοθεί άμεση βοήθεια ε, στους ανθρώπους, ε, οι Ισπανικές αρχές πρέπει να αξιολογήσουν τις ζημιές για να δουν εάν φτάνει το κατόφλι του 1,5% του ΑΕΠ της περιφέρειας. Αυτό είναι βασική προϋπόθεση για μια επιτυχή αίτηση. Οι Ισπανικές αρχές γνωρίζουν ε, τις ε, συνθήκες ε, και βεβαίως η Κομισιόν είναι έτοιμη για να δώσει κάθε βοήθεια. Αξιολογούμε μια προηγούμενη Ισπανική έτσι που λάβαμε τον Νοέμβριο που περιλαμβάνει την περιφέρεια της Βαλένθιας, Μούρθια, Καστίγια Λαμάντσα και Ανδαλουσία για τα καιρικά φαινόμενα του Σεπτεμβρίου που μας πέρασε. Οι πληροφορίες μας δόθηκαν μόλις αυτήν την εβδομάδα ε, και έχει δοθεί ήδη μια προκαταβολή 5,7 εκατομμυρίων ευρώ. Στο μέλλον όμως γνωρίζουμε ότι πρέπει να είμαστε έτοιμοι να κάνουμε περισσότερα. Αυτά τα οποία συνέβησαν στην Ισπανία είναι δυστυχώς πρόγευση των όσων ε, θα έρθουν καθώς συνεχίζεται η κλιματική αλλαγή. Το Ταμείο Αλληλεγγύης βεβαίως είναι μια στήριξη αλλά πρέπει να δρούμε και προληπτικά. Γι' αυτό τα τελευταία χρόνια η Κομισιόν ρίχνει ιδιαίτερο βάρος στην πρόληψη, την κλιματική προσαρμογή και την διαχείριση του κινδύνου. Για γιατί οι τοπικέ και περιφερειακέ αρχές είναι οι πρώτε που αντιμετωπίζουν τι θεομηνίες. Γιατί είναι οι πρώτε αυτέ που θα πρέπει να επενδύσουν όσον αφορά το μέλλον και έτσι συμβάλλουν σε βιώσιμη ανάπτυξη. Έχουμε με αυτό το πνεύμα που διαπνέει την πολιτική συνοχή 14 με 20 για να κάνουμε την προσαρμογή και την πρόληψη των κινδύνων. Έχουμε ε, ένα ολόκληρο πλωστάσιο για να υποστηρίξουμε αυτές τις αρχές για την διάβρωση, της ε, δασοπυρκαγιές και τις άλλες ε, θεομηνίες, καταστροφές και να έχουμε συστήματα έγκυρες προειδοποίησης, προπαρασκευή στρατηγικών και κατευθυντηρίων και επίσης ε, συνειδητοποίηση, βιώσιμη διαχείριση των δασών και της γης. Επίσης είδαμε ότι θα πρέπει να υπάρξει υποδομή πράσινη για παιδιάδες και αστικές περιοχές. Επίσης ενθαρρύνουμε τα κράτη μέλη το ώστε να γίνει αξιολόγηση και έτσι να προλάβουμε και τις επιπτώσεις της πλημμύρας. Ε, υλικό, εξοπλισμός, υποδομές και μονάδες πολιτικής προστασίας. Επίσης βοηθάμε σε βελτίωση και σε συστήματα έγκαιρες προειδοποίησεις, να έχουμε αισθητήρε και δορυφόρους, ε, οπότε να υπάρχουν όλα τα στοιχεία για γεωλογικά φαινόμενα, αλλά και πλημμύρες και άλλα φαινόμενα. Οπότε έτσι νομίζω ότι θα μπορέσουμε να παρακολουθήσουμε, να υποπτεύσουμε, να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε και να υπάρξει και συντονισμός. Τέλος, ε, θέλουμε ευελιξία στο πρόγραμμα συνοχής, και οι τροποποιήσεις του προγράμματος μπορεί να προταθούν και έτσι μπορούμε να κατευθύνουμε τους πόρους εκεί που χρειάζονται περισσότερο. Οπότε, εάν πρέπει να επιφέρουμε αλλαγές, ακόμη μπορούμε να το κάνουμε σε αυτή τη φάση χρηματοδότησης. Η πρότασή μας για την συνοχή μετά το 20 καλύπτεται και στην, ε, στους στόχους που έχουμε για το κλίμα και την προσαρμογή, προπαρασκευή σε εξοπλισμό, καταφύγια, υποδομές, σύστημα έγκυς προειδοποίησης και κατάρτιση εκπαίδευση, για πολιτική προστασία σε σχετικές μονάδες και αυτό θα είναι διασυνορικού χαρακτήρα και σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε κύριε Αντιπρόεδρε για την παρέμβασή σας. Περνάμε στους συναδέλφους. Πρώτα κυρία Δολόρες Μονσεράτ για δύο λεπτά. Παρακαλώ να τηρείτε το χρόνο σας. Δεν μπορώ να ξεκινήσω χωρίς να α, θυμηθώ τα άτομα που έχασαν τη ζωή τους και τις οικογένειές τους, τους αγνοούμενους, τους, τραυματίες, τραυματίες. Μεταφέρω την στοργή και την συμπαράστασή μας. Πρόσφατα είχαμε την καταιγίδα Gloria και πριν από λίγους μήνες άλλη καταιγίδα, την Τάνα. Τόσοι άνθρωποι είδαν τις επιχειρήσεις τους στα σπίτια τους, ε, τα χωράφια τους, ε, ζωές τους να καταστρέφονται. Είδαμε πόσο απαραίτητα για την οικονομία και το οικοσύστημα με σύστημα όπως το Δέλτα του Εύρου που είναι μοναδικό οικοσύστημα για την Ευρώπη και την Ισπανία που είναι τρίτος παραγωγός ρυζιού στην Ευρώπη. Εξαφανίστηκαν καλλιέργειες ε, και οι ζημιές είναι ύψους 4 εκατομμύριων ευρώ. Στην Βαλέσια τα εσπεριδοειδή, τα παρακυπευτικά και η κτηνοτροφία υπέστησαν ζημίες περίπου 63 εκατομμύρια ευρώ. Οι Βαλεαρίδες έχασαν ολόκληρες ακτές. Η Ανταλουσία, η Μούρσια, η Καστίγια Λαμάντζα, η Αραγών, όλες περιοχές που επλήγησαν. Θέλουμε άμεση αντίδραση και από την κυβέρνηση της Ισπανίας. Θέλουμε η κυβέρνηση της Ισπανίας να κάνει γρήγορη αξιολόγηση των ζημιών, να επισπεύσει την αποζημίωση, να κινητοποιήσει το Ταμείο Αλληλεγγύης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να ανακηρύξει ως ε, ζώνες καταστροφής τις ε, ε, πληγήσεις περιοχές. Θα πρέπει επίση να αυξήσουμε τον προπολογισμό τη κοινή γεωργική πολιτική για να έχουμε περισσότερα κονδύλια που θα χρηματοδοτούν την πρόληψη κινδύνων για του γεωργού και κτηνοτρόφου. Θέλουμε ένα Green Deal που θα είναι φιλόδοξο και θα προστατεύει το περιβάλλον από τι κλιματικέ αλλαγές. Θα βελτιώνει τι ε, υποδομέ, ε, την καθαριότητα και την ε, εξυγίαση των δασών και των ποταμιών μας για να αποφύγουμε ακραία καιρικά φαινόμενα οι Ισπανοί που επλήγησαν από την καταιγίδα δεν μπορούν να περιμένουν ούτε μια μέρα παραπάνω και ακούραστα το Ισπανικό Λαϊκό Κόμμα θα στέκεται στο πλευρό τους και θα κάνουμε τα δύνατα δυνατά για να αποζημιωθούν το συντομότερο δυνατό. Η κυρία Κριστίνα Μαέστρη Μαρτίν Δελμάργο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μόνο σε μετά από λίγους μήνες κοινοβουλευτικής θητείας και ήδη έχουμε τη συζήτηση για την τρίτη θεομηνία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τρίτη φυσική καταστροφή και πολύ φοβάμαι ότι δεν θα είναι και η τελευταία. Γιατί οι κλιματικές αλλαγές είναι μια αναφυσβήτητη πραγματικότητα. Ε, είναι προφανέστατο και από τις τελευταίες ε, καταιγίδες και τα κράτη φαινόμενα. Πάνω από 500 εκατομμύρια στην Ευρωπαϊκή Ένωση εκτίθενται σε αυτά τα φαινόμενα από κίνδυνο ε, από κίνδυνο πλημμυρών ή από πλημμύρες ε, σε παράκτης περιοχές. Οπότε το πρόβλημα αυτό δεν είναι μόνο της Ισπανίας, αλλά του συνόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε σοβαρά και να λάβουμε μέτρα για να το αντιμετωπίσουμε. Αλλά θα πρέπει κατεπηγόντως να ενεργοποιηθεί το Ταμείο Αλληλεγγύης. Πάρα αυτά. Το χρειαζόμαστε γιατί και αυτό θα συνάδει στη συνοχή. Σήμερα είναι η Ισπανία, αλλά αύριο θα είναι μια άλλη χώρα. Θα πρέπει να έχουν πρόσβαση για να χορηγηθούν γρήγορα αποζημιώσεις ε, στους ε, πληγέντες. Βέβαια δεν μπορούμε να αποζημιώσουμε το χαμό την απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής, αλλά τουλάχιστον να αποζημιώσουμε τις οικογένειες ή τους ε, κλάδους που επλήγησαν από την τελευταία καταιγίδα. Οπότε ταχύτητα και ελαστικότητα, όπως είπατε κύριε Πρόεδρε, για την εφαρμογή αυτού του Ταμείου. Σας ευχαριστώ. Η Σουζάνα Σολή Πέρε για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Η καταιγίδα Κλώρια χτύπησε αμήλικτα την Ισπανία. 14 νεκροί, 83 τραυματίε, 2 αγνοούμενοι. Ε, Ολέθρια ως απολογισμός. Ε, οι Αραγών, οι Βαλεαρίδες, η Μούρση, η Ανταλουσία είχαν εκατομμύρια ζημίες ε, στη γεωργία, την κτηνοτροφία, στα σπίτια. Ε, καταστράφηκε οι παραγωγές περιδοειδών, χάθηκαν παραλίες. Ε, μιλούμε για περιοχές που εξαρτώνται από τον τουρισμό και την γεωργία και κτηνοτροφία. Και δυστυχώς δεν είναι μεμονωμένα αυτά τα φαινόμενα. Πριν από λίγους μήνες είχαμε την καταιγίδα Ντάνα και οι πυρογνώμονες μας βεβαιώνουν ότι τέτοια κρέα και φαινόμενα θα αυξηθούν. Θα θέλαμε λοιπόν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποτελεσματικά μέτρα και αντίδραση. Εγώ θα σα πρότεινα τρει δράσει. Καταρχήν, το Ταμείο Αλληλεγγύη θα πρέπει να το ενεργοποιήσουμε και αν τέτοια ακραία καιρικά φαινόμενα αυξηθούν, θα πρέπει να αυξήσουμε και την πρικοδότηση του Ταμείου Αλληλεγγύη για να μπορούμε να αποζημιώσουμε του πληγέντε. Δεύτερον, θα πρέπει να διευκολύνουμε ε, και να επιταχύνουμε τι διαδικασίε, να μην είναι χρονοβόρε και γραφειοκρατικέ. Ακόμη οι γεωργοί αγρότε τη Ισπανία περιμένουν τι αποζημιώσει από την καταιγίδα Ντάνα. Επίση, να βελτιώσουμε τα συστήματα πρόληψη κινδύνου και πρόληψη θεομηνιών καθώ και προσαρμογή στι κλιματικέ αλλαγές. Αυτό είναι απαραίτητο για να σώσουμε ανθρώπινε ζωέ. Επίση, θα πρέπει να εφαρμόσουμε μία από τι θεμελιώδει αξίες τη Ευρωπαϊκή Ένωση την αλληλεγγύη, γιατί τώρα είναι που τη χρειαζόμαστε περισσότερο από ποτέ. Ευχαριστώ. Για ένα λεπτό, η κυρία Διάννα Ρίβα Ιχινέρ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πρόεδρε την περασμένη εβδομάδα ο Γιγλώνα και η καταιγίδα Γλώρια χτύπησαν την Καλονία και την υπόλοιπη Ισπανία. Πάνω από 13 ε, άνθρωποι έχασαν τη ζωή του και βλέπουμε ότι η αλλαγή του κλίματο και στην οικολογία και στη γεωργία έχει ε, συνέπειε χωρί προηγούμενο και ακριβώ αυτό συμβαίνει λόγω τη αλλαγή του κλίματο. Οπότε το πέρασμα αυτή ε, ε, τη καταιγίδα χτύπησε και, ακόμα και τη θάλασσα, τα, τα παράλια, όλε τι υποδομέ και στην λεκάνη Τορδέα Ιβέρ και λέμε τώρα ότι προκατρακτικά μόνο στην Βαρκελόνη είναι 4 εκατομμύρια ζημίες και 16 στον πρωτογενή τομέα 16 εκατομμύρια οπότε χρειάζεται γρήγορη αντίδραση και γι' αυτό ζητούμε από την Επιτροπή και από την κυβέρνηση τα εξή τρία πρώτα πρώτα επιγόντως να ενεργοποιήσουν τους πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξη και να συγχρηματοδοτήσουν την αποκατάσταση ζημιών. Δεύτερον, όπως είπατε, να ενεργοποιηθεί το Ταμείο Ελληνική, αλλά τελευταίο να υπάρχει συγκεκριμένο πρόγραμμα δράσης για την ε, ε, Μεσόγειο και για το Δέλτα του ποταμού Εύρου και να προχωρήσουν τα σχέδια της καταλαγικής κυβέρνησης και των τοπικών φορέων. Σας ευχαριστώ. Για ένα λεπτό τώρα ο Μάρκο Ντρεώστο. Πρόεδρε, ευχαριστώ και θέλω πρώτα-πρώτα να εκφράσω την ελληνική μου προς τους ε, Ισπανούς ε, συναδέλφους αλλά και την Ισπανία γενικότερα για τα όσα υπέστησαν από αυτήν την ε, πλημμύρα και θα πρέπει να ενεργοποιήσουμε την προστασία του του μηχανισμού πολιτικής προστασίας τόσο ώστε να κάνουμε κάτι για αυτή τη φυσική καταστροφή θα πρέπει όμως να υπάρχει μια καινούργια νοοτροπία για πρόληψη ε, καινούργιες στρατηγικές και μακρόπνες ούτως ώστε να μας βοηθήσουν να αποφύγουμε ή τουλάχιστον να συγκρατήσουμε το κόστος και σε ανθρώπινε ζωέ και σε ε, οικονομική ζημία. Οπότε θα πρέπει να υπάρχει επαρκής κατάρτιση του κόσμου, του προσωπικού, ε, πολιτικής προστασίας. Ε, έχουμε βέβαια και την καινούρια πρόταση κανονισμού για αυτό το σκοπό. Είμαστε διαθέσιμοι να βοηθήσουμε όποτε χρειάζεται για τέτοιες ε, συμφορές. Σας ευχαριστώ. Έκλεισε και ο κατάλογος των ομιλητών στη διαδικασία Catch the Eye. Κυρία Βηγιανόεβα Ρουίς, ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η καταιγίδα Γκλώρια χτύπησε αμήλικτα την Ισπανία. Ε, Βαλερια, Βαλαρίδες, Μούρση, Ανταλουσία είναι από τις πληγήσεις περιοχές. 14 νεκρούς θρυνούμε και δεκάδες τραυματίες. Ήταν καταστροφικά τα αποτελέσματα της Γλόριας: επιχειρήσεις, ε, ε, ακτές, καλλιέργειες, στέγη. Αυτό οφείλεται στην κακή πολεδομική και χωροταξική πολιτική ανεύθυνων και διαφθαρμένων πολιτικών που κατέστρεψαν τις ακτές και παραλίες μας. Τέτοια ακραία καιρικά φαινόμενα επηρεάζουν τη χώρα μας που κατά το 2019 είχε πολλές πλημμύρες και υπερχείληση υδάτων στην Ανταλουσία, στη χώρα των Βάσκων, στην Αβάρα και οι ζημίες ε, είναι πολλών εκατομμυρίων για την περιοχή και την οικονομία μας. Θέλουμε λοιπόν ενίσχυση για να ενεργοποιηθεί η, το Ταμείο Αλληλεγγύης. Θα πρέπει να αλλάξουν τα κριτήρια ώστε να μην λαμβάνονται μόνο μεμονωμένα τις τελευταίες καταιγίδες αλλά ως το σύνολο του ετήσιου μέσου όρου. Επίση, θέλουμε να καταπολεμηθεί η πολεοδομική διαφθορά και απάτη και πολιτικέ για να αντιμετωπίσουμε την κλιματική αλλαγή. Α μην περιμένουμε την επόμενη συμφορά για να αντιδράσουμε. Είναι ζήτημα ζωή και θανάτου. Σας ευχαριστώ. Ο Αντώνη Κομίνη Ολιβέρας έχει το λόγο για ένα λεπτό. Micro. Σας ευχαριστώ. Την περασμένη εβδομάδα όντως επλήγησαν οι παραλίες και ακτές της Καταλωνίας και της Βαλένθια ε, τις καταιγίδες που όλος παραδόξως την αποκαλούμε γλώρια ή ευδοξία και έπληξε και την ε, Βόρεια Καταλωνία αλλά και αυτόνομες περιοχές όπως τη Μούρσια, την ε, Ανταλουσία, την Αραγών. Στην Καταλωνία, στη Ζηρώνα είχαμε καταστροφή πολλών καλλιεργιών και πολλών κατοικιών. Σίγουρα ο λόγος είναι η κλιματική αλλαγή. Αυτό είναι ο πρωταρχικός λόγος. Στην περίπτωση όμως του Δέλτα του Εύρου ενισχύθηκε η καταστροφή από την κατάσταση ε, της, του Δέλτα του, ε, ποταμού, ποταμιού αυτού και πριν την θεομηνία. Γιατί δυστυχώς ε, κατεβαίνουν οι ζήματα μέχρι τις εκβολές και το Δέλτα με αποτέλεσμα να, να μην γίνεται καλή εκαθάριση των υδάτων. Έχουμε χάσει ήδη εκατοντάδες εκτάρια ε, και μετά την καταιγίδα τρία χιλιόμετρα μπήκε μέσα στην ενδοχώρα το αλμυρό νερό. Χάσαμε 15 ε, ε, εκατομμύρια εκτάρια στη Γυρόνα. Τι προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να ανακτήσουμε αυτές τις χαμένες περιοχές, τις γέες που χάσαμε λόγω του, της καταιγίδας. Ο Εστέμπαν Κονσάλες πώς έχει το λόγο. Μπορεί να φανταστείτε κύριε Επίτροπε ότι τι ζημία έπαθε η πατρίδα μας. Μία ε, πλημμύρα είναι μια καταστροφή. Δύο πλημμύρες μέσα σε λίγους μήνες είναι μια κλιματική αλλαγή καταστροφική. Τον Σεπτέμβριο η ζημία στην περιοχή της ε, ε, 1,5 ε, δι, 62 εκατομμύρια ευρώ στη συνέχεια ε, ήταν η ζημία ε, και χάθηκαν επίσης ανθρώπινες ζωές. Όμως δεν έχει έρθει η βοήθεια από την Ευρώπη. Το Ταμείο Ελληνικής από το Σεπτέμβριο ακόμη δεν έχει ενεργοποιηθεί. Το έχουμε ζητήσει ως κυβέρνηση και δεν έχει γίνει τίποτα για τις κοίτες των ποταμών, για τις όχθες των ποταμών οπότε ε, τελικά αυτή η αλλαγή του κρεμμυς χτυπήσει μόνο εμάς εμείς είμαστε στην πρώτη γραμμή αλλά όλους θα τους χτυπήσει πρόκειται να ξανασυμβεί αυτό και ε, σε μεγάλο βαθμό αυτή η ζημία μπορεί να αποφευθεί. Χρειαζόμαστε κάτι να γίνει για την Βαλένθια, για την Αλμπουφέρα που είναι ένα κόσμο με τις φύσεις και θα πρέπει επομένω κάτι να γίνει και τα ταμεία της μετάβασης για την οικολογική μετάφαση δεν θα πρέπει μόνο να λαμβάνουν υπόψη την αλλαγή της οικονομίας αλλά θα πρέπει να φροντίσουν να και να καλύψουν και την προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος. Όλα αυτά τα οποία έπαθε η χώρα μας θα πρέπει να ληφθούν υπόψη, οπότε και οι επιχειρήσεις και η γεωργία και ο κόσμος που έχουν ε, ζημιωθεί ε, θα πρέπει να γίνει κάτι και κυρίως για τις ανθρώπινες ζωές που χάθηκαν. Συνάδελφοι παρακαλώ να τηρήσετε τα όσο προβλέπει ο κατάλογος των αγορητών και να κάνουμε ησυχή και να σεβαστούμε του ομιλητέ. Το λόγο έχει η κυρία Μακουλάδα Ροντρίγκε Πινιέρο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Πρόεδρε και κύριε Επίτροπε, 14 ήταν τα θύματα τη καταιγίδα. Αυτό ήταν για δεύτερη φορά μέσα σε τέσσερι μήνε. Στι ακτέ, σε παιδιάδε, ε, υπέστη μελώ αυτέ τι ισοποδοτικέ καταστροφέ και αυτά γίνανε ιδίως στην περιοχή της Βαλένθια, την εκλογική μου περιφέρεια. Ε, είμαστε πιο ευάλωτες στην Ευρώπη, οπότε θα πρέπει κάτι να κάνει ε, επιγόντως η Επιτροπή να καλύψει τον κόσμο να συνεργαστεί με τις αρχές της χώρας και ε, σε κατεπήγοντες ρυθμούς να επιστατευθούν όλοι οι πόροι που υπάρχουν στα ταμεία ούτως ώστε σύντομα κάτι να γίνει και επίση είναι σημαντικό κάτι να γίνει μέσω μακροπρόθεσμα και έτσι στο μέλλον να συγκρατήσουμε τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής. Γι' αυτό κύριε Επίτροπε πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εκπονήσει κάποια στρατηγική για την αλλαγή του κλίματος αλλά συγκεκριμένα για την ε, Μεσόγειο πιέζει ο χρόνος η Αλμπουφέρα, το Δέλτα του Εύρου στη, στη Μούρφια επίσης ε, είναι χώροι φυσικής ομορφιάς φυσι, ε, μεγάλης αξίας και θα πρέπει να συνεργαστούν όλοι οι συναρμόδιοι να μην χαθεί άλλη ανθρώπινη ζωή ε, περιμένει από εμά ο κόσμος κάτι να κάνουμε πρέπει να τους απογοητεύσουμε Συνάδελφοι, να σας ζητήσω και πάλι να σέβεστε τους ομιλητές. Σας παρακαλώ λίγη ησυχία. Τελευταίος ομιλητής στον κατάλογο. Πώς πει Για ένα λεπτό. Dear colleagues, Συνάδελφοι, σας παρακαλώ να κάνετε ησυχία για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση. Διδάλλως, θα καθυστερήσουν οι ψηφοφορίες. Να δώσω λοιπόν το λόγο στον συναδελφό μας Γύρι Πόσπισιλ. Για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε και θα προσπαθήσω να είμαι σύντομο. Να εκφράσω την αλληλεγγύη μου και την συμπαράστασή μου στο λαό της Ισπανίας. Η Επιτροπή θα πρέπει να παρέχει βοήθεια όσο πιο γρήγορα γίνεται. Στην χώρα μου έχουμε πολύ καλές εμπειρίες με το Ταμείο Ελεγγύης. Το μοναδικό πρόβλημα ήταν η διάρκεια για την επεξεργασία των αιτήσεων. Αν θα μπορούσε λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει ό,τι μπορεί προκειμένου να διεκπαιρεωθούν γρήγορα αυτές οι αιτήσει. Το Ταμείο Αλληλεγγύης είναι σπουδαίο εργαλείο. Αλλά αν χρειάζεται τα κράτη-μέλη να περιμένουν μισό έτος μέχρι ότου καταφτάσουν οι πόροι αυτοί, η καθυστέρηση αυτή θα είναι καθοριστική. Και πιστεύω ότι θα πρέπει να αναφερθεί ε, να αναφερθεί το Ταμείο Αλληλεγγύης. Θα χρειαστεί επίσης ε, πιο πολύ χρηματοδότηση στα κράτη τα οποία πλήττονται από την αλλαγή του κλίματος και θα πρέπει να βρούμε ένα μηχανισμό για να μπορούμε να αντιδρούμε με πιο ευέλικτο τρόπο. Αν χρειάζεται κάθε φορά μήνες για να εξετάσουμε την κάθε αίτηση και μετά να αποφασίζει το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο και τελικά η όλη διαδικασία να παίρνει 12 μήνε, δεν ξέρω τι νόημα έχει. Να προσπαθήσουμε λοιπόν να βοηθήσουμε την Ισπανία και να καταστήσουμε τη διαδικασία πιο αποτελεσματική, να μειώσουμε το χρόνο αναμονή. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ. Περνάμε στη διαδικασία Catch the Eye τώρα. Το λόγο έχει η Ρόζα Σταράς Φεραγκούτ. Ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η καταιγίδα Γκλώρια ε, μάστησε την Ισπανία και κυρίως ε, τη Μεσόγειο. Κύματα ύψους 14 μέτρων στην γενέτειρά μου της Βαλεαρίδες ε, έχουν ε, αποδεκατήσει παραλίες, έχουν χτυπήσει τη Βαρκελόνη, τη Βαλένσια, τη Μαόν. Είχαμε νεκρούς και αγνοωμένους τεράστιες ζημιές, ανυπολόγιστες, προβλήματα στον ανεφοδιασμό. Όλα αυτά έχουν αντίκτυπο και ανθρώπινο και οικονομικό και κοινωνικό σε, όλη την Ισπανία. Μανακόρ, Σελβένσο, Φέλανιτς, Σάντανη ήταν από τους δήμους των Βαλεαρίδων που επλήγησαν δραματικά από την τελευταία καταιγίδα. Ζητούμε λοιπόν την ενεργοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης πρόσφατα στην προηγούμενη κοινοβουλευτική θητεία έγινε μια τροποποίηση για να καταργηθούν οι γραφειοκρατικές διαδικασίες. Θα πρέπει λοιπόν να αναζωογονήσουμε το πνεύμα της Ευρωπαϊκής Αλληλεγγύης που είναι η καρδιά, η ψυχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό χρειάζονται οι περιοχές της Ισπανίας που επλήγησαν από την καταιγίδα. Ευχαριστώ. Συνάδελφοι, παρακαλώ. Θέρμο παρακαλώ. Ας δείξουμε σεβασμό προς τους ομιλητές και να ολοκληρώσουμε τη διαδικασία Catch the Eye. Το λόγο έχει τώρα η Αλήση Άμσγκινε για ένα λεπτό. No va. Está rojo. Micro. Micro. Es que no funciona. Que no está rojo. Δεν ανάβει το λαμπάκι, λέει ο μιλήτρια. Δεν δουλεύει. Ε. micro now. Is, now working? Yeah, it's working. Okay. Gracias, presidente. Gloria tiene que ser una Πρόεδρε, θα, αυτό πάλι είναι ένα καμπανάκι κινδύνου για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να λάβει δράση γιατί οι συνέπειε αλλαγή του κλίματο χτύπησαν την ε, περιοχή τη Μεσογείου στην ε, Ισπανία και στην Μαγιόρκη είχαμε μεγάλε καταστροφέ, αλλά και τον Οκτώβριο έγινε το ίδιο. Την περασμένη εβδομάδα το Gloria χτύπησε βαλερίδες νήσου, Καταλωνία και Βαλένθια και είχαμε 14 νεκρούς στι βαλερίδες, 12 ε, ε, αγνοούνται και θέλω να που εκφράσω την συμπαράστασή μου στις οικογένειές τους ε, οπότε λοιπόν, θα πρέπει ε, να γίνει κάτι γιατί είναι συχνή η, η, το φαινόμενο αυτό στις περιοχές μας και θα πρέπει επομένως να υπάρχει ο μηχανισμός στα πλαίσια του Ταμείου Αλληλεγγύης για να ενεργούμε κάποιους ε, πόρους κατεπηγόντως για τις περιοχές που χτυπήθηκαν από αυτή την κακογερία εκτός από τις ηλικίε και ανθρώπινες ζημίες είχαμε πρόβλημα για τον ανεφοδιασμό σχεδιασμό των ε, ειδών διατροφής. Άλλος ένας λόγος επομένως να λάβετε υπόψη το ότι είμαστε μειονεκτούσα περιοχή στις βαλέρίδε ε, νήσους. Σας ευχαριστώ. Η συνάδελφος Ελικάος έχει το λόγο για ένα λεπτό. Colleagues, Συνάδελφοι, σήμερα συμμετέχω στην τελευταία μου συζήτηση ως βουλευτής ε, του Ηνωμένου Βασιλείου και ως πράσινη πρέπει να πω ότι είναι λυπηρό το γεγονός ότι είναι αυτή η τελευταία συζήτηση μια συζήτηση αλληλεγγύης για φυσική καταστροφή στην Ισπανία. Θέλω να εκφράσω την αλληλεγγύη μου και την ε, συμπαράστασή μου προ το λαό τη Ισπανία. Δεν μπορούμε να αποκαλούμε τέτοιες, ε, τέτοια καιρικά φαινόμενα ω φυσικά φαινόμενα, γιατί τη αλλαγή του κλίματο θα καταστεί όλο και πιο έντονα τα φαινόμενα αυτά. Χρειαζόμαστε λοιπόν μια πιο ταχεία και πιο δυναμική ευρωπαϊκή αντίδραση για την αλλαγή του κλίματο. Σήμερα έχουμε 28 νέου μαζί μα στις εξέδρε από τα West Midlands. Η δικιά του γενιά λοιπόν είναι αυτή που έχει φωνάξει και η φωνή του έχει ακουστεί. Θα πρέπει να είμαστε πιο γρήγοροι και πιο δυναμικοί σε ό,τι αφορά την αντίδραση στην κλιματική και οικολογική κρίση. και παρά το γεγονό ότι δεν θα είμαι πλέον μέλο του Κοινοβουλίου για, λόγω του Brexit, θα επιστρέψω στον Εμένο Βασίλειο για να ζητήσω να προωθηθεί αυτή η γρήγορη ανταπόκριση στην αλλαγή του κλίματο. Και σα καλώ να υψώσετε κι εσεί το επίπεδο τη φιλοδοξία και ελπίζω η αλληλεγγύη να συνεχίσει να επικρατεί όλο και πιο ισχυρή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλουμε λοιπόν να ανταποκριθούμε στι προκλήσει τι οποίε αντιμετωπίζουν όλοι μαζί. Σας ευχαριστούμε κυρία Τζόνς και τελευταία παρέμβαση στο Catch the Eye, η κυρία Γκυλάρ Μαρσάλη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να εκφράσω την αλληλεγγύη μου προς τα θύματα του, της καταιγίδα Gloria που χτύπησε με μεγάλη δρυμύτητα την ανατολική, τις ανατολικές ακτές της Ισπανίας. Δυστυχώς είχαμε και νεκρούς και τεράστιες ζημιές, κυρίως στη Γεωργία. Το περασμένο Σεπτέμβριο, όπως είπαν και άλλοι συνάδελφοι, ε, ζήσαμε και άλλη καταιγίδα, την καταιγίδα Ντάνα, που επίσης προκάλεσε σοβαρές ζημιές στην Ισπανική Γεωργία. Δυστυχώς οι αγρότες μας ακόμη δεν έχουν λάβει τις αποζημιώσεις και τις ενισχύσεις που τους είχαμε υποσχεθεί. Και η νέα καταιγίδα, η Γκλώρια, ουσιαστικά έπληξε ακόμη περισσότερο τους παραγωγούς οποροκυπευτικών, ε, εσπεριδοειδών και τους κτηνοτρόφους που είναι τα πρώτα θύματα αυτής της καταστροφής. Ευχαριστώ την ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αλληλεγγύη, αλλά επαναλαμβάνω, είναι επιτακτική ανάγκη να ε, ανταποκριθούμε άμεσα και αποτελεσματικά μέσω της κοινή γεωργικής πολιτικής, του Ταμείου Συνοχής και του Ταμείου Αλληλεγγύης. Θα πρέπει να ενεργοποιηθούν όλα τα κονδύλια από τους τρεις αυτούς προϋπολογισμούς. Σας ευχαριστώ. Και για να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση αυτή, το λόγο έχει ο Αντιπρόεδρος Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μάρος Σεφτσοβίτς. Συνάδελφοι, Σα παρακαλώ, αφήστε μα να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Και είναι χαρά μου να μπορώ να απαντήσω σε αυτέ τι πολύ έντονε συναισθηματικές παρεμβάσει των συναδέλφων, των προβουλευτών, ιδιαίτερα των Ισπανών για την ζημιέ που προκλήθηκαν, την καταστροφή που προκλήθηκε από την καταιγίδα Γκλώρια. Γιατί νομίζω ότι αυτή η καταστροφή μα δεν είναι ένα πρέτερο παράδειγμα κλιματική αλλαγή, η οποία δεν είναι δυνατόν να συνεχίσουμε να την αγνοούμε. Γιατί έχει καταστεί κατεπίγουσα ανάγκη και συμφωνώ με την κυρία Μοντσεράτ λοιπόν, η οποία είπε ότι θα πρέπει να δράσουμε και να ενεργήσουμε γρήγορα, με ευελιξία και ταχύτητα. Να σα εξασφαλ... να διαβεβαιώσω κύριε Πρόεδρε και αγαπητοί βουλευτέ ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προσαρμόσει το πρόγραμμα εργασία τη και την ταχύτητα δρασή για να προσαρμοστεί στι προκλήσει των επόμενων ετών. Και θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι κατανοώ πολύ καλά αυτό που είπε η Λαμαρό ότι σε ό,τι αφορά την έκταση της καταστροφής αυτής, σε ό,τι αφορά και την τοπική οικονομία, κατανοούμε τις δραματικές συνέπειες. Να ευχαριστήσω τον κύριο Γκοντζάλες Πόντς για την πολύ γλαφυρή εικόνα που μας έδωσε ότι δεν πρόκειται για μια-δυο φυσικέ καταστροφέ, αλλά μια σειρά φυσικών καταστροφών που μπορούν να καταστρέψουν ολόκληρε περιοχέ. Και να σα εξασφα... σας διαβεβαιώσω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι δεσμευμένη για να βοηθήσει την Ισπανία και τα άλλα κράτη-μέλη αν πληχθούν από φυσικέ καταστροφέ με όποιο τρόπο δυνατό. Αυτό που έχω να πω μόνο είναι ότι όλοι θα πρέπει να δράσουμε και να αντιδράμε πιο γρήγορα γιατί ξέρουμε ότι χρειάζεται πρώτα σωστή εφαρμογή τη σχετική νομοθεσία για να μπορέσουμε να δράσουμε γρήγορα, για να κινητοποιηθούν τα απαραίτητα κονδύλια. Και να σα ε, πω ότι δεν θα καθυστερήσουμε και δεν καθυστερήσαμε ούτε μία μέρα η κινητοποίηση όμως των πόρων χρειάζεται την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και άρα παίρνει χρόνο. Γι' αυτό λοιπόν κινητοποιήσαμε μόνο τις προκαταρκτικέ αυτέ πληρωμέ για την καταστροφή Ντάνα και περιμένουμε την αίτηση τη Ισπανική κυβέρνηση για την καταστροφή που έφερε η καταιγίδα Γλώρια! Το Ταμείο Αλληλεγγύης, να πω, ωστόσο, δεν είναι το μοναδικό εργαλείο που έχουμε. Τα CAP, η CAP και τα διορθωτικά ταμεία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την αντιμετώπιση τέτοιων φυσικών καταστροφών. Αυτό λοιπόν ίσω είναι μια συζήτηση για το μέλλον. Τι μπορούμε να κάνουμε από κοινού για να εξασφαλίσουμε την πιο γρήγορη κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύη και ποια άλλα μέσα και εργαλεία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να βοηθήσουμε τον κόσμο που βρίσκεται σε τέτοιε καταστροφέ. Τέτοιε καταστροφέ, οι οποίε δυστυχώ θα τι βλέπουμε όλο και πιο συχνά λόγω τη κλιματική αλλαγή. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κύριε Αντιπρόεδρε και με αυτή την παρέμβαση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ολοκληρώσαμε τη συζήτηση και θα περάσουμε στις ψηφοφορίες. Καλημέρα. morning, Καλημέρα συνάδελφοι και τώρα να ψηφίσουμε και βλέπω ότι έχουμε έτοιμα από τον κύριο Τζομπασκή να πάρει το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι. Είμαι αντίθετο στην απόφαση που έλαβε ο πρόεδρος ο κύριος Σασόλη για το άρθρο 13 του κανονισμού το οποίο προβλέπει ότι τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πρέπει να τηρούν την τάξη στην αίθουσα της Ολομέλειας δεν μπορούν να φέρουν πινακίδες ε, ε, σημαίες, εθνικές σημαίες αλλά οι εθνικές σημαίες δεν είναι οποιοδήποτε σύμβολα είναι ένα εθνικό σύμβολο είναι η εθνική μου σημαία δεν είναι ένα οποιοδήποτε πόστερ δεν μπορούμε να απαγορέψουμε λοιπόν τις εθνικές σημαίε. Σε κάποιες περιπτώσεις επιτρέπεται στους συναδέλφου να υψώνουν εδώ σύμβολα τα οποία είναι διαφιλονικούμενα. Γι' αυτό λοιπόν επιμένω η διάσκεψη των Πρόεδρων να ανακαλέσει την απόφαση αυτή που έλαβε ο προεδρό. Γιατί εγώ θα βάλω την σημαία μου εδώ μπροστά, αν θέλει κάποιο να την αφαιρέσει, να το κάνει για τη βία. Κύριε Τζαμπάσκη, δεν πρόκειται να ξεκινήσετε αυτή τη στιγμή η συζήτηση για το θέμα αυτό, αλλά θα ήθελα να διαβάσετε τον κανονισμό με προσοχή και κυρίως το άρθρο 13, όπου αναφέρεται με σαφήνεια ότι τα μέλη, οι βουλευτές δεν θα φέρουν οποιαδήποτε τέτοια πινακίδα και φυσικά έχουν γενικά την υποχρέωση να σέβονται την αξιοπρέπεια της Ολομέλειας. Γι' αυτό λοιπόν, γι αυτό, λοιπόν ο Πρόεδρος αποφάσισε να ακολουθηθούν έτσι οι κανόνε. Κύριε Τζαμπάσκι, θα σας αναφέρω στον ε, Πρόεδρο, θα αναφέρω το θέμα σας, αλλά δεν θα το συζητήσουμε τώρα. Διαδικαστικό από την κυρία Ιντφέλντ. Σας παρακαλώ να σεβαστείτε την Ολομέλεια, αδελφή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε και να ζητήσω την προσοχή για λίγα δεύτερα για ένα θέμα το οποίο επίσης σχετίζεται με την κοινοβουλευτική δημοκρατία και στι σχέσει ε, ε, μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ρωσίας. Γιατί προχθές πληροφορηθήκαμε ότι ένας ε, Ολλανδός βουλευτής ο οποίος επικρίνει ιδιαίτερω το ρωσικό καθεστώς μία από τις βασικές δυνάμεις από τον νόμο Μακνίξη, μπήκε στη μαύρη λίστα και το απαγορεύτηκε να μπει στη χώρα, όπως και κάποια μέλη εδώ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και προτείνω να επιδείξουμε αλληλεγγύη από την πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να έρθουμε σε επαφή με τον κύριο Μπορέλ και να ζητήσουμε την παρέμβασή του στις ε, ρωσικές αρχές. Θα δώσω το μήνυμα λοιπόν αυτό, κυρία Εντφέλτ, στον Πρόεδρο. Και άλλο ένα διαδικαστικό από τον κύριο Λάγκο Uh, uh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ένα διαδικαστικό σύμφωνα 195 του κανονισμού για την 181 ε, παραβίαση του άρθρου 181 από τον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου. Πρόεδρε, ο Πρόεδρο του Κοινοβουλίου θεώρησε ότι όλε οι τροπολογίε μα για την έκθεση τη ε, της Επιτροπής ε, Τζούρι μη παραδεκτέ. Τι είναι μη παραδεκτό για το γεγονός ότι θα πρέπει η εθνική νομοθεσία για τις εκλογές να ερμηνεύεται σύμφωνα με το κοινωτικό δίκαιο. Τι είναι μη παραδεκτό ότι οι κοινοβουλευτικές διαδικασίες θα πρέπει να εξετάζονται σε σχέση με το Κοινοβούλιο. Τίποτε εδώ δεν είναι μη παραδεκτό. Μπορεί να μην συμφωνεί επί τη ουσία ο πρόεδρος, αλλά δεν επαφείται σε αυτό να αποφασίσει και να αποφανθεί επί τη ουσία. Εμείς αποφασίζουμε. Η πλειοψηφία του Κοινοβουλίου αποφασίζει επ' αυτόν. Το μόνο που κλήθησε να αποφασίσει είναι την παραδεκτότητα του αιτήματο. Η τροπολογία δεν ανέφερε ούτε ονόματα, ούτε άλλε πληροφορίε εκτό ε, πεδίο εφαρμογή. Η απόφαση αυτή θεωρώ ότι ακολουθεί την οδό της πολιτικής διαμόρφωσης των αποφάσεων που λαμβάνονται στο Κοινοβούλιο και κυρίως του κ. Γιουνκέρεως, ο οποίος και πάλι ε, ξεπέρασε τα, τις αρμοδιότητές του. Δεν είναι βασιλιάς. Είμαστε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν είμαστε σε συνταγματική μοναρχία. Ας αφήσουμε λοιπόν το Κοινοβούλιο εμάς να αποφασίσουμε από αυτών των θεμάτων. Συνάδελφοι, θα ήθελα να πω ότι βάσει των κανόνα και του εσωτερικού κανονισμού που οφείλουμε όλοι να σεβαστούμε, η απόφαση περί μη παραδεκτού ή παραδεκτού είναι ε, αρμοδιότητα του Προέδρου. Και περνάμε στις ψηφοφορίες. Διαδικαστικό? Όχι, οπότε δεν θα το δεχτώ. Δεν είναι θέμα μπλε κάρτας. Περνάμε στις ψηφοφορίες. Χρονοδιάγραμμα των περιόδων συνόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το 2021. Is point of order? Είναι όντως διαδικαστικό. Καλώς, έχετε το λόγο. Για τις σημαίες. Συγγνώμη, συγγνώμη, συγγνώμη. Δεν θα γίνει συζήτηση για τις σημαίες. Μόνο διαδικαστικό θα δεχτώ. Χθες ήταν απόφαση του Προέδρου, θα παραπέμψω το ζήτημα στον Πρόεδρο και ίσως χρειαστεί κάποια ζήτηση. Ναι, αλλά θέλω να αναφερθώ σε κάτι που έγινε χθε λέει. Όχι, Κάποιο κατέβασε σημαία χθε. Συγγνώμη, αλλά το θέμα σα δεν είναι διαδικαστικό. Διαδικαστικό υπάρχει. Παρακαλώ. Αφορά ένα διαδικαστικό ζήτημα. Η αντιπροσωπεία του κόμματό μα, που ήταν η μεγαλύτερη μετά τι εκλογέ, εκπροσωπεί περίπου 5,4 εκατομμύρια πολίτε. Δυστυχώ υπάρχουν διακοπέ στο μικρόφωνο του. Συγγνώμη, δεν ήταν διαδικαστικό ούτε το δικό σας. Περνάμε στις ψηφοφορίες. Ψηφίζουμε για το χρονοδιάγραμμα των περιόδων συνόδου του Κοινοβουλίου για το 2021. Έχω λάβει δύο τροπολογίε. Ψηφίζουμε την τροπολογία 2, διανατάσσεως τη χειρό. Ποιο είναι υπέρ, παρακαλώ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε την τροπολογία 1 με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. The vote is closed. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Η πρόταση της ε, διάσκεψης των Προέδρων που ε, ανακοινώθηκε στις 16 Ιανουαρίου έχει εγκριθεί μετά την τροποποίηση. Χρονοδιάγραμμα τώρα των περίοδων Συνόδου του Κοινοβουλίου για το 2022. Δεν έχω λάβει τροπολογίε για το χρονοδιάγραμμα των περίοδων Συνόδου του Κοινοβουλίου του 2022, οπότε η ανακοινωθή σα 16 Ιανουαρίου πρόταση τη διάσκεψη των Προέδρων εγκρίνεται χωρί αλλαγέ. Και περνάμε στον έλεγχο τη εντολή, έκθεση Νετσίνγκα. Ψηφίζουμε την παράγραφο 3, πρώτο τμήμα, διανατάσσεως της χειρός. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα ποιος είναι υπέρ κατά αποχές θα πρότεινα να κάνουμε έναν ηλεκτρονικό έλεγχο άρχεται η ψηφοφορία τέλος ψηφοφορίας εγκρίνεται ψηφίσουμε την παράγραφο 6 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα. Διανατάσσεω της χειρός. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Αιτιολογική ε, σκέψη L. Αρχικό κείμενο. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές θα κάνουμε και πάλι ηλεκτρονική επαλήθευση. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία για την έκθεση Νετσίγκα με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. εγκρίνεται και συγχαρητήρια στην εισηγήτρια. Περνάμε σε εκθέσει την άλλη. Κάποιο ζήτησε το λόγο ή όχι. Η κυρία Ρίκνερ. Ρέγνερ. Έχετε το λόγο. Can we open the micro for three... Να ανοίξει το μικρόφωνο. Come on. Was ist denn jetzt hier? Nein, warum hinten unser Tisch? Hier, was Olga, nein, geht, ruf sie mal zu dir. Dein mal aus. Hier ist Na, geht doch nicht. Yes, does it work? Have you found any? Λειτουργεί το μικρόφωνο. Ναι, εδώ βρίσκομαι. Πολύ ωραία. Τέλεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνετε το λόγο πριν την ψηφοφορία αυτή και θα ήθελα να επενθυμίσω σε όλους όσοι ψηφίζουν το ψήφισμα για την ε, ισότητα των οφείλων στα θεσμικά οργανά το Μάρτιο του 2019 το ψήφισμά μας το οποίο αναφέρει ότι θα πρέπει να υπάρχει η ισότητα των φύλων στις ε, ψηφοφορίες. Ε, όλοι οι υποψήφοι εδώ είναι άνδρες. Σας υπενθυμίζω λοιπόν το ψήφισμα αυτό. Ευχαριστώ και θα συνεχίσουμε λοιπόν την ψηφοφορία. Πρώτη έκθεση της κυρία Δινάρη για τον διορισμό του Πατρό Ματσιάρο με μυστική ψηφοφορία. The vote is closed. Πέρασε. Εγκρίθηκε δεύτερη έκθεση την άλλη για την ε, δορισμό του Τινοχείου του Σαουρίνα και πάλι με πιστική ψηφοφορία. Έναρξη ψηφοφορία. The vote is closed. Πέρασε. Εγκρίθηκε. Επόμενη έκθεση την άλλη για τον διορισμό του Γιάνντε Καρπεντιέ και πάλι με μυστική ψηφοφορία. Έναρξη παρακαλώ ψηφοφορία. The vote is closed. Πέρασε. And it has been... Εγκρίθηκε. Επόμενη έκταση την άλλη για το διορισμό του Τζέρι Κρός. Μυστική ψηφοφορία και πάλι. Έναρξη. The vote is closed. Πέρας. And it has been rejected. Απορρίφθηκε. Και περνάμε στο επόμενο θέμα σε ό,τι αφορά τις ενστάσεις στο σημείο 113 για το του τιτανίου και το σύνολο του ψηφίσματος με ανάταση του χειρόσπου. Υπέρ. Κατά. Απόχες. Απορρίφθηκε. Αν θέλετε μπορούμε να κάνουμε ηλεκτρονικό έλεγχο, αν και το αποτέλεσμα ήταν ξεκάθαρο. Έναρξη ψηφοφορία. The vote is closed. Πέρας. Απορρίφθηκε με μεγάλη διαφορά. Και περνάμε λοιπόν στο επόμενο θέμα. Κοινό φορτιστή για κινητό ραδιοεξοπλισμό. Ετλική σκέψη Α υπέρ κατά απόχες εγκρίνεται εντελογική σκέψη β σε δύο τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ κατά απόχες εγκρίθηκε δεύτερο τμήμα υπέρ κατά απόχες εγκρίθηκε τροπολογία 1 με ονομαστική κλίση παρακαλώ έναρξη πέρας Απορρίφθηκε. Το ψήφισμα στο σύνολό του με ονομαστική κλίση. Έναρξη ψηφορία. Πέρα. Εγκρίθηκε. Και τώρα να περάσουμε στο επόμενο σημείο για το αμυστολογικό χάσμα. Πρόταση ψηφίσματος της ομάδος ECR Ψηφίζουμε το σύνολο του ψηφίσματος με ονομαστική κλίση, παρακαλώ. The vote is closed. Πέρας ψηφορίας. Απορρίφθηκε. Ψηφίζουμε λοιπόν το ψήφισμα των τεσσάρων πολιτικών ομάδων, τροπολογία 7, με ονομαστική κλίση, έναρξη. Πέρας. Απορρίπτεται. Ψηφίζουμε τώρα την παράγραφο 2 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα, διαντάσταση της χειρός, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ζητείτε έλεγχος για το δεύτερο τμήμα. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά παρακαλώ. Πέρας. Εγκρίθηκε. Ψηφίζουμε τώρα την τροπολογία Α με ονομαστική κλίση. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 9. Με ονομαστική κλίση παρακαλώ. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία υπαριθμών 1. Πρώτο τμήμα με ονομαστική κλίση. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα με ονομαστική κλίση. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. Τρίτο τμήμα. Με ονομαστική κλίση ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. Τέταρτο τμήμα. Με ονομαστική κλίση πάλι. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. Το αρχικό λοιπόν κείμενο καταπίπτει και περνάμε στην τροπολογία 2 με ονομαστική κλίση. Ψηφίζουμε. The vote is closed. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Six and two parts. Παράγραφος 6 σε δύο τμήματα. Το πρώτο τμήμα διαμετάσσεως της χειρός. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται και αυτό. Παράγραφος 9, αρχικό κείμενο. Πρώτο τμήμα. Ποιος είναι υπέρ. Against. κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 10. Διανατάσσω της χειρός υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 11, πρώτο τμήμα. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Παράγραφος 13. Σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 12 με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. The vote is closed. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 13. Διανατάσσεως της χειρός. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία. The vote Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Περνάμε στην τροπολογία 14 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. The vote is closed. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 15. Πρώτο τμήμα με ονομαστική κλίση. Άρχεται ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα τώρα με ονομαστική κλίση. Άρχεται ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Ε, Διανατάσσεω χειρό τρία Τροπολογία κατά αποχέ. Απορρίπτεται. Τροπολογία 4. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 5. Με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 6. Διανατάσσεω της χειρός. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ψηφίζουμε το σύνολο του ψηφίσματος όπως έχει τροποποιηθεί με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας και εγκρίνεται. Μια και είναι η τελευταία μας ψηφοφορία παρουσία των Βρετανών συναδέλφων, θα ήθελα και εγώ να τους ευχαριστήσω για όλο το έργο τους ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να τους ευχηθώ καλή τύχη. Thank Σας ευχαριστώ. Ολοκληρώσαμε τις ψηφοφορίες. Δύο λεπτά διάλειμμα και θα συνεχίσουμε με τις αιτιολογήσεις ψήφου. Συνάδελφοι, παρακαλώ να περάσουμε στις αιτιολογήσεις ψήφου. Οπότε όσοι δεν θα λάβουν μέρος στη συζήτηση, στην παρουσίαση μάλλον των επεξηγήσεων ψήφου, παρακαλώ να εγκαταλείψουν την αίθουσα της Ολομελίας αθόρυβα για να περάσουμε στους ομιλητές. Περνάμε στις αιτιολογήσεις ψήφου. Πρώτα αυτές που μας απέμειναν από χθε, αλλά και μία ανακοίνωση. Η ομάδα Renew ανακοίνωσε τις εξή αλλαγές στους διορισμούς. Μπλατ Μάριος Πακός θα αντικαθεστεί στον Σαφάτ Μοχαμέτ στην ε, Επιτροπή Πολιτισμού και Εκπαίδευσης με ισχύ από την ημέρα της ανακοίνωσης. Παρακαλώ και πάλι συνάδελφοι όσοι δεν θα έχουν επεξηγήσει ψήφου να φύγουν από την αίθουσα θόρυβα για να μπορούμε οι υπόλοιποι να συνεχίσουμε. Οπότε αρχίζουμε με την επεξήγηση ψήφων. Ε, η επεξήγηση που δεν έγιναν χθε και μετά θα συνεχίσουμε με τα όσα ψήφισαμε σήμερα. Έχουμε πάρα πολλά αιτήματα για επεξηγήσεις ψήφου. Αλλά Μέχρι τις μισή μόνο μπορούμε να συνεδριάσουμε. Οπότε όποιοι δεν προλάβουν θα υποβάλουν τις επεξηγήσεις τους εγγράφους. Η πρώτη συνάδελφος που έχει ζητήσει τον λόγο είναι η κυρία Σόντροβα. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πρόεδρε που μου δίνετε τον λόγο. Χθε κάναμε την ψηφοφορία για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου και της Βορείου Ιρλανδίας. Ήταν για μένα η πιο δύσκολη ψηφοφορία της θητείας μου. Εγώ κατά της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου. Παρ' όλα αυτά ψήφισα υπέρ της συμφωνίας διότι θεωρώ ότι θα πρέπει η αποχώρηση να γίνει επί τη βάση συμφωνίας και θα πρέπει έφτακτα να ρυθμιστεί το καθεστώς που διέπει τους Βρετανούς στην Ευρώπη και Ευρωπαίους στην Βρετανία και να υπάρχει αγαστή συνεργασία μεταξύ των δύο πλευρών στο μέλλον. Γι' αυτό και ψήφισα υπέρ της συμφωνίας. Πάντως είμαι πάρα πολύ στεναχωρημένη για αυτήν την αποχώρηση. Δεν νομίζω ότι ήταν κάτι απαραίτητο αυτό το οποίο... Κυρία έχετε το λόγο τώρα. Σήμερα Έχουμε εκατοντάδες χιλιάδων πολιτών του Ηνωμένου Βασιλείου που είναι στεναχωρημένοι γιατί έχασαν την ευρωπαϊκή ηθαγένεια. Παρακαλώ να είσαστε γενναιόδοροι μαζί μας, να είστε μεγαλόψυχοι. Να μην ε, μας φερθείτε όπως σας φέρθηκαν αυτοί που θέλουν το Brexit. Τα πρώτα θύματα του λαϊκισμού είμαστε εμείς, ας είμαστε τα μόνα θύματα. Δεν ήθελα αυτή την επονίδιστη συμφωνία, βέβαια σε καλύτερη θέση είναι η Ένωση παρά το Ηνωμένο Βασίλειο. Δεν το καταλαβαίνει όμως αυτό ο κόσμος στην ε, χώρα μου. Σας ευχαριστούμε για την ευγενική σας ε, συμπεριφορά. Αντίο. Next Επομένη, η κυρία Γκίμπσον. Ένα λεπτό. Ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο σήμερα. Ε, εκφράζω εκατομμύρια συμπολιτών μου και είμαι πάρα πολύ στεναχωρημένη. Ε, αισθάνομαι πάρα πολύ μεγάλη απώλεια δικαιώματα, ελευθερίες, την ευρωπαϊκή μου ηθαγένεια, ένα τμήμα της ταυτότητάς μου που θεωρώ ότι είναι πολύτιμη. Στα βάθη της καρδιάς μου ξέρω ότι το Brexit είναι λάθος και δεν νομίζω ότι ποτέ θα μπορέσω να συγχωρήσω αυτούς τους εγωιστές ε, πολιτικούς που μας οδήγησαν εδώ. Ε, είμαστε σπουδαίο έθνο, αλλά είμαστε πιο σπουδαίοι όταν είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, είμαι πάρα πολύ απογοητευμένη. For one minute, Για ένα λεπτό το λόγο έχει ο κύριος η κυρία Πρόφη. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Χθε εδώ στο συνέδριο τη Ελεομέλεια, μαζί με του φιλελεύθερου Δημοκράτε. καταψήφισε αυτή την συμφωνία για τον Brexit και αυτό γιατί πιστεύω ότι αυτή η συμφωνία απόσυρση αποχώρηση αποτελεί κακή συμφωνία για την Ηνωμένο Βασίλειο. Δεν υπάρχει καμία συμφωνία που να είναι καλή για το Ηνωμένο Βασίλειο παρά μόνο παραμονή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι επόμενοι μήνε μα επιφυλάσσουν ανασφάλεια όχι μόνο για του πολίτε μα, αλλά και για του Βρετανού που μένουν στην Ευρώπη και για του πολίτε τη Ευρωπαϊκή Ένωση που μένουν στην Ηνωμένο ε, Βασίλειο και Είμαι πραγματικά πολύ καταπογοτευμένη από τον Μπόριση Τζόνσον και για το γεγονός ότι δεν αγωνίστηκε γι' αυτό η διαπραγματευτική ομάδα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ελπίζω στου επόμενου μήνες να μας υποστηρίξετε, να μην υποκύψετε στις πίεσεις του Μπόρι Τζόνσον. Θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε στενά ω γείτονε για να καταπολεμήσουμε την αλλαγή του κλίματος και για να αντιτηρηθεί σε δύσκολες εποχές η ειρήνη στον κόσμο. Ελπίζουμε να παραμείνουμε στενοί φίλοι και σύμμαχοι και μία μέρα να επιστρέψουμε. Thank you, Mr. Ευχαριστώ. Ο κύριος Πάταν για ένα λεπτό. Είμαι περήφανος που ψήφισα υπέρ τη ε, συμφωνία αποχώρηση και που εκπλήρωσα τη δημοκρατική εντολή του Βρετανικού λαού να βγούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Συμφωνία είναι βέβαια πολύ ατελή, αλλά ε, ο, Πρωθυπουργό του Τζόνσον υποσχέθηκε ε, ποικιλία σε ό,τι αφορά πολλά ζητήματα. Ο κύριο Φερχόφστατ πήρε το λόγο χθε και επιβεβαίωσε την απόφασή μου ότι η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου ήταν Σωστή. Είπε ότι ο λόγος για τον οποίο αποχωρεί η Μεγάλη Βρετανία είναι ότι είχε πολλές ελευθερίες. Ήθελε εκχώρηση λοιπόν κυριαρχία. Αυτό δεν είναι το μάθημα όμως που διδαχθήκαμε από τον Ηνωμένο Βασίλειο. Θέλουμε να αποστασιοποιηθούμε από ένα τέτοιο υπερκράτο, γιατί οποιαδήποτε τέτοια απόπειρα μακρινή από τους πολίτες πάντα θα καταλήξει σε αποτυχία. Επόμενο ομιλητή, η κυρία Ward. Ευχαριστώ. Ήταν ε, προνόμιο και χαρά να υπηρετώ από το 2014 την, ε, τη Βόρεια Ανατολική Εκλογική Περιφέρεια της Αγγλίας συμμετείχα σε πολλά προγράμματα, ε, την δράση που έγινε μετά Erasmus και που έφερε κοντά τους νέους ξεπερνώντας τα σύνορα. Εγώ ψήφισα κατά της συμφωνίας αποχώρησης γιατί δεν μπορώ καλή την πίστη να επικυρώσω μια συμφωνία που θα καταστρέψει την οικονομία, θα αποδυναμώσει τα δικαιώματα των πολιτών και την κοινωνική προστασία, θα περιορίσει τις ε, ευκαιρίες και δυνατότητες των νέων, θα απειλήσει την ασφάλεια, τη σταθερότητα και την ειρήνη και θα καταστρέψει την διεθνή φήμη του Ηνωμένου Βασιλείου πολλοί θα πούν ότι είναι ώρα να το αποδεχτούμε. Εγώ πιστεύω ότι είναι η ώρα να πούμε την αλήθεια και να ζητήσουμε λογοδοσία. Και δεν είναι θέμα ότι θα χάσω εγώ τη δουλειά μου ως Ευρωβουλευτής. Χιλιάδες θέσεις απασχόλησης θα απειληθούν και πολλές οικογένειες και κοινότητες θα επηρεαστούν και περισσότερο σε περιθωριοποιημένες κοινότητες αστερημένες ενώ η κυβέρνηση στο Westminster κοφεύει και μας αγνοεί. Σας ευχαριστώ. Επόμενη ομιλήτρια, η κυρία Ντελούση για ένα λεπτό. Δεν ήταν εύκολο να ψηφίσουμε υπέρ της ε, συμφωνίας αποχώρησης χθες, αλλά ε, ο Μπόρις έκανε χάρη και στις δικές μας πιέσεις τροπολογίες και είπε ότι δεν θα υπάρξει καμία παράταση μετά το 2020 και θα υπάρχουν συνθήκες ισότιμου ανταγωνισμού. Και έτσι έδωσε στη στρατηγική του Brexit μια δημοκρατική εντολή που θα πρέπει το κόμμα του Brexit να τη σεβαστεί. Ελπίζουμε να τηρήσει υποσχέσει τον Μπόρι Τζόνσον. Θα το περιμένουμε πάντω. Και αυτή, αυτό το όμορφο δημοκρατικό κίνημα που ανθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο θα είναι έμπνευση και σε εκείνου που πιστεύουν ότι ε, η δημοκρατία μερικέ φορέ κινδυνεύει. Γιατί θα πρέπει να βρούμε την ασφαλιστική δικλίδα μεταξύ του κόσμου και των εξουσιών που μας εκχωρεί. Ε, ειρηνικά διαδήλωσαν εκατομμύρια πολίτες όταν θεώρησαν ότι αγνοείται η ψήφο του. Και αποδείξαμε σε όλο τον κόσμο ότι μπορούμε να επιτύχουμε ειρηνική αλλαγή μέσω του εκλογικού αποτελέσματος και κατεβαίνοντα κάλπε. Η κυρία Φόξ για ένα λεπτό. Ο κύριος... Κυρία Φόξ, συγγνώμη. Εγώ ψήφισα υπέρ μετά το μήνυμα πολλών ψηφοφόρων από το Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτό δεν είναι αντίο αλλά εις το επανειδήν. Όχι γιατί θα επιστρέψουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά γιατί θα σας ξαναδούμε πολύ σύντομα ως φίλοι και ίσοι, ισότιμοι, όπως κάθε κράτος μέλος που εκπροσωπείται εδώ. Δεν χρειαζόμαστε την Ευρωπαϊκή Ένωση να διαχειριστεί τις φιλίες και τη συνεργασία μας, Ευρωπαίοι συνάδελφοι. Θα κρατήσουμε επαφές. Εγώ είμαι υπερήφανη Ευρωπαία. Ε, αγαπώ την Ευρώπη, όχι την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά ανάγκη είδα ότι το καλύτερο τρόπο για να υπερασπιστούν τα δικαιώματα των πολιτών είναι η παρακαταθήκη του Ρουσό, του Διαφωτιστών, ε, ε, η Ευρώπη των Εθνών Κρατών. Θέλουμε τον ύμνο της ελευθερίας και όχι τον ευρωπαϊκό ύμνο. Και ευχαριστώ όσους ήταν ανοιχτόμυαλοι και την ανεβήκον ε, για τη δημοκρατία και την ελευθερία. Καλή τύχη λοιπόν, εις το επανειδήν και θα κρατήσουμε την επαφή μας. Ο κύριος, ο κύριος ένα λεπτό, υπερψήφισα την συμφωνία και ο λόγος είναι ότι χρειάζεται έφτακτη αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να το διευκολύνω. Εψήφισα αυτήν την συμφωνία που θα διαμορφώσει τις μέλους σχέσεις μας με τις δύο πραγματεύσεις αλλιώς θα είχαμε ένα άτακτο Brexit με πάρα πολύ σκληρές συνέπειες και για τα δύο μέρη και την Βόρεια Ιρλανδία που με αφορά δεν θέλουμε ε, αδιαπέραστα σύνορα αλλά θα πρέπει τώρα να τολμήσουμε να προστατεύσουμε τα δικαιώματα του κόσμου αλλιώς αυτά πρόκειται να καταπατηθούν και να ακυρωθούν λίγο λίγο οι Ιρλανδοί που θέλουν να παραμείνουν Ευρωπαίοι που ζουν στην Ιρλανδία να έχουν ε, κατοχυρωμένα τα δικαιώματά τους και αυτό θα γίνει μόνο εάν εξασφαλίσουμε το να συνεχίσουν να ισχύουν τα όσο προβλέπει η συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής για τις ε, σχέσεις Ένωσης Ηνωμένου Βασιλείου. Ευχαριστούμε. Χουκ, ένα λεπτό. Σα ευχαριστούμε και για τον ύμνο και για την συμπεριφορά σας. Είναι κάτι που εντυπωσίασε ε, τον ε, λαό μας όταν ε, χάθηκε πλειοψηφία από την κυβέρνηση και ε, είχαμε κάποιον ηγέτη που συγκέντρωνε τη συνένεση όλου του πολιτικού φάσματος τότε ήταν μια ελπίδα να σταματήσει το Brexit αλλά δεν το καταφέραμε θα πρέπει τώρα οι προοδευτικοί να προσπαθήσουν να ξεπεράσουν τα λάθη και τους διχασμούς του παρελθόντος ο συμβασμός δεν είναι κάτι κακό έτσι βρίσκονται οι λύσεις ε, εάν φαγωνόμαστε μεταξύ μας δυναμώνει η αντίπαλή μας Επομένως δεν θα πρέπει να απογοητεύσουμε τους ε, νέους που θέλουμε στην Ευρώπη ε, και θα πρέπει να πέσει μέχρι το 24 ο Τζόνσον, να ξαναγίνουμε μεγάλο έθνος και θα πρέπει να προχωρήσουμε χέρι-χέρι όχι μόνο ε, όπως κάναμε εδώ αλλά συνέχεια στο μέλλον. Κιουτσούκ, ένα λεπτό. Εγώ υπερψήφισα τη συμφωνία αποχώρησης. Όχι γιατί μου αρέσει, όχι γιατί θεωρώ ότι είναι τέλεια, αλλά γιατί δεν υπάρχει άλλη λύση. Αυτό που χρειάζεται πάνω απ' όλα είναι το εξής. Ρεαλιστική συνεννόηση που θα διαμορφώσει τις μέλουσες σχέσεις των δύο μερών. Εύτακτο να είναι το Brexit. Επίσης, πρέπει να συνεχιστεί ο δημιουργικός διάλογος και να έχουμε πάντα στο μυαλό μας τη σχέση Ένωσης Βρετανίας το ζήτημα είναι μπορούμε να έχουμε μια σφαιρική ολοκληρωμένη σχέση με τη Βρετανία όταν έχουμε μόνο 11 μήνες για να ολοκληρώσουμε τις διαπραγματεύσεις εγώ θεωρώ ότι δεν μπορούμε να τα καταφέρουμε έτσι και με προβληματίζει το εξή. Θα συζητήσουμε για ασφάλεια, περιβάλλον, οικονομικές σχέσεις, αλλά τι θα γίνει με τα δικαιώματα του κόσμου, Ευρωπαϊκής Ένωσης, Βρετανών, και αυτό θα πρέπει να μπει στο θεματολόγιο. Πολύ σημαντικό και εγώ προ τα εκεί θα προσπαθήσω. Ευχαριστώ. Ο κ. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν πραγματικά θλιβερή η χθεσινή ημέρα όταν εγκρίθηκε η Συμφωνία αποχώρηση από το Κοινοβούλιο εδώ. Εγκρίθηκε με μεγάλη πλειοψηφία και δυστυχώ θα φύγουμε αύριο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά θα το κάνουμε χωρίς την υποστήριξή μου γιατί δεν μπόρεσα να υποστηρίξω και να υπερψηφίσω αυτή τη συμφωνία χτες. Αποδέχομαι τα γεγονότα όπω εξελίσσονται. Αποδέχομαι το γεγονός ότι πλέον αποχωρούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά αν μπορώ να το δεχτώ αυτό, αυτοί οι οποίοι η συντηρητική, το κόμμα του Brexit και όλοι οι υπόλοιποι θα πρέπει να αποδεχτούν την ευθύνη για αυτά που θα ακολουθήσουν από εδώ και πέρα. Και πιστεύω ειλικρινά και ελπίζω ότι μπορούμε να χαράξουμε έναν δρόμο που θα κάνει όλη αυτή τη δουλειά για τη χώρα μας, υπέρ της χώρας μας, αλλά πολύ φοβάμαι ότι αυτό είναι κάτι το αδύνατο. Ευχαριστώ. Για ένα λεπτό, κύριε Σκοβούτ. Η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου είναι κάτι το πολύ θλιβερό ό,τι αφορά την ε, ολοκλήρωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ήταν πολύ χρήσιμο και ωφέλιμο ε, μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρά το γεγονός ότι έγινε η εκστρατεία, δημιουργήθηκαν πολλές ψεύδεις ειδήσει οι οποίες και κυκλοφόρησαν. Ο λαός της Βρετανίας αποφάσισε τώρα να στραφούμε προς το μέλλον και είμαι βέβαιος ε, ως Ευρωπαίος από τη θα πρέπει στο μέλλον είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπορούμε να αποτύχουμε και να δώσουμε και στους Ουαλούς και στους Σκοτσέζους και στους Ιρλανδούς και στους Άγγλους την ε, υπόσχεση ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναχτές τις αγκαλιές στην αγκαλιά της. Ε, δεν θα είστε ποτέ μακριά μας. Thank Σας ευχαριστώ. Επόμενη ομιλήτρια κυρία Ραφαέλα για ένα λεπτό. Βρετανοί φίλοι. Χτες αντιμετώπισα μια πραγματικά αδύνατη επιλογή και στο τέλος αποφάσισα να υπερψηφίσω για την, τα δικαιώματα του Βρετανικού λαού. Κανείς δεν κερδίζει από το Brexit και εδώ στο Κοινοβούλιο χάνουμε και αγαπητούς φίλους και πολύτιμους συναδέλφους. Θα χάσω τον γειτονά μου εδώ, Τι γειτονισά μου εδώ στο Κοινοβούλιο. Λουίζα, φτάσαμε και δύο μαζί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και με φιλοδοξίες και ακόμα είχα την ελπίδα να αποτρέψω το Brexit. Ήταν μεγάλη μου τιμή να κάθομαι δίπλα σου και στις συνεδριάσεις της Επιτροπής και εδώ στην Ολομέλεια και πάνω απ' όλα έχεις γίνει και στενή μου φίλη. Το Brexit μπορεί να αρθώσει πολλά εμπόδια, αλλά αυτό δεν θα μπει στη μέση της φιλίας μας. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, ευχαριστώ και όλους τους Βρετανούς συναδέλφους και προσβλέπω την ημέρα που θα είσαστε και πάλι ανάμεσά μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Λεμπρετών για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, Ελάχιστε ψηφοφορίε είναι ιστορικέ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έγινε όμω μια τέτοια στι 29 Ιανουαρίου για να επικυρωθεί η συμφωνία του Brexit και είμαι υπερήφανο που ψήφισα υπέρ τη συμφωνία περί αποχώρηση θα έπρεπε να γίνει αποδεκτό το Brexit, γιατί θα πρέπει, ε, οφείλαμε να σεβαστούμε την κυριαρχία του Βρετανικού λαού, του αξιοθαύμαστου του Βρετανικού λαού, που για, για έδειξε και πάλι την θρηλυκή του αντίσταση στην αντικσότητα. Τρει φορέ χρειάστηκε να ψηφίσουν για τον Brexit. Το 2016 πρώτα με δημοψήφισμα. Το Μάιο του 2019 δεύτερη φορά με μαζική υποστήριξη του Brexit Party. Και το Δεκέμβρη του 2019 τρίτη φορά δίνοντα τον Boris Johnson την κοινοβουλευτική πλειοψηφία που χρειαζόταν. Κάθε φορά ο Βρετανικό λαό αντέδρασε με αποφασιστικότητα στην φιλοευρωπαϊκή προπαγάνδα και κατέριψε τι παρελκυστικές τακτικές του Γιούνκερ, του Σκεφερχόφστατ. Μπράβο σας Βρετανοί συνάδελφοι και καλή επιτυχία στο επόμενο στάδιο, την εθνική σας ε, ιστορία. Σας ευχαριστώ κύριο Σμίλερ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ ψήφισα υπέρ της αποχώρησης ε, για να αποτρέψουμε το νομικό και δικαιικό χάος που θα επικρατούσε με ένα άτακτο Brexit. Θέλουμε να σεβαστούμε και να προστατεύσουμε τα θεμελιώδη δικαιώματα των Ευρωπαίων υπηκών που διαβιούν στην ε, ε, Μεγάλη Βρετανία. Η μεγαλύτερη τέτοια μειοψηφία είναι οι Πολωνοί συμπολίτε μου. Σίγουρα για όλου του υπέρμαχου τη ολοκλήρωση ήταν μια θλιβερή η χθεσινή στιγμή. Εγώ ψήφισα πάντω υπέρ τη αποχώρηση γιατί μα ε, υποχρεώνει να διαφυλάξουμε ε, και στην Μεγάλη Βρετανία την υπεροχή του ενωσιακού δικαίου στη μεταβατική περίοδο και το σεβασμό των αποφάσεων του ΔΕΚ και των βασικών υποχρεώσεων που απορρέουν από τη συνθήκη. Θα πρέπει τέτοια συνεργασία να έχουμε σε όλα τα κράτη-μέλη και όχι μόνο σε μια χώρα που αποχωρεί. Ας μην ξεχνούμε ότι αυτά τα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες είναι η πεμπτουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας ευχαριστώ Ο κύριος Χάναν για ένα λεπτό, αλλά δεν τον βλέπω στην αίθουσα. Και περνάμε στον κύριο Λόπες Αγγιλάρ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Χθες ε, είπαμε τον τελικό μας λόγο ε, για το Brexit. Είναι όμως και πέφτει η αυλαία. Όχι. Α, ακούσαμε τόσες πολλές ε, γλώσσες, τόσες πολλά σχόλια. εμείς μαζί με τους εργατικούς στο σοσιαλιστές ψηφίσαμε ευχαρίστως κατά του όχι, κατά της αποχώρησης. Και φυσικά δεν είναι εδώ το πέρας των διαπραγματεύσεων. Έχουμε πολλά εκκρεμή θέματα, θεμελιώδη δικαιώματα, ελευθερίες, ε, προστασία δεδομένων, διαχείριση συνόρων, άσυλο, ασφάλεια, δικαστική συνεργασία. Και για να τα διευθετήσουμε όλα αυτά θα πρέπει να αντλήσουμε δύο διδάγματα. Καταρχήν θα πρέπει να μείνουμε κοντά για να συνεχίσουμε τις διαπραγματεύσεις, να συνεργαστούμε για να καταπολεμήσουμε καλύτερα την παραπληροφόρηση, τα fake news, να κρατήσουμε σύσσωμη και συσπηρωμένη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θα μας λείψουν οι θορυβόδεις ε, υπέρμαχοι του Brexit. Αυτό που θα μας λείψει αυτό που θα μας λείψουν είναι οι αξιολάτρευτοι, πολύ αγαπημένοι μας Βρετανοί φίλοι. Αυτοί θα μας λείψουν. Σας ευχαριστώ που ήσασταν εδώ. Σας ευχαριστώ για την επιθυμία και τη βούλησή σας να επιστρέψετε. Ευχαριστώ. Εμείς σας ευχαριστούμε κύριε Λόπες Αγγιλάρ. Κυρία Γιώβεβα, η επόμενη ομιλήτρια. Ευχαριστώ πολύ. Μετά τρισήμιση χρόνια ε, αυτού του πολιτικού σύριαλ. Φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Βεβαίω και θα ήθελα να παραμείνει η Βρετανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά ψήφισα υπέρ τη συμφωνία γιατί καλύτερα να έχουμε αποχώρηση έφτακτη παρά χαοτική. Πάροντο. Θα έχουμε πολλές προκλήσεις ε, στην μεταβατική περίπου θα ακολουθήσει. Αύριο θα χάσουμε ένα μέλος της ευρωπαϊκής οικογένειας. Αυτό είναι δεδομένο και είναι δεδομένο ότι θα μας λείψουν. Καλά, όχι όλοι, κάποιοι εξ αυτών. Πάντως θα πρέπει να αντιλήσουμε συμπεράσματα από το πώς φτάσαμε στο Brexit να προβληματιστούμε για το πώς είναι τα πράγματα σήμερα, σε τι κατάσταση βρίσκεται η δημοκρατία μας και δεν θα πρέπει να έχουμε επανέλειψη τέτοιων φαινομένων στο μέλλον. Ελπίζω αντλήσαμε κάποια μαθήματα από αυτό και επίσης ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να κάνουμε όλε τι μεταρρυθμίσει που χρειάζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτω ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να βρίσκεται πιο κοντά στον κόσμο και να σταματήσει η παραπληροφόρηση και η χειραγώγηση. Σα ευχαριστώ. Ο επόμενο, ο κύριο Overgard Νίλσεν. Η χθεσινή ψηφοφορία για τη συμφωνία αποχώρηση με έφερε μπροστά σε ένα δύσκολο δίλημα. Όσο έχει η συμφωνία, είναι βελτίωση του αρχικού κειμένου. Αλλά εγώ δεν φανταζόμουν έτσι το Brexit. Έχουμε το θέμα του Ιρλανδέζικου συνόρου, τα σχετικά με τους ανήλικους πρόσφυγες ε, και όλα αυτά μόνο χαρά δεν μου έφεραν ε, σε σχέση με την υπόθεση. Παρ' όλα αυτά κατέβηκα στις εκλογές με δημοκρατικές αρχές και ήθελα να αποκατασταθεί η εθνική κυριαρχία στο Κοινοβούλιο ε, όπως ε, ο Τζόνσον αλλά δεν μπορούμε ούτε εγώ ούτε κανένας άλλος να ανατρέψουμε τη δημοκρατική ε, απόφαση του λαού του 2016 και δεν θέλω να πω ότι με παραμύθιασε, με έπεισε τέλο πάντων ο Πρωθυπουργό καθόλου. Συνεχίζω και έχω επιφυλάξει για τι ε, υποσχέσεις του Τζόνσον προ ε, αυτούς που θέλουμε να φύγουμε και ε, θα ήθελα να καλυφθεί όλο ο κόσμο και όχι μόνο η συντηρητική και νομίζω αυτά τα 7,5 εκατομμύρια ελπίζω ότι δεν θα τα απογοητεύσει ο Μπόρες το ΜΑΚ ένα λεπτό Συνάδελφοι, είναι πάρα πολύ μεγάλη στεναχώρια μας τώρα. Εγώ προέρχομαι από χώρα της Ανατολικής Ευρώπης και θεωρώ ότι είναι κρίμα που η τόσο ισχυρή ένωση ισχυρή και γιατί ήταν μέλος της ευρωπαϊκής οικογένειας τόσα χρόνια η Βρετανία μας βοήθησε να προσεγγίσουμε την Ευρώπη αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση και να γίνουμε και εμείς μέλη της Ευρωπαϊκής Οικογένειας. Οπότε ευχαριστώ όλους πολιτικούς και συνεργάτες τους από τη Βρετανία. Μας βοήθησαν να είμαστε όλοι μαζί μέλη της οικογένειας και γι' αυτό ψήφισα υπέρ της συμφωνίας αλλά ήταν δύσκολη επιλογή μου μια που γνωρίζω ότι είναι πάνω από 355 τα εκατομμύρια στην Ευρωπαϊκή Ένωση και επίσης πάρα πολλοί Ρουμάνοι στην Βρετανία. Άρα θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε να προστατεύσουμε αυτούς τους ανθρώπους. Ευχαριστώ κύριε Σικόρσκι. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Και ήθελα να εξηγήσω γιατί καταψήφισα τη συμφωνία αποχώρησης. Όχι επειδή δεν εκτιμώ το έργο του Μισελ Μπαρνιέ και της ομάδας του. Ήταν μόνο η μορφή, ήταν μοναδική μορφή η οποία ήταν δυνατή για τη συμφωνία αποχώρηση. Πιστεύω όμω το Brexit είναι κακή ιδέα. Και αυτό ήταν ο μοναδικό τρόπο με τον οποίο μπόρεσα να πιστοποιήσω αυτή την πεποίθησή μου. Ήταν κακή ιδέα. Αποτέλεσμα ε, χρόνων δυσφήμισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Βρετανικό τύπο και κακής ε, παρουσίασης ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της δηλίας των Βρετανών πολιτικών. Μία έκκληση μόνο προς τους πολιτικούς έχω να κάνω. Ό,τι και να συμβεί μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένου Βασιλείου, εσείς το ψηφίσατε, εσείς το ζητήσατε, μην μας κατηγορήσετε εμάς λοιπόν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η ε, κυρία Τόπτσον, η επόμενη ομιλητρία. Δεν τη βλέπω όμω στην αίθουσα. Η ε, κυρία Κούμπουλα να η επόμενη. Ευχαριστώ πρόεδρε. Και χθε καταψήφισα. Μάλλον ψήφισα αντίθετα με τις επιθυμίες μου και είμαι ιδιαίτερα λυπημένη για τους Βρετανούς που ήθελαν να παραμένουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Λυπάμαι ιδιαίτερα γιατί οι ψηφοφόροι μου ούτε αυτοί επιθυμούσαν το Brexit, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση εργάζεται για τους ανθρώπους, για να έχουμε ένα καλύτερο κόσμο, για να μπορούμε να ζούμε σε ένα ειρηνικό καθεστώς, το πρόγραμμα Εράσμους για τους φοιτητέ, η πολιτική για το κλίμα, η πολιτική για το περιβάλλον, η πολιτική για καλύτερη κινητικότητα, για αγωνικές άδειες, για να βελτιωθεί η ζωή των παιδιών εργαζόμαστε σε πάρα πολλού τομεί για να υπάρξει ευημερία για τον κόσμο και προσπαθούμε να δημιουργούμε έναν κόσμο πιο δίκαιο, πιο σωστό. Η μοίρα μας λοιπόν μας φέρνει μαζί. Γι' αυτό λοιπόν και στο μέλλον θα συνεχίσω να εργάζομαι και να θυμάμαι και τις δικές τους επιθυμίες και τις δικές τους ανάγκες. Σας ευχαριστώ πολύ, συνάδελφοι του Λέμπερ. Γεια σας. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Γουάλλας, για ένα λεπτό. Η Ιρλανδία θα ήθελε να παραμείνει το Ηνωμένο Βασίλειο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό η ψήφος του λαού τη μεγάλη Βρετανία το 2016 να γίνει σεβαστή. Ψηφίσαμε όχι στην Ίκαια και όχι στη Λισιβόνα. Ήταν ε, λάθο η απάντησή μα Ξανά έβαλαν να ψηφίσουμε. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα λοιπόν αυτό. Το αποτέλεσμα είναι ότι και οι Βρετανοί ψήφισαν κατά τον περασμένο μήνα και αν ο Τζέρι Κόρμπιν ε, που είναι αντιφιλελευθερίστης είχε προσπίσει τα δικαιώματα στην ίδια το κόμμα του, δεν θα είχαμε φτάσει εδώ. Γιατί οι Βρετανοί ήδη είχαν αποφανθεί, ήδη είχαν κάνει την επιλογή του και έκαναν την επιλογή του για δεύτερη φορά, είτε μα αρέσει είτε όχι. Καταλαβαίνουμε ε, και έχουμε μεγάλη συνέφεια με το λαό τη Μεγάλη Βρετανία. Δεν μα αρέσουν πάντα οι κυβερνήσει του, αλλά με το λαό δεν έχουμε τίποτα. Και θα θα μας λείψουν γιατί πραγματικά υπήρχαν ε, από κάποιοι εξαιρετικοί ομιλητέ από την ομάδα του Brexit και θα λείψουν. μας λείψουν. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Επόμενο ομιλητή. ο κύριο Λόπες Ιστορή Βάιτ. Κύριε Πρόεδρε, είμαι Ισπανός. Εκπροσωπώ την Ισπανία, μια χώρα που για αιώνες ολόκληρους είχε προβληματική, πολύ προβληματική σχέση και μόνιμες διαμάχες και μάχες ε, με το Ηνωμένο Βασίλειο. Τα τελευταία 40 χρόνια όμως μάθαμε να, τον αγγλοσεβασμό και την συνύπαρξη. Οι Ισπανοί ε, ανακάλυψαν και ένα άλλο Ηνωμένο Βασίλειο. Κρίμα που με τη δράση αυτών που θέλουν το τέλος αυτό που κατέστρεψαν την ενότητα της Ευρώπης, όχι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την ενότητα της Ευρώπης, μας έβαλαν όλους σε κίνδυνο. Θα πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους στο μέλλον, όπως είπε ένα συνάδελφος. Να μην το γλιτώσουν όπως έκανε ο Φαράς μετά το δημοψήφισμα, να μην δραπετεύσουν. θα επιστρέψουν οι εθνικισμοί, ε, το μίσος που προκάλεσαν αυτοί οι άνθρωποι εμείς στηρίζουμε τους φίλους μας, πραγματικούς Βρετανούς, τους γνήσους Βρετανούς που έχουν τον αγώνα και το θάρρος να ρέει στις φλέβες τους. Εμείς θα συνεχίσουμε παρόλα αυτά να συνεργαζόμαστε μαζί τους γιατί τους εκτιμούμε και ανακαλύψαμε την πραγματική σας ταυτότητα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την πραγματική σας ουσία. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Βρετσιονοβά για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Χθες και εγώ, όπως και πολλοί άλλοι συνάδελφοι στην Ολομέλεια, ψήφισα υπέρ της συμφωνίας ε, περί αποχώρησης. Λυπούμε για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, αλλά τουλάχιστον να φροντίσουμε οι μελλοντικέ μας σχέσεις να είναι όσο το δυνατό καλύτερες γίνεται. Και το Brexit θα πρέπει να το, να το αντιμετωπίσουμε ως προειδοποίηση. Ε, χτύπησε το καμπανάκι δυσαρέσκεια και δυσφορία κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρατηρείται και σε άλλα και στη Τσεχία ίσως στο Ηνωμένο Βασίλειο ήταν πολύ πιο έντονη αυτή η δυσαρέσκεια αλλά επαναλαμβάνω δυσφορία και δυσαρέσκεια υπάρχει και σε άλλα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό θα πρέπει να το έχουμε υπόψη όταν μιλούμε για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ας ε, κάνουμε μία παύση και ας αναθεωρήσουμε και αξιολογήσουμε τις ε, δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μερικές είναι περιτές. Θα πρέπει κάποιες αρμοδιότητες να επιστρέψουν στα κράτη-μέλη. Ο κύριος Ματζίτ Ματζίτ απουσιάζει. Περνάμε στην κυρία Ρόουετ για ένα λεπτό. Ε, με θλίβει βαθύτατα το γεγονό ότι οι διαπραγματευτέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση και τώρα και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποκλήθηκαν στι απειλέ του Μπόρι Τζόνσον και δέχτηκαν μια λευκό επιταγή με το ψευδό επιχείρημα ότι προσφέρει μια έφτακτη αποχώρηση. Εγώ καταψήφισα την ε, συμφωνία περί αποχώρηση γιατί δεν δίνει βάση για εμπιστοσύνη και αντιβαίνει στη δεδηλωμένη βούληση των ε, συνελεύσεών μας για τον βουλών μας και θέλει να πραγματοποιήσει πριν το 2021 το Brexit πάση θυσία και δεν προσφέρει ασφαλιστικές δικλείδες σε περίπτωση που δεν θα γίνει. Ε, είναι ε, αυτό το θλιβερό γεγονός η ανάκτηση του ελέγχου ε, και η αποχώρηση από τους 28 τότε θα δουν ότι το Ηνωμένο Βασίλειο έχασε το μεγαλείο του. Εμείς ε, χάσαμε τον αγώνα αλλά και σίγουρα ε, το κόμμα μου και σίγουρα ένας μικρός κύκλος ημών ελπίζουμε ότι θα επιστρέψουμε, ότι τα πράγματα θα γίνουν πάλι καλύτερα και όχι χειρότερα από τώρα. Ευχαριστώ. Ρόλαντ, για ένα λεπτό. Φοβερή οδή προ τον Brexit, λίγο στενάχωρη. Εγώ ψήφισα υπέρ της συμφωνίας γιατί πιστεύω στη δημοκρατία. Αυτό το Σύριαλ κράτησε σχεδόν τέσσερα χρόνια και τελικά ξεκαθαρίστηκε αυτό με τις εκλογές ξεκαθαρίστηκε και τελικά υλοποιήθηκε το Brexit και εμείς το κόμμα του Brexit εξελέγημε εκεί που δεν θέλαμε να βρισκόμαστε εδώ για να αλλάξουμε τον ρούν της ιστορίας το κόμμα του Brexit θα πρέπει αυτό να πιστωθεί αυτό που έγινε αυτή τη βδομάδα μόνο με τη δική μας ταραλία στάση ε, κόντρα στο καθεστώς, κόντρα στο δικοματισμό τελικά πετύχαμε αυτό που η σπουδαία χώρα μας ε, ψήφισε την αποχώρηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, για αυτό και είμαι πάρα πολύ περήφανος είναι ένα κατόρθωμα για όλους εμάς δεν ε, με νοιάζουν τα κροκοδίλια δάκρυα μην ε, στεναχωριέστε το μέλλον θα είναι ρόδινο για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δείξαμε ποιο είναι ο δρόμο Ο Θεό μαζί σας. Ο κύριος Πόσπισιλ. Ένα λεπτό, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Εγώ συμφώνησα και ψήφισα αυτή τη συμφωνία, αλλά σας ξεκαθαρίζω ότι προσωπικά είμαι 100% κόντρα στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου. Είναι κάτι που μου φέρνει μεγάλη στεναχώρια και βεβαίως δημοκρατικά θεωρώ ότι πρέπει να γίνει σεβαστή η θέληση του βρετανικού λαού, δεν μπορώ να κάνω τίποτε άλλο, αλλά θέλω να υποστηρίξω την συμφωνία που θα φέρει κάποιους κανόνες αυτή την αποχώρηση και θα προστατεύσουμε τους Βρετανούς που ζουν στην Αγγλία και δεν θα είναι άτακτη η αποχώρηση. Οπότε νομίζω ότι κάνουμε ό,τι μπορούμε και να είμαστε καλοί γείτονες με αγαστές εμπορικές επίσης σχέσεις κυρία Ντέιλι και εσείς λεπτό ευχαριστώ πρόεδρε όχι με τίποτα δεν με χαροποιεί το ότι είχαμε αυτούς τους ύμνους και τα δάκρυα και τις συμβουλές από αυτούς που θέλουν να μείνουν αυτό δείχνει το ότι δεν υπάρχει εδώ ενότητα τι έγινε με τις εκλογές και γιατί καταλήξαμε εδώ που είχαμε ένα τόσο σπουδαίο μέλος το οποίο αποχώρησε και ε, ε, να χτες τι κάνουμε ε, τίποτα, κουνούσαν το δάχτυλο σε όλους εκτός από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Την Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει τα προβλήματά της. Την Ευρωπαϊκή Ένωση που επιτρέπει να παρακάμπτονται όλοι οι δημοσιονομικοί κανόνες και να πληρώνουν την ύφη ο κόσμος και να σιωπά όταν βλέπουμε να φυλακίζονται στις πανικές φυλακές οι Καταλανοί σύντροφοι. Εγώ πίστεψα υπέρ της συμφωνίας. Όχι, δεν θέλω αδιαπέραστα σύνορα, αλλά αν γίνει κάτι τέτοιο, ε, τότε την ευθύνη θα την φέρει το κόμμα, τα κόμματα που θέλουν την παραμονή και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Φιτζέραλτ. Είδαμε λοιπόν σήμερα το πρωί και χθε πόσο βαθιά είναι τα αισθήματα που έχουν άλλε χώρε και άλλα μέλη για την αποχώρηση, την απώλεια του Ηνωμένου Βασιλείου. Αυτά ήταν ειλικρινή. Ειλικρινή γιατί βάζουν ένα τέλο σε μία ένταξη 47 ετών οικοδόμηση Ειρηνή, συνεργασία 47 έτη, 47 έτη όπου Ρίξαμε τα σύνορα και τα εμπόδια. Το θέμα λοιπόν ήταν ε, η δημοκρατία και η δημοκρατία στον Ηνωμένο Βασίλειο έπαιξε μεγάλο ρόλο θα ήθελα να ευχαριστήσω του συναδέλφου από τη Μεγάλη Βρετανία. Το θέμα όμω είναι πώ θα διαμορφωθεί το μέλλον. Κανεί δεν ξέρει ποιο θα είναι το μέλλον του Ηνωμένου Βασιλείου. Θα δούμε πώ θα πάει λοιπόν το Ηνωμένο Βασίλειο. Αλλά τώρα είναι η στιγμή να οικοδομήσουμε σε αυτό το νέο πλαίσιο νέε σχέσει και ελπίζω, ελπίζω αυτέ οι διαπραγματεύσει να γίνουν με ένα τέτοιο τρόπο που να μα επιτρέψουν να πετύχουμε μια συμφωνία και να μην αποκλίνουμε από τα πρότυπα τα οποία μα έβαλαν στο γκρουπ αυτό πρότυπα για το περιβάλλον, για την ασφάλεια των τροφίμων, αλλά ας βάλουμε πάνω απ' όλα τα συμφέροντα των πολιτών μας και των επιχειρήσεων μας που θέλουν τις πιο στενές σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση και το μέλλον. Ευχαριστώ η κυρία Βυσνιεύσκα για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι αγαπητοί συνάδελφοι, εγώ σέβομαι την κυρίαρχη απόφαση των Βρετανών και γι' αυτό ψήφισε υπέρ της συμφωνίας περί αποχώρησης. Και η αποχώρηση ε, της... Ε, αποχώρηση της, του Ηνωμένου Βασιλείου θα είναι ψυχρολουσία ε, στους θερμόμυαλους ε, φεντεραλιστές. Και ε, δεν θα πρέπει να έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση δυνατότητα να μπλοκάρει τα κράτη-μέλη. Θα πρέπει να συγκρατήσουμε την ανεξέλεκτη μετανάστευση. Θα πρέπει τα κράτη-μέλη να ανακτήσουν κάποιες αρμοδιότητες. Γιατί ε, θα πρέπει να καταπολεμήσουμε την κυριαρχία του ΔΕΚ και την υπερβολική ρύθμιση. Σίγουρα η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα είναι ίδια χωρί του Βρετανού, αλλά θα πρέπει να διδαχθούμε από το πάθημά μα. Και σίγουρα θα πρέπει να σκεφτούμε τι συμβαίνει και να στείλουμε να δείξουμε κόκκινη κάρτα σε αυτούς που λαχταρούν και έχουν βλέψεις προς το φεντεραλισμό στην ε, ομοσπονδιοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Ο κύριος Άριος Βόλσκι. Πρόεδρε, καταψήφισα τη συμφωνία του Brexit. Όχι γιατί ήμουν αντίθετο με την ε, συμφωνία, αλλά γιατί ήμουν αντίθετο με τον Brexit. Το Brexit είναι κάτι παραπάνω από έγκλημα. Είναι σφάλμα, για να αναφέρω τον Ταλή Ουρβάν. Αποτελεί μια αποτυχία, ένα σφάλμα και ένα ευρωπαϊκό δράμα ιστορικών διαστάσεων με μακροπρόθεσμες γεωπολιτικές συνέπειες τις οποίες ακόμα δεν κατανοούμε, δεν αντιλαμβανόμαστε και οι δύο πλευρές πρέπει να κατηγορηθούν και πολύ λυπάμαι ότι δεν φαίνεται οποιαδήποτε αντίληψη για το τι χάσαμε, γιατί χάσαμε την, τον Εμένο Βασίλειο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι πιο ασθενής, δεν θα είναι πλήρης χωρίς ε, το Ηνωμένο Βασίλειο από πολιτικής άποψης, από οικονομικής άποψης, γιατί είναι μεγάλη η οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου και θα είμαστε και πιο ασθενείς ε, και από στρατιωτικής άποψη και μια πιο ασθενή Ευρωπαϊκή Ένωση θα αντιμετωπίζει όλο και μεγαλύτερες απειλές από το εξωτερικό. Θα πρέπει λοιπόν να διερωτηθούμε γιατί συμβαίνουν όλα αυτά. Ευχαριστώ. Η κυρία Τζόουνς για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους Ουαλούς που μου έδωσαν την ευκαιρία να τους εκπροσωπήσω, να εκπροσωπήσω την άποψή τους και την ε, προτίμησή τους να παραμείνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ήταν σπουδαία αυτή η περίοδος, αλλά ήταν και άσχημη. Σπουδαία περίοδος γιατί εξασφαλίσαμε τα δικαιώματα και την αλληλεγγύη των εκπροσώπων μας και όσοι υπερψήφισαν ε, στο δημοψήφισμα για την παραμονή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ουαλία, όλα τα δικαιώματα για την ίση αμοιβή και τις ίσες συντάξεις. Ήταν χαρά μας η συνεργασία. Ο Τζόνσον λοιπόν στο μέλλον θα πρέπει να λουστεί τις συνέπειες του Brexit και η Ουαλία θα έχει τη θέση που της αναλογεί στο παγκόσμιο προσκήνιο γιατί έχουμε κοινέ αξίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση και με όλου τον κόσμο. Και τέλος να πω και να ευχαριστώ προς τους συναδέλφου και προς τους υπαλλήλους ε, και του γραφείου μου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τον γιο μου για τον οποίο τα ξεκίνησα όλα αυτά την επόμενη γενιά. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ. Ο κύριο Ζόνιτσα για ένα λεπτό έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Χθες εγώ ψήφισα αυτό που μου ζήτησαν ε, οι Βρετανοί πολίτες. Εμείς στην Πολωνία γνωρίζουμε τι εστί κυριαρχία και χαιρετίζουμε και σεβόμαστε την κυρίαρχη βούληση των πολιτών του Ηνωμένου Βασιλείου. Και θυμόμαστε ε, εμείς η Πολωνία ότι στην Αγγλία ε, υπογράφηκε μια σημαντική διακήρυξη των θεμελιωδών ελευθεριών πριν από 800 χρόνια αλλά και χθες είχαμε μια ημερομηνία ορόσημο, μια μετεχμιακή ημερομηνία που πιστεύουμε ότι θα ανοίξει το δρόμο για αγαστές σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένου Βασιλείου. Και θα ήθελα τα εθνικά κοινοβούλια να κρίνουν τη σχέση μεταξύ της Μεγάλης Βρετανίας ε, και των Εθνικών Κοινοβουλίων. Νομίζω ότι θα είναι καλύτερη κατάσταση αν αφήσουμε την κατάσταση στα χέρια των Εθνικών Βουλευτών. Ε, θα ήθελα να ευχηθώ καλή τύχη στην ε, Μεγάλη Βρετανία και να μην ξεχάσουν τους Πολωνούς πολίτες που συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη αυτής της χώρας. Σας ευχαριστώ. Δεν βλέπω τον κύριο Πόλτσακ στην αίθουσα, οπότε ο κύριο Τζαμπάσκι για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Εγώ ψήφισα υπέρ της Συμφωνίας Αποχώρησης, ε, σεβόμενος την κυρίαρχη βούληση του Βρετανικού λαού. Αυτή ήταν απόφαση των Βρετανών πολιτών. Απόφαση που την έλαβαν κυρίαρχα, όχι γιατί κάποιος τους πίεσε ή κάποιος επέμεινε, αλλά ύψωσαν τη φωνή τους κατά των Βρετανών γραφειοκρατών ε, που ήθελαν να εκχωρήσουν σημαντικές αρμοδιότητες. Και η σημερινή συζήτηση είναι χαρακτηριστική και η χθεσινή ψηφοφορία ε, συμβολική. Ε, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν επέτρεψε τη χρήση των εθνικών σημεών στην Ολομέλεια. Ε, για τέτοιους λόγους ψηφίζουν να αποχωρήσουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση κάποιοι Ευρωπαίοι πολίτες όταν ε, νιώθουν ε, ότι δεν είναι ευπρόσδεκτοι, όταν νιώθουν καταπίεση οι πολίτες, φυσικά θα θέλουν ε, να αποχωρήσουν. Δεν μπορούμε να στερούμε το δικαίωμα να χρησιμοποιούν του σημαία τους οι πολίτες. Αυτό θα πρέπει να μάθουν οι Βρετανοί γραφειοκράτες αν θέλουν στο μέλλον να έχουν μια Ευρωπαϊκή Ένωση. Για το σημείο αυτό, ο τελευταίος ομιλητής. Ευχαριστώ. Ε, θα πρέπει κάποιο να μπει για να βγει. Ε, γι' αυτό και εμείς ήρθαμε εδώ. εμείς και οι συναδελφοί φυσικά και είναι πονίδες στη συνθήκη, αλλά εγώ με δυσκολία την υπερψήφισα. Είπε ο δεν θα υπάρχει καμία παράταση μετά την 31 του στην υπόθεση της εξόδου γιατί πρόκειται να εγκαταλείψουμε αυτήν την αντι, ανταγωνιστική ε, ψευδέστηση. Οπότε ε, έτσι η χώρα μας μπόρεσε να έχει ατού διαπραγματευτά. Οπότε και εμείς μπορούμε να αποχωρήσουμε από την κακή συμφωνία, να προστατεύσουμε την ε, αλληλεία, την άμυνα, να έχουμε δική μας νομοθεσία, να δίνουν λόγο οι πολιτικά. Οπότε είδατε ότι όλα αυτό τελικά ήταν ένα αριστούργημα. Ήταν ένα λουλούδι το οποίο όλο ένα και καλύτερα μυρίζει. Ε, γι' αυτό και εγώ το ενέκρινα. Πάμε τώρα στο επόμενο σημείο. Έχουμε το χρονοδιάγραμμα του Κοινοβουλίου για το 21. Ο κύριος Πόσπης λέει το λόγο πρώτος. Κυρία Πρόεδρε, ψήφισα υπέρ αυτού του χρονοδιαγράμματος διότι ήθελα όμως να σας εξηγήσω γιατί το έκανα αυτό θεωρώ ότι κατά τη διαδικασία της έγκρισης αυτού του προγράμματος δεν λάβαμε υπόψη τη δουλειά που κάνουμε στις χώρες μας γιατί δεν δουλεύουμε μόνο εδώ, δουλεύουμε και στις χώρες μας πάντως ψήφισα υπέρ ε, αυτού του προγράμματος εργασιών αλλά νομίζω ότι δεν μας έχετε παραχωρήσει αρκετές εβδομάδες να περάσουμε σε εκλογικέ περιφέρειες και αυτό όχι και να κάνουμε διακοπές αλλά να έχουν περισσότερο χρόνο για δουλειά, πολιτική δουλειά στη χώρα μας και στην ε, Τσεχία ξέρετε ε, λέμε ότι δεν είναι κοντά μας η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν είναι κοντά στον κόσμο αν δεν μπορούμε να πάμε να δουλέψουμε ε, στην ε, εκλογή μας περιφέρεια, δεν μπορούμε να εξηγούμε στον κόσμο τι γίνεται και καθυστερεί η ολοκλήρωση. Ο επόμενος ομιλητής για το ίδιο θέμα. Όχι, ήταν μόνο ένας, μόνο ομιλητής, αλλά τώρα είναι πάλι ο κύριος Ποσπίσιλ. Και για το 22 ισχύουν τα ίδια θα πρέπει οι ευρωβουλευτές να έχουν χρόνο να δουλέψουν στην χώρα τους. Ε, αν έχουμε περισσότερες εβδομάδε εκεί, δεν δουλεύουμε λιγότερο. Ε, αντίθετα, είναι πάρα πολύ σημαντική η δουλειά που κάνουμε ε, στην πατρίδα μας. Ε, έτσι μπορούμε να ανασχέσουμε τον αντιευρωπαϊσμό και θα πρέπει εμείς που είμαστε φιλοευρωπαίοι να μπορούμε να εξηγήσουμε στον κόσμο, στους φοιτητέ και στα παιδιά τι γίνεται. Αλλά για να το κάνουμε χρειάζεται αρκετό χρόνος. Άρα να ληφθεί υπόψη ότι αυτό που ζητάμε δεν σημαίνει λιγότερη δουλειά. Σημαίνει περισσότερη πολιτική δουλειά στην πατρίδα μας. Για το επόμενο θέμα σε ό,τι αφορά για τους κοινούς φορτιστέ ε, για τις ε, κίνητε συσκευέ, ε, Η επόμενη μιλήτρια. Η κυρία Σόιδροβα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σε τελική ανάλυση υποστήριξα αυτό το ψήφισμα και συμφωνώ με την έκκληση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δράσει για να τραποποιηθεί η οδηγία για τις φορτιστές. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να προωθήσει την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών. Οι Ευρωπαίοι πολίτε παράγουν 16 κιλά ανά έτος ηλεκτρονικών απορριμμάτων, 10 κιλά πάνω από το παγκόσμιο μέσο όρο. Αν θέλουμε λοιπόν να εφαρμόσουμε την Πράσινη Συμφωνία, οι κοινοί φορτιστές θα αποτελέσουν ένα μικρό βήμα για την προστασία του περιβάλλοντος μας και για την εξοικονόμηση πόρων. Να κατανοήσουμε ότι το θέμα αυτό δεν είναι μόνο οι φορτιστές για τα κινητά, αλλά και για τα μπλέτες και άλλες γενικές συσκευές. Γι' αυτό και υποστήριξα την πρόταση αυτή. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε κ. Πάτων είναι επόμενος ομιλητής. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Υπερψήφισα υπέρ τη σύσταση για την τυποποίηση τέτοιων φορτιστών, γιατί πιο νοικοκυριό δεν έχει ολόκληρα ε, κυβότια τέτοιων ε, φορτιστών και καλώδιων. Έχω τέσσερα παιδιά με μετά από τόσα χρόνια και όλους τους φορτιστές για τις αβοντόβουτσες, για τις ταμπλέτες. Έχουμε τέσσερα μεγάλα κουτιά γεμάτα με καλώδια και φορτιστές. Υπάρχουν λοιπόν διάφορα προγράμματα για την ε, ανακύκλωση των ε, συσκευών αυτών, των φορτιστών αυτών. Αλλά λέμε δεν βαριέσαι, ίσω μα χρειαστούν κάποια στιγμή και τελικά δεν τα πετάμε. Και έτσι παράγουμε όλο μεγαλύτερη ποσότητα τέτοιων ε, φορτιστών. Αυτό είναι γελίο, είναι περιττό και έχει έρθει το πλήρωμα του χρόνου να αλλάξει ω μέτρο. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Βίσνια φυσικά για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, φυσικά υπερψήφισα την πρόταση για τους κοινού φορτιστές, για το φορητό ραδιοεξοπλισμό. Γιατί θεωρώ ότι η παρούσα κατάσταση είναι παράλογη τελείως. Ε, γεμίζουμε τα γραφεία μας, τα σπίτια μας με ένα σωρό σύρματα, καλώδια και φορτιστές που δεν έχουν καμία άλλη χρήση. Κάθε φορά που αγοράζουμε νέο τάμπλετ, νέο, νέα συσκευή, ε, αγοράζουμε και ή λαμβάνουμε και νέο φορτιστή. Συνεχώς συσσωρεύουμε νέους φορτιστές με το κάθε καινούριο τηλέφωνο. Αυτή είναι πραγματικά μια αλλοπρόσελη παράλογη κατάσταση. Και είναι δυνατόν ο ίδιος ε, παραγωγός για το πιο επικαιροποιημένο και πιο σύγχρονο κινητό να διαθέτει στην αγορά και νέο φορτιστή για την ίδια μάρκα. Νομίζω ότι σίγουρα η πρόταση για τον κοινό φορτιστή είναι αναφυσβήτητα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση και γι' αυτό υπερψήφισα. Ο κύριος Κέλεχερ, για ένα λεπτό. Για το ψήφισμα λοιπόν και εγώ το υπερψήφισα γιατί στην παρούσα φάση θα πρέπει να υποδεχτούμε ότι σε ό,τι αφορά την περιβαλλοντική ζημιά που προκαλείται από τον όγκο των φορτιστών και των καλωδίων είναι κάτι πραγματικά ε, και σίγουρα έχουμε τη δυνατότητα σε ό,τι αφορά την τεχνολογία καινοτομία για να εξασφαλίσουμε ότι μπορούμε να αναπτύξουμε ένα ενιαίο καλώδιο, ένα ενιαίο φορτιστή το οποίο και θα εξυπηρετεί όλες τις ανάγκες όπως αναφέρεται στο ψήφισμα. Δεν χωράει αμφιβολία ότι έχουμε γεμάτα σερτάρια και κουτιά σε όλα τα σπίτια στην Ευρωπαϊκή Ένωση με παλιέ τέτοιε συσκευέ και φροντιστέ. Όπω είπε ένα προηγούμενο ομιλητή, πάντα τα φυλάμε σε περίπτωση που τα χρειαστούμε στο μέλλον. Δεν γίνεται όμω ποτέ αυτό. Απλά κάφονται εκεί πέρα και σχηματίζουν χιλιόμετρα χρησιμοποιητών τέτοιων καλωδίων και φορτιστών. Καλό λοιπόν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δράσει, να συνομιλήσει με τη βιομηχανία και να εξασφαλίσει ότι ο στόχος του ψηφίσματος αυτός θα εκπληρωθεί για να έχουμε πραγματικά ενιαίες, ενιαίες συσκευές. Ευχαριστώ. Η κυρία Γκάντσα, δεν τη βλέπω στην αίθουσα όμω. Και περνάμε στον κύριο Λόπε Ιστούρη Βάιτ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Επιτέλους, επιτέλους ε, χρειάστηκε να απευθύνουμε έκκληση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να μας βοηθήσει είναι ε, ένα από τα μικρά λιθαράκια που μας βοηθούν να πλησιάσουμε καλύτερα και να δρέψουμε τους καρπούς της ψηφιακής επανάστασης. Το κάναμε με την προαγωγή. Να σταματήσουμε να μαζεύουμε χιλιόμετρα καλωδίων και σειρμάτων που τελικά είναι άχρηστα. Απλώς γεμίζουν τα σιρτάρια και τα ντουλάπια μας. Νομίζω ότι τέτοιου είδου ε, προτάσεις γίνονται πολύ ενθουσιοδός αποδεκτές από τους Ευρωπαίους πολίτες. Έχω και εγώ κουτιά ολόκληρα στο σπίτι σπίτι μου με άχρηστα καλώδια. Και εγώ είμαι υπέρ τη ελευθερία αγορά, αλλά πραγματικά μερικέ φορέ νιώθω ότι με χρησιμοποιούν οι παραγωγοί. Και παρακαλώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή α αναλάβει άμεσα δράση να εισακουστεί η βούληση των Ευρωπαίων Πολιτών και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δεν χρειαζόμαστε διαφορετικού φορτιστέ για τι συσκευέ μα. Ευχαριστώ. Η κυρία Πελτιέ, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Ε, και εγώ ψήφισα υπέρ του ψηφίσματο για να στείλουμε ηχηρό μήνυμα προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εδώ και δέκα χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απλώ συζητά. Θα πρέπει επιτέλου να δράσει. Δεν μπορεί να επαφίεται στην καλή βούληση των ε, παραγωγών τη της βιομηχανίας της ψηφιακής. Επίσης, ε, το λόμπι το, της ψηφιακής ε, παραγωγής άσκησε πιέσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Χρειαζόμαστε κοινωνικά ε, μέτρα και περιβαλλοντικά για να μειώσουμε τα ηλεκτρονικά μας απόβλητα. Αν δεν δράσουμε, αν δεν έχουμε κοινό φορτιστή, πώς θέλετε να δράσουμε για τον πλανήτη, να αντιμετωπίσουμε αυτή την περιβαλλοντική και κλιματική έκτακτη ανάγκη. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει πάρα αυτά δράση και να επιβάλλει υποχρεωτικά μέτρα για τα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ. Η κυρία Βρέτσιονοβά για ένα λεπτό. Μάλιστα. Καλησπέρα σας και πάλι κυρία Πρόεδρε και αγαπητοί συνάδελφοι. Εγώ δεν ψήφισα υπέρ του ψηφίσματος αυτού. Και φυσικά με ενοχλεί που ε, για κάθε νέα συσκευή έχουμε και νέο φορτιστή, αλλά αυτό θα μπορούσαμε να το αποκαλέσουμε και τεχνολογική εξέλιξη. Τα τελευταία χρόνια, τελευταία πενταετία, βλέπουμε τεράστιες διαφορές. Έχουμε πολλαπλάσιους ε, φορτιστές από ό,τι στο παρελθόν. Ένας κοινό φορτιστής όμως θα εμποδίσει και θα σταματήσει αυτές τις τεχνολογικές εξελίξεις, γιατί είναι ραγδαίες οι εξελίξεις αυτές. Και φορτιστές που θα υπάρχουν στην Ασία, στις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν θα είναι διαθέσιμοι για τους Ευρωπαίους πολίτες. Δεν θα υποδείξουμε εμείς την βιομηχανία την παράγει σίγουρα θα πρέπει να προστατεύσουμε την ανθρώπινη υγεία, αλλά δεν νομίζω ότι απειλείται από τους φορτιστές. Ευχαριστώ. Κυρία Γκλάβακ, ευχαριστώ πολύ. Εγώ τάχθηκα υπέρ του ψηφίσματος γιατί θεωρώ ότι είναι πολύ θετικό και μάλιστα το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα εδώ και 10 χρόνια ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει κοινό φορτιστή για το ραδιοεξοπλισμό. Σίγουρα η ελεύθερη αγορά είναι ακρογωνιαίος λίθος ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και σημαντικός παράγοντας οικονομικής ανάπτυξης. Στον κόσμο όμως έχουμε 50 εκατομμύρια ε, τόνους απόβλητα και εμείς έχουμε 12,3 εκατομμύρια τόνους απόβλητα το χρόνο. Οπότε ε, ένα μεγάλο τμήμα των παγκόσμιων αποβλήτων το παράγουμε εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και σίγουρα ένας τρόπος για να μειώσουμε αυτόν τον όγκο των αποβλήτων είναι να έχουμε κοινό φορτιστή του ραδιοεξοπλισμού. Γιατί δεν μπορούμε με την αγορά κάθε νέα συσκευή να αγοράζει ή να λαμβάνει και καινούριο φορτιστή Ευρωπαίος πολίτης. Και ο κοινό φορτιστής είναι και καλό περιβαλλοντικό μέτρο αλλά και καλό μέτρο για την οικονομία ε, που μπορεί να κάνει ο καταναλωτής. Δεν χρειάζεται να αγοράζει κάθε φορά νέο φορτιστή. Οπότε με τον κοινό φορτιστή δεν θα προστατεύσουμε μόνο και θα εξυπηρετήσουμε τον καταναλωτή, αλλά ταυτόχρονα θα συμβάλλουμε στην προστασία του περιβάλλοντος και στο μετριασμό των κλιματικών αλλαγών. Ευχαριστώ. Κύριος Γόλας, ευχαριστώ Πρόεδρε. 50 εκατομμύρια τόνοι είναι τα 6 κιλά ανάτομο και πρόκειται για μια γενιά αποβλήτων το 16 ήταν πάνω από 12 εκατομμύρια εκείνη η πάνω από 16 κιλά ανά άτομο τρεις φορές και έχουμε επίσης ηλεκτρονικά gadget αλλά έχουμε και τους φορτιστές που συμβάλλουν σε αυτά οι συμφωνίε με τη βιομηχανία δεν έλυσαν το πρόβλημα. Οι καταναλωτέ για νέε συσκευέ αγοράζουν νέους φορτιστές. Είναι τρελό αυτό ενώ έχουμε την κλιματική κρίση. Έχουμε ακτιβιστέ που κοντράρουν τον κοινό φορτιστή τρόμος κομισιόν κάτι θέλει να κάνει αλλά θα πρέπει να λάβει υπόψη τα συμφέροντα των καταναλωτών και του κόσμου Και τι γίνεται με το 13 δις που χρωστάει η Apple στην Ιρλανδία δεν τα παίρνει η κυβέρνηση ενώ τα χρειάζεται. Κέλλη, ένα λεπτό. Ψήφισα υπέρ αυτής της πρότασης. Το ζήτησε το ΕΛΚ τόσο καιρό που είμαι εδώ βουλευτής. Η, το λέει η κοινή λογική να έχουμε κοινό φορτιστή για όλες τις συσκευές τα κινητά, τα τάμπλετ κλπ. Θα έχουμε έτσι λιγότερα απόβλητα, λιγότερα αξεσουάρ. Μα ο κόσμος γι' αυτό μας εκλέγει. Είναι έτσι πιο εύκολη η ζωή του κόσμου. Άρα έτσι θα κάνουμε τη διαφορά για την καθημερινή ζωή του κόσμου. Θα έχουμε έτσι λιγότερα απόβλητα, λιγότερα σκουπίδια όπως είπε ο κύριος Γόλας. Θέλουμε με το ψήφισμα να υπάρχει μια τέτοια πρόταση που μέσα σε εξάμεινο να υπάρχει ο κοινός φορτιστής. Εκρεμεί αυτό πολύ καιρό. Χρειάστηκε πολύ κόπος αλλά να κάναμε πρόοδο σε αυτό το σημαντικό θέμα. Ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε ο τελευταίος για αυτό το θέμα τώρα. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Να σας το πω στα Ιταλικά. Δεν υπερψήφισα αυτό το κείμενο σχετικά με την ε, δυνατότητα να έχουμε κοινή, κοινό φορτιστή για τις συσκευές μας και για, και για τα κινητά μας βέβαια γιατί νομίζω ότι αυτό θα περιορίσει την ελευθερία επιλογής του καταναλωτή. Επίσης, θα ήθελα να σας πω ε, κάτι μεθοδολογικά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, εάν θέλει να αποκτήσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην γεωπολιτική σκακέρα θα πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι ο ρόλος της δεν είναι το να παρεμβαίνει στην ελεύθερη πρωτοβουλία των ε, πραγματικά παραγόντων των πλούτων και ενώ τις επιχειρήσεις. Αυτό πρέπει να κάνει είναι να έρει τους φραγμούς στην ελεύθερη κυκλοφορία των ε, εμπορευμάτων. Άρα, προσοχή να μην πέφτουμε θύματα των ακτιβιστών για το περιβάλλον και του λαϊκισμού τους. Θα πρέπει να υπάρχουν κάποιες πολιτικές επί τη βάση τεκμηρίωσης και επιστημονικών συμπερασμάτων. Ευχαριστώ. Πάμε τώρα στο επόμενο, στο μισθολογικό χάσμα ανδρών και γυναικών. Κυρία Σόιντροβα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που δίνετε το λόγο, Πρόεδρε. Κυρίε και κύριοι, το μισθολογικό χάσμα είναι 16% στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό αποτελεί μια βασική αδικία και παρά το γεγονός ότι έχουν γίνει κάποιες πρόοδοι σε κάποιες χώρες, αυτή η βελτίωση είναι πολύ αργή και είναι αλήθεια ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει λάβει διάφορα μέτρα για να βοηθήσει τα κράτη-μέλη να βελτιώσουν και να διορθώσουν την κατάσταση αυτή γιατί πρόκειται για θέμα επικουρικότητας και είναι στο χέρι των κρατών μελών η βελτίωση αυτή. Πιστεύω ότι η οδηγία για την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικού και οικογενειακού βίου είναι πολύ θετική γιατί θεωρώ ότι μπορεί να βοηθήσει τους γονείς και να ανελεχθούν επαγγελματικά και να εκπληρώσουν τα καθήκοντά τους στην οικογένειά τους. Εγώ απήχα όμως την ψηφοφορία αυτή γιατί διαφωνώ με το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να επιβάλλει υπερβολικές υποχρεώσεις για τα κρατημέλη και τις επιχειρήσεις προκειμένου να τροποποιηθεί η νομοθεσία, για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά την ευελιξία, σε ό,τι αφορά την εργασία τους. Σας ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε, στην κλίμακα των ευρωπαϊκών αξιών η ισότητα ανδρών και γυναικών πρέπει μόνο να ε, υπόκειται στον έλεγχο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αλλά δεν θα πρέπει να θεωρούμε ότι κυρίως οι γυναίκες θα πρέπει να φροντίζουν ε, τους ηλικιωμένους και τα παιδιά ή ότι αυτή δίνει δουλειά σημαντική ε, για αυτό υποστηρίζει την οικογένεια. αυτό θα είναι μια πολιτική επανάσταση και θα μπορούν να μπαίνουν στην οικονομία οι γυναίκες και θα έχουμε περισσότερη ανάπτυξη. Εγώ δεν ψήφισα υπέρ αυτού του κειμένου γιατί ε, βέβαια ήταν κάτι που το θέλουν όλοι αλλά νομίζω ότι έτσι η Κομισιόν ανακατεύεται με ε, θέματα οικονομικά των πολιτών και θέματα εθνικής αρμοδιότητας γιατί θα πρέπει νομίζω ε, να μην ρίχνουμε το βάρος στις ε, επιχειρήσεις και κυρίως στις μικρομεσαίες. Φυσικά θα πρέπει να μιλάμε μόνο για το χάσμα, αλλά θα πρέπει να μιλάμε για την ισότητα μεταχείριση για τις πολιτικές που βοηθάνε τις γυναίκες να εργάζονται. Thank you very much, Mr. Patton. Ευχαριστώ, κύριε Πάτεν, για ένα λεπτό υποστήριξα το ψήφισμα για πιο σωστή και δίκαιη αμοιβή. Προφανώς και οι γυναίκες θα πρέπει να αμοιβούνται σωστά στην αγορά εργασίας και το Ηνωμένο Βασίλειο, όπως και σε πολλά άλλα θέματα, είναι πολύ πιο μπροστά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί όμως το Ηνωμένο Βασίλειο θα πρέπει να αναγνωρίσει ότι το ίδιο θα πρέπει να ισχύει ως ισότητα για τις εθνικές μειονότητες και άλλες μειονότητες. Εγώ έχω μιλήσει για το θεσμικό ρατσισμό σε επανειλημμένα εδώ. Το γεγονός ότι έχουμε με 10% των Ευρωπαίων πολιτών από φιλετική και άλλες μειονότητες και ποτέ δεν έχουμε δει εδώ μαύρο επίτροπο ή σε άλλες θέσεις. Έχω να πω ότι κανένας κανένα ε, άτομο ε, μαύρο δεν έχει ε, εμφανιστεί σε οποιοδήποτε Προεδρείο Επιτροπής. Αυτό είναι λοιπόν πραγματικά παράδεκτο σε ό,τι αφορά και τι διακρίσει μεταξύ των φίλων και πέρα από όλα αυτά που διακηρύττουν ποτέ δεν πρόκειται να είναι ενωμένοι στην πολυμορφία εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αν δεν ρυθμίσουν τα εσωτερικά τους πρώτα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Βυζνιέσκα. Ευχαριστώ. Εγώ συμμετείχα στη σύνταξη του ψηφίσματος ε, του ECR για το μισθολογικό χάσμα. Και αυτό το πρόβλημα το διαπιστώνουμε το, και το συζητούμε όχι μόνο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά διαπιστώνουμε ότι υπάρχει μισθολογικό χάσμα 16% στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μάλιστα στην Πολωνία έχουμε από τα λιγότερα μισθολογικά χάσματα μεταξύ των κρατών μελών. Το ψήφισμα που συνέταξε εκ μέρους του ECR ζητά προσπάθειες ε, προκειμένου να έχουμε ισότητα των μισθών μεταξύ των φύλων σε εθνικό επίπεδο. Επίσης ε, ζήτησα περισσότερες, ε, περισσότερους βρεφονιπιακούς σταθμούς και υπηρεσίες φροντίδας προς τα παιδιά, γιατί συνήθως ε, οι γυναίκες ασχολούνται με τη φροντίδα των παιδιών και μένουν κάπως πίσω στην ε, επαγγελματική του σταδιοδρομία. Θα πρέπει λοιπόν να γίνεται καλύτερη συμφιλίωση του επαγγελματικού με το προσωπικό βίο. Ε, βέβαια, καταψηφίσατε το δικό μας ψήφισμα του ECR, αλλά υπερψηφίσατε ε, ψήφισμα που καταστρατηγεί την επικουρικότητα ε, και ουσιαστικά προκρίνει κάποιες διατάξεις που είναι επιβλαβείς για την επιχειρηματικότητα. Ευχαριστώ. Κύριος Μίλλερ για ένα λεπτό. Okay. Ευχαριστώ κι εγώ. Εγώ υπερψήφισα το ψήφισμα γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να εξισώσει τους μισθούς ε, και να καταπολεμήσει το μισθολογικό χάσμα των φύλων. Όπως αναφέρθηκε, ε, τα στοιχεία μας δείχνουν ότι οι γυναίκες στην Ευρωπαϊκή Ένωση αμείβονται 16% ε, λιγότερο από τους άντρες και μάλιστα ε, κατά μέσο όρο μπορούν και δύο μήνες να εργάζονται χωρίς αμοιβή. Ε, επίσης πολύ συχνά ε, λόγω της μερικής απασχόλησης ε, δεν έχουν συχνά προαγωγές ή ασχολούνται περισσότερο με τη φροντίδα των παιδιών και μένουν πίσω στα επαγγελματικά τους. Νομίζω ότι μια και ισότητα των φύλων είναι από τις θεμελιώδεις αρχές θα πρέπει να καταπολεμήσουμε το μισθολογικό χάσμα και να έχουμε δράσεις ώστε να αποφύγουμε τον επαγγελματικό διαχωρισμό τα ανδροκρατούμενα επαγγέλματα και να εγκρίνουμε μέτρα που θα μας επιτρέψουν να γεφυρώσουμε το μισθολογικό χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών. Σας ευχαριστώ κυρία Ward για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ. Την επόμενη εβδομάδα μετά από 47 χρόνια ε, της... Παραμονή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση που ήμασταν ε, προοδευτικέ ε, δυνάμεις δεν θα είμαστε πια για να υποστηρίξουμε αυτή τη γεφύρωση του μισθολογικού χάσματο. Θα ήθελα να επενέσω τι αδερφές από το Εργατικό Κόμμα που έδωσαν τόσα χρόνια μάχη για την ισότητα των φύλων. Θέλει πηγή έμπνευση για εμά και τι μελλοντικέ γενιέ, ώστε να μην είμαι η τελευταία εκπρόσωπο του Εργατικού κόμματο που θα λαμβάνει το λόγο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα ήθελα να απαντήσω φωτιρμή στην Τζέινι Μπούκαν, Μπάρμπαρα Κάσλ, Αν Κλόετ, Τζόι Κουίν, Κριστίν Κρόλε, Κάρολ Τάνκ. Πολίν Γκριν, Κριστίν Οντί, Μέλ Ριντ, Ανίτα Πόλακ, Άντζελα Μπίλιγχαμ, Μοτούλ, Βερόνικα Χάτσταφ, Γκλένι Σκίνοκ, Έλενετ Μόργαν, Σούζαν Μόντιγκτον, Άλιν Μακάρθη, Λίντα Μακάβαν, Λίντα Γκίλ, Κάθριν Στάλλερ, Μέρι Χόνεμπολ, Σμόλβουτ Άντερσον, Αναλυστότ, Τερέζα Γκρίφιν, Τζούντιθ Κέρτον Ντάρλινγκ, Κλέρ Μούντι, Άλεξ Μέερ και τέλος στη Τζάκι Τζόουνς. Ένα λεπτό, ο κύριος Κέλεχερ. Και εγώ θεωρώ και υπερψήφισα το κείμενο που φέρνει κάποια δικαιοσύνη γιατί ακόμα υπάρχουν στο χώρο εργασίας ανισότητες. Και θέλω η Ευρώπη να προάγει την ισότητα. Να αναγνωρίζεται επίσης και η διαφορετικότητα στο χώρο εργασίας και για ίση εργασία να υπάρχει ίση αμοιβή. Πρέπει να προσπαθήσουμε όχι μόνο να γεφυρωθεί αυτό το χάσμα θα πρέπει να το εξαλείψουμε. Ευχαριστούμε. Έχω κανένα λεπτό. Ανάθεμα. Δεν πρέπει να υπάρχει τέτοια ανισότητα. 16% είναι το χάσμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Χειρότερα στη χώρα μας. Και γιατί οι αρμόδιοι και σε μεγάλες εταιρείες και στο δημόσιο τομέα θεωρούν ότι θα πρέπει να υπάρχει ισότητα. Το ίδιο γίνεται και στις προσλήψεις και ιδίω σε ορισμένου τομεί. Ε, αυτά όλα εξηγούνται γιατί σε διευθυντικέ θέσει είναι κυρίω άντρε. Ανέκαθεν ω Ευρωβουλευτή είχα στο μυαλό μου το μέλλον της μικρής μου κόρη. Οπότε σε αυτή την τελευταία παρουσία εδώ ζητώ κάτι να γίνει για την ισότητα ανδρών και γυναικών. Ο κύριος Λόπεθ Ιστούριτ White έχει το λόγο. Κυρία Πρόεδρε, ψήφισα θετικά. Όχι για να υποκύψω στην φυλακιστική γραμμή της ε, αριστεράς ούτε για να είμαι υπέρ αυτού του απαρχαιωμένου φεμινισμού όπως είπε και ο κύριος Χουκ και εγώ έχω στο μυαλό τις δύο μικρές μου κόρες το μέλλον τους και άρα θα πρέπει να υπάρχει δικαιοσύνη να μην υπάρχει αυτό το χάσμα εις βάρος των γυναικών και έχουμε στη χώρα μας ξέρετε το ίδιο πρόβλημα και, και η κυβέρνηση αριστερή που δεν κάνει τίποτα είναι πάρα πολλές οι γυναίκες που υφίστανται τις συνέπειες αυτού του χάσματος άρα είναι λογικό να ψηφίσουμε υπέρ αυτού του κειμένου αυτής της προτάσεως και αυτό κάνει το Λαϊκό Κόμμα και στην Ισπανία και στην Ευρώπη Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε Αγαπητοί συνάδελφοι, αυτό το ψήφισμα είναι απαραίτητο γιατί υπενθυμίζει τις οικονομικές ανισότητες που είναι διαφορετικές μεταξύ ανδρών και γυναικών. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν έχουμε 40% χάσμα μισθολογικό σε ό,τι αφορά και τη συμμετοχή επίσης στην αγορά εργασίας. Αυτή η ανισότητα υφίσταται και στην σύνταξη. Οι συντάξει των γυναικών είναι 37% πιο χαμηλές από αυτές των ανδρών τη στιγμή που ψηφίζουμε το ψήφισμα αυτό στην Ευρώπη έχουμε ένα σύστημα, μεταρρυθμίζουμε το σύστημα συνταξιβότησης ε, μετά από έκκληση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη Γαλλία θέλει να προσαρμοστεί το σύστημα των συντάξεων μετά από έκκληση του, ε, του Πρόεδρου και αυτό, τα πρώτα θύματα θα είναι οι γυναίκες. Θέλω λοιπόν να στείλω ένα μήνυμα εδώ στην αίθουσα προς τον λαό της Γαλλίας και να σας πω ότι η αντιπροσωπεία μας θα αγωνιστεί και θα κάνει τα δύνατα δυνατά για να μπορέσει να αποφευχθεί αυτό το πολύ αρνητικό πρόγραμμα. Ευχαριστώ κυρία Σαϊμπή για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πρόεδρε ψηφίσαμε ένα κείμενο για το μισθολογικό χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών και εδώ πέρα διαπιστώνουμε λοιπόν ότι το χάσμα το μισθολογικό μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 37%, 37% και κάτι άλλο ενδιαφέρον είναι ότι έχουμε κράτη-μέλη που προσπαθούν να δώσουν ένα ελάχιστο επίπεδο στις γυναίκες για τι ε, συντάξει. και ο πρόεδρο Μακρόν κάνει ακριβώς το αντίθετο με τη μεταρρύθμιση του συνταξιδετικού συστήματος στην Γαλλία και οι μεγάλοι χαμένοι και οι μεγάλε συντημένες ήταν οι γυναίκες για το, οι διακοπές στην σταδιοδρομία των γυναικών λόγω εγκυμοσύνη η μερική απασχόληση, όλα αυτά έχουν ως συνέπεια ότι οι γυναίκες δεν μαζεύουν τελικά αυτά που χρειάζονται για να βγουν στη σύνταξη. Θα ήθελα λοιπόν να απευθύνω από εδώ μια έκκληση προς τον κύριο Μακρόν. Έχετε δύο επιλογές. Είτε θα συνεχίσετε να κάνετε τον καλό μαθητή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να καταστρέφετε το συνταξιωτικό μας σύστημα, είτε θα ακούσετε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και που είναι η δημοκρατικά αιρετοί εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας συστήνω το δεύτερο σε ό,τι αφορά τη μεταρρύθμιση του συνταξιδοτικού συστήματος. Ε, συνάδελφοι, δεν έχουμε χρόνο στην διάθεσή μας να τηρείτε τα χρονικά όρια. Ο κύριος Ράιλε, για ένα λεπτό, ευχαριστώ πολύ πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Τι συζητάμε σήμερα, συζητάμε την αρχή της ίσης αμοιβή για ίση εργασία. Και αυτό πέρα από το, τη διάσταση του φίλου. Αυτό είναι κάτι το αυτονόητο για μένα, αλλά δεν ήταν πάντα έτσι. Και πολλά έχουμε πετύχει τον τελευταίο καιρό. Ο 20 ο αιωνα ήταν ο αιώνα τη χειραφέτηση. Διαπιστώνουμε λοιπόν σήμερα ότι, οι γυναίκες στην Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθούν να βγάζουν 16% πιο λίγα από ότι οι άντρες. Είναι σκανδαλώδε. Αλλά διερωτώμαστε γιατί. Καταρχάς και να είμαστε ειλικρινεί, επειδή οι γυναίκε, κάνουν παιδιά. Και έτσι αφιερώνουν πιο πολύ στην χρόνο στην τροφή των παιδιών και τους χρειάζεται πιο πολύ χρόνος μέχρι ότου αποκτήσουν δεξιότητες. Αυτό είναι το πρόβλημα λοιπόν. Χρειαζόμαστε μια σωστή πολιτική για την οικογένεια γιατί οι γυναίκες οι οποίες κάνουν παιδιά θα πρέπει να είναι στο επίκεντρο. Και αυτό που είναι ενδεικτικό είναι ότι αυτή η διαφορά μης θεολογική είναι πολύ πιο χαμηλή σε χώρες όπως η Πολωνία που έχουν δυτική κυβέρνηση από σε ευλελεύθερες χώρες. Ευχαριστώ πολύ, λέει η Πρόεδρος κανονικά θα έπρεπε να τελειώσουμε στην παρούσα φάση, αλλά θα επιτρέψει να συνεχίσουμε. Η κυρία Ντάλη, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι είναι ντροπή και όνειδος που στην Ευρωπαϊκή Ένωση εν 2020 οι γυναίκες κερδίζουν κατά 16% λιγότερο την ώρα από τους άντρες πριν να δούμε καν τις άνιση, τα άνισα ποσοστά μεταξύ ανδρών και γυναικών. Φυσικά οι γυναίκες υφίστανται το κόστος της μητρότητας, της μη αναγνώρισης ε, και αμοιβή της ε, εργασίας της οικιακής ή της φροντίδας ε, εξαρτημένων ατόμων στο σπίτι. Οπότε υπάρχουν πολλά καλά στο ψήφισμα, αλλά κράτησα στάση αποχής γιατί ε, ασχολούμαστε με τα συμπτώματα και όχι με τις αιτίε, την αρρύθμιστη επισφαλή απασχόληση που πλήττει δυσανάλογα τις γυναίκες και επίσης έχουμε το χάσμα μεταξύ των φύλων. Δυστυχώς δεν είναι πλήρες το ε, ψήφισμα θα πρέπει να σταματήσουν οι γυναίκες επιτέλους μερικές φορές θα δουλεύουν σαν σκλάβες. Θα πρέπει να διορθώσουμε το σύστημα ριζικά. Ο κύριος Γουάλλας. Ε, οι στατιστικές για το μισθολογικό χάσμα επισημάνθηκαν από τους συναδέλφους και είναι αναφυσβήτητα ντροπή δεν μας περιποιεί καθόλου τιμή η κατάσταση αυτή. Επίσης αυτό είναι το αποτέλεσμα μακροχρόνιων νεοφιλελεύθερων πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επιδεινώνουν την ε, άνηση μεταχείρισης βάρων των γυναικών και αυξάνουν το μισθολογικό χάσμα ζητούσαμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μην προωθήσει στάσεις πολιτική που αυξάνουν τις επισφαλείς τη εργασίας, την απορρίθμιση του ωραρίου και τη απασχόλησης, τη μείωση των μισθών, την ιδιωτικοποίηση δημοσίων υπηρεσιών και των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης. Όλα αυτά υπονομεύουν το έργο των συνδικάτων και παρόλα αυτά είναι πραγματικότητα. Δείτε η πατρίδα μου, η Ιρλανδία, πόσο αργά αναγνώρισε τα αναπαραγωγικά δικαιώματα των γυναικών. Χρειάστηκαν τόσα χρόνια για να το κάνει. Οι αιτίε όμω του μισθολογικού χάσματο μεταξύ ανδρών και γυναικών απορρέει και από την απορρίθμιση της εργασίας και την υποβάθμιση της ε, εργασίας, την απαξίωση της. Θα πρέπει επιτέλους να αλλάξουν τα πράγματα. Ευχαριστώ. Δεν βλέπω την κυρία Βρετσιονοβά στην αίθουσα, οπότε το λόγο έχει η κυρία Φιτζέρολτ η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν ανέκαθεν υπερασπιστής, υπέρμαχος της ισότητας. Φαίνεται και στο ψήφισμα και ευχαριστώ τους συναδέλφους που το υπερψήφισαν. Είναι πολύ σημαντικό ψήφισμα και είχαμε αγαστή συνεργασία υπερκομματική και το ΕΛΚ ήταν αναφαδόν υπέρ του ψηφίσματος ήταν μια σύστασή μας από το 2014 και δεν αναλύθησαν αρκετές δράσεις για να μειωθεί το μισθολογικό χάσμα των φύλων. Ούτε το συνταξιοδοτικό χάσμα μειώθηκε. Είναι της τάξης του 36% και το μισθολογικό χάσμα είναι στο 16%. Θα ήθελα να πω λοιπόν στις επιχειρήσεις, στις εταιρείες, εθνικές και πολυεθνικές, στις κυβερνήσεις και στα ΜΜΕ να ξυπνήσουν γιατί αναμένεται μια οδηγία που θα καταστήσει υποχρεωτική τη διαφάνεια στους μισθούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα ενισχύσει τα δικαιώματα των εργαζομένων, τη διαφάνεια στους μισθούς και τη συγκρισιμότητα μεταξύ των διαφόρων θέσεων απασχόλησης. Είναι απολύτως απαραίτητο και το ψήφισμα για το μισθολογικό χάσμα και την καταπολέμησή του στέλνει το χειρό μήνυμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ότι είμαστε σοβαροί και θα το διεκδικήσουμε. Θα πρέπει βέβαια μετά τη σύσταση του 2014 φαίνεται ότι κάποιες χώρες ε, ε, ψήφισαν αύξηση των μισθών των γυναικών. Κάτι που είναι θετικό. Κολλά, Εμείς οι πειρατές ψηφίσαμε υπέρ αυτού του ψηφίσματος διότι πρόκειται για ένα σοβαρό θέμα που πρέπει να επιληθεί όμως ψηφίσαμε κατά της παραγράφου 13 που αφορά κάποιες ποσοστώσεις για τα δύο φύλλα. Δεν είναι ο σωστός τρόπος ε, έτσι να γεφυρωθεί το χάσμα. Θεωρούμε ότι οι δεξιότητες, η γνώση, ε, αυτά είναι ε, θησαυρή θέματα που δεν ανοίγουν σε συγκεκριμένο φύλλο. Άρα χρειάζεται κάποια μακρόπνοη λύση που δεν είναι οι ποσοστώσεις να εδληφθούν μέτρα για διαφάνεια και προσβασιμότητα σε υπηρεσίες πλαισίωσης των ανηλίκων, σε λογικές τιμές και έτσι να μπορούν καλύτερα να συμμετάσχουν στην αγορά εργασίας οι γυναίκες αυτά που λέει η παράγραφος 13 ε, θα συνεχίσουμε να βρίσκουν αντίθετους αυτές οι ποσοστές. Ο κύριος Πόλτσακ δεν είναι εδώ λέει πρόεδρος. Άρα ο επόμενος είναι ο κύριος, η κυρία Τζόνς. Εσάς ευχαριστώ. Με ενθουσιάζει ότι τη τελευταία μου ψηφοφορία εδώ μου έδωσε την ευκαιρία να ψηφίσω ναι για τα δικαιώματα των γυναικών για να μπορέσει να γεφυρωθεί αυτό το χάσμα το μισθολογικό ακόμα έχουν πολλή δουλειά μπροστά μας αλλά το εργατικό κόμμα έχει παρελθόν υπέρ της ε, αλληλεγγύης αξιοπρέπειας και υπέρ των δικαιωμάτων των εργασιακών και στην Ευρώπη και στη Βρετανία και στην Ουαλία θα συνεχίσουμε στην ίδια διαδρομή και να ελπίσουμε ότι δεν θα χάσουν τα δικαιώματά μας με την κυβέρνηση Τζόνσον οι ανήλικοι και οι γυναίκες είναι οι πιο ευάλωτοι σε σχέση με τα μισθολογικά σε σχέση με την βία θα πρέπει μόνο σε αυτά όλα να τα αντιμετωπίσουμε. Τέλος, ευχαριστούμε όλους όσους στάθηκαν στο πλάι μας και θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε υπέρ της Ουαλίας ισότητας, αλληλεγγύης και αξιοπρέπειας. Ο κύριος Χάουαρθ. Ένα λεπτό. Κυρία Πρόεδρε, είναι ιδανικό ότι εμεί ε, για τελευταία φορά ψηφίζουμε εδώ για εμεί οι εργατικοί για τη γεφύρωση του χάσματο για ένα θέμα που εμεί θεωρούμε ότι είναι αυτονόητο η ισότητα σημαίνει ισότητα ε, και στα μισθολογικά δεν συμφωνούν όλοι να γιατί φτάσαμε στο να ψηφίσουμε για τελευταία φορά για μια προοδευτική κοινωνία κάποια θέματα τα θεωρεί αυτονόητα ε, τότε αρχίζουν τα προβλήματα Οπότε πρέπει να δώσουμε και άλλες μάχες. Επομένως, ε, όταν έχουμε τέτοιες ανισότητες και μετά χάνονται θέσεις εργασίας, αυτό. Αλλά ενώ να συνεχίσω στα γαλλικά το πρόβλημα ε, υπάρχει και εδώ στο Κοινοβούλιο. Θέλω να ευχαριστήσω το προσωπικό ασφαλείας, το προσωπικό των εστιατορίων, όλους τους ε, οδηγούς. Σας ευχαριστώ για το όσα κάνατε. Καλή τύχη, καλό κουράγιο και στο επανειδή. Ο κύριος, κυρία Φόξ είναι η τελευταία ομιλήτρια. Δεν το ψήφισα αυτό το κείμενο, γιατί δεν πιστεύω ότι πρέπει να γεφρώσουμε το χάσμα αλλά υπάρχουν και άλλα θέματα και άλλα κενά που δεν τα συζητούμε. Έχουμε τους ευρωκράτες που χρησιμοπληρώνονται αλλά για το προσωπικό κανείς δεν λέει τίποτα για τους κλητήρες, τους οδηγούς τους καθαρίστριες τους ε, μεταφραστές ε, όλοι αυτοί που τόσο μας έχουν βοηθήσει ε, και είναι αντικειμενικοί δεν έχουν προτιμήσει κομματικές βοήθησαν και εμάς το κόμμα του Brexit όλοι αυτοί τις εργατικές τάξεις παντού στην Ευρώπη που γίνονται με τη λιτότητα ακόμα πιο φτωχοί οι οικονομικές αποφάσεις των Βρυξελών τους θεωρούν παράπλευρη απώλεια θύματα των μεγάλων εταιριών και ε, έχουμε την δεξιά, τα κίτρινα γυλαίκα ε, αυτά είχα να σας πω σε αυτή μου την τελευταία αγόρευση να μην δαιμονοποιείτε τους πολίτες αλληλεγγύη με την εργατική τάξη όταν αντιδρά και ελπίζω ότι η αντίδραση της εργατικής τάξης θα φέρει την νίκη. Σας ευχαριστώ. Πέρας τη συζήτηση λέει η Πρόεδρος. Έχουμε τα πρακτικά τα οποία πρόκειται να υποβληθούν στην επόμενη Ολομέλεια προς έγκριση. Εάν δεν έχετε κάποια ένσταση θα προωθήσω αρμοδίως αυτά τα κείμενα τα οποία ψηφίσαμε. Οπότε διακόπτεται τώρα η σύνοδος πέρα συνεδριάσεως. Ευχαριστώ τους ε, διερμηνείς. Have